So, colleagues, let's get Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο και σοβαρό είναι και ε, είναι πραγματικά η κατάλληλη στιγμή για να το συζητήσουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μία ε, μελέτη την οποία ε, ε, ξεπώνησε για μας το τμήμα C ε, των πολιτικών μελετών. Τώρα πλέον είναι έτοιμη αυτή η έκθεση και μπορείτε να την πάρετε αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο ανάγνωσμα και σας το συστήνω. Λοιπόν, Τώρα φτάσαμε στην εξέταση του σημείου 21 και συγκεκριμένα την αναφορά 0967 του 2012, 1418, 0446, καθώς επίσης και την 0289 και 0906 πάνω στο ίδιο θέμα. Θα δώσω το λόγο στη Ζακλίν Κοτεχίλ, η οποία εκπροσωπεί τον Δήμαρχο του Πάσχα, καθώς επίσης και την ε, Κριστίν Κόρτινσεν Μπεκιάρντ Γένσεν. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσω, η γραμματεία ανέφερε ότι έχω 5 λεπτά για κάθε αναφορά. Είναι εντάξει. Όχι για κάθε αναφορά. Για καθέναν από τους ομιλητές, κάθε ομιλήτρια. Όχι, όχι, λέει η ομιλήτρια. Ναι, υπάρχουν πολλές ε, αναφορές, οπότε έχετε, ναι, πέντε λεπτά έχετε. 10 uh, Ωραία, 10 λεπτά σας δίνουμε λοιπόν. Πάρτε 10 λεπτά. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που με καλέσατε να προσώσω την αναφορά μου που κάνει έκκληση για δικαιώματα ψήφου για ε, Βρετανούς ε, ε, υπηκόους που ζουν σε κράτη-μέλη. Είχε ε, παρουσιάσει και μια αναφορά μια από την Ισπανία, μια Βρετανή. Οι Βρετανοί πολίτες ήδη ζουν στην αβεβαιότητα και σε μειωμένα έσοδα. Η οικογένειά μου δεν είχε δίκαιο να ψηφίσει στο δημοψήφισμα που επηρέασε τι ζωέ μας. Έχουμε και ε, την υποστήριξη διαφόρων εκστρατιών ε, από πολίτες Βρετανούς που υποφέρουν από το Brexit. Έξι χρόνια μετά την αποδοχή της αναφοράς μου. Δεδομένη στις θέσεις της Επιτροπής, ε, η αφαίρεση των δικαιωμάτων ψήφου είναι εθνική αρμοδιότητα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επιθυμήσουμε στην Επιτροπή και στα μέλη εδώ σήμερα ότι η ίδια Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα αυτό της αφαίρεσης των πολιτικών δικαιωμάτων το 2010. Υποστηρίζει τις ε, αξιώσεις αυτής της αναφοράς και επανέλαβε τις συστάσεις στην περσινή έκθεση. Η Επιτροπή αυτή επίσης υποστήριξε την ε, αναφορά αυτή το 2014 και τον Ιούνιο του 2016, εβδομάδες μετά από το δημοψήφισμα, όπου η γενική διάθεση ήταν πάρα πολύ θλιβερή. Έχουν γίνει δράσεις ε, μπροστά στην Βρετανική κυβέρνηση. Νομίζαμε ότι λύθηκε το 2015, όπου μας προσχέθηκαν ότι οι Βρετανοί ε, θα είχαν δικαιώματα ψήφου για όλη του τη ζωή. Αλλά τελικά αυτό δεν πέρασε ω νομοθεσία σε καμιά από τι εκλογέ, εκλογές, ε, οι οποίε ήταν σημαντικέ ε, για την όλη διαδικασία του Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να μην μα υπολογίσει στο δημοψήφισμα και δεν συμμετείχαμε εμεί στην πιο σημαντική απόφαση τη ζωή μα μετά από πολλέ ψευδεί υποσχέσει. Καταλαβαίνετε πόσο είμαι δύσπιστη όσον αφορά την προτινόμενη νομοθεσία. Το χειρότερο είναι ότι δεν αναφέρεται στη... Ότι αναφέρεται ότι εμεί αποκλειόμαστε από οποιαδήποτε ψηφοφόρια αν υπάρξει και δεύτερο δημοψήφισμα. Είναι βέβαια η κατάσταση και χαοτική στη Μεγάλη Βρετανία. Ε, λέει ο κ. Μπαρνιώτα, επομένει 25% να διασαφινιστεί από το συμφωνία. Περνάει ο χρόνος, έχουμε το πρόβλημα των σύνορων της Ιρλανδίας. Ε, για πιθανή απάτη έχει συζητηθεί από τους ε, υπαρμαχούς της ε, αποχώρησης. Εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να καταρρεύσει η συμφωνία χωρίς καμία εγγύηση για τα δικαιώματα των πολιτών. Η σημερινή κοινοβουλευτική ψηφοφορία μας δίνει την επιλογή συμφωνίας ή καμία συμφωνίας και προσπαθεί αντιπολίτευση να υπερασπίσει ενδεχομένως και ένα νέο δημοψήφισμα. Αυτό αποκτά όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη όσο μαθαίνουμε ποιες θα είναι ε, οι συνέπειες του Brexit. Το κοινοβούλιο αυτό θα ψηφίσουν ε, τη συμφωνία απόσυρσης. Θεωρούμε ότι δίκιο θα ήταν και οι Βρετανοί να πούν την απόψή τους. Αν υπάρξουν προώρες εκλογές ή νέο δημοψήφισμα, αυτό που θα ήταν καταστρεπτικό θα ήταν να μην έχουμε εμείς το δικαίωμα ψήφου. Το θέμα δεν είναι απλά ε, του, Μεγάλου, ε, του, Μεγάλου, του Ηνωμένου Βασιλείου επηρεάζει τους ε, Δανούς πολίτες, τους Κύπρους πολίτες, πολι, όσοι πολίτες χάνουν το δικαίωμα ψήφου που ζουν σε άλλες χώρες ως Ευρωπαίοι πολίτες και δεν μπορούν να ψηφίσουν ούτε στη χώρα κατοικία τους όπως τα παιδιά μου, εκεί όπου εργάζονται και πληρώνουν φόρους δεν μπορούν να ψηφίσουν. Η δημοκρατική συμμετοχή είχε αναγνωριστεί από την ε, Κομισιόν ε, ως δικαίωμα της ελευθερίας κυκλοφορίας ε, των προσώπων. Δυστυχώ δεν έχουμε διασφαλή ψήφο, δικαίωμα ψήφου για όλου του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο θα ήταν διαφορετικό αν αυτά τα 4,5 εκατομμύρια Βρετανών είχαν δικαίωμα ψήφου. Ε, Εσεί λέτε ότι δεν έχετε πραγματική εξουσία, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχετε. Έχω δει ποιο είναι το αποτέλεσμα των δράσεων του Κοινοβουλίου ε, για θέματα περιβαλλοντικά στι περιοχέ μα. Με τον Brexit έχετε σίγουρα εξουσία ε, ψηφίζοντα την τελική συμφωνία. Συμφωνία που δεν αναφέρει τα πολιτικά δικαιώματα των Βρετανών πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών μετά από ότι ο Brexit στη μεταβατική περίοδο. Το να έχουμε το δικαίωμα να, ψηφίσουμε στη χώρα κατοικία μα οι ισπανικές αρχές δεν μας έχουν πει τι θα γίνει στη συνέχεια. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν γνωρίζει. Το δικαίωμα ψήφου και πολιτικής εκπροσώψης είναι θεμελιώδη στοιχεία της δημοκρατικής κοινωνίας. Πράγμα για το οποίο πολλοί κόσμος πολεμά και πεθαίνει. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερασπίσει το δικαίωμα των πολιτών του να ψηφίζουν οι Βρετανοί πολίτε δεν καλύπτονται από καμία συνταγματική διάταξη που να ορίζει τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει του ούτε να του διασφαλίζει το δικαίωμα ψήφου. Η συνθήκη τη Λισαβόνα μα παρέχει σαφά δικαιώματα ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια και το δικαίωμα να ψηφίσουμε σε τοπικέ και περιφερειακέ εκλογέ, το οποίο χάνουμε, ενισχύοντα περαιτέρω ε, τη δική μα δημοκρατική συμμετοχή. Μπορεί να καταλήξουμε να μην μπορούμε να ψηφίσουμε πουθενά. Σήμερα εξακολουθούμε να είμαστε πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δικαιώματά μα. Για αναφορά το άρθρο 50 μπορεί να διακοπεί, να ανακοπεί, επιτρέποντα την κατάσταση να αναστραφεί. Αν υπάρξει ψηφοφορία για την τελική συμφωνία απόσυρση, είναι δημοκρατικό δικαίωμα όλων των Βρετανών πολιτών να πούν την άποψή του. Για άλλη μια φορά, κάνω έκκληση προ τα μέλη τη Επιτροπή σα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσετε επιγόντω για να αποκτήσουμε εμεί το δικαίωμα ψήφου είναι σίγουρα εθνικό, εθνική αρμοδιότητα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πράγματα υπερασπιζόμενη τι δημοκρατικέ αρχέ τη συνθήκη όπου αναφέρεται ότι κάθε πολίτη υποχρεούται να συμμετέχει, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή τη Ένωση. Και εμεί θα απευθυνθούμε στο Βρετανική κυβέρνηση να του ζητήσουμε να άρει αυτή την απερχαιωμένη διάταξη ώστε να μπορούμε εμεί να ψηφίζουμε στι ευρωεκλογέ και στα δημοψηφίσματα θα πρέπει να γίνει μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια ώστε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση των πολιτών που έχουν χάσει το δικαίωμα ψήφου, ώστε να υλοποιήσει τη συστάση της Επιτροπή, ενδεχομένως και διαδικασία κατά ή κάποια ε, διαδικασία στο δικαστήριο. Τέλος, για τα πολιτικά δικαιώματα των ε, Βρετανών και των Ευρωπαίων πολιτών εάν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ και να επισημάνω ότι όλο αυτό έχει παρατραβήξει. Η παρέμβαση σα τώρα είναι κρίσιμη σημασία. Η ενωμένη σα φωνή θα έχει αποτέλεσμα και η δημοκρατική αδικία που αντιμετωπίζουμε όλοι εμεί που έχουμε χάσει το δικαίωμα ψήφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε επιτέλου να επιληθεί. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που επιμένετε. Είναι η τρίτη φορά που έρχεστε εδώ και κάθε φορά την άφηξή σας την εκτιμάμε δεόντως. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην επόμενη ομιλήτρια. You need to, you need to open your microphone. That's it. Good. Thank you very much. I'm not a politician. Δεν είμαι πολιτικός, είμαι Βρετανή πολίτης και Ευρωπαία πολίτης. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούν ότι η προστασία των πολιτών είναι κάτι το σημαντικό για μια συμφωνία που θα ακολουθήσει το Brexit. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για να δούμε σε ποιο βαθμό παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια και οι Ευρωπαίοι πολίτες παραβιάζονται τα δικαιώματά τους όσων κατοικούν τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ δεν έχω άμεση πρόσβαση στα, στους Βρετανούς βουλευτές, δεν είμαι εκλογέας και γι' αυτό θα ήθελα να με ακούσετε. Έχω τα ίδια δικαιώματα με τους Βρετανούς πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο να ψηφίζω σε θέματα σχετικά με την Ένωση. Όμως οι Βρετανοί πολίτες σαν και εμένα που έχουν ζήσει σε άλλη χώρα για πάνω από 15 χρόνια εξαιρέθηκαν από τη συμμετοχή στις πιο σημαντικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο ή μάλλον δημοψήφισμα το δημοψήφισμα αυτό για την ιδιότητα μέλους της ε, Βρετανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάτι το σημαντικότατο για την καθημερινότητά μας όπως ε, και για τη ζωή των Βρετανών που ζουν στις άλλες χώρες της Ένωσης. Εγώ θα χάσω το διαβατήριό μου. <clears throat> Η αποχώρηση από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει συνταγματικές συνέπειες και θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και ε, την ζωή των πολιτών εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Αν αποδεχθώ ότι έχασα το δικαίωμα ψήφου γιατί χρησιμοποίησα το δικαίωμά μου να ζήσω σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κάτι το οποίο δεν έχω κάνει, τότε οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για πάνω από 15 χρόνια θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν αντί για μένα μιας και είναι μόνιμοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, πληρώνουν φόρους εκεί και ζουν τις ζωές τους εκεί. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο αρνούμενο <clears throat> και ε, στους Βρετανούς πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα το δικαίωμα και στους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα ψήφου δημιούργησαν και οδήγησαν σε ένα δημοψήφισμα τελικά το οποίο αγνόησε τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν τα δικαιώματα που τους απέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο πολύ συχνά λέγει ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει το Brexit σεβόμενο ε, το καθήκον του να ε, σεβαστεί την επιθυμία του λαού. Αλλά πώς ε, ένα τέτοιο αποτελέσματα μπορεί να θεωρηθεί σαν βούληση του λαού όταν τόσα μέλη του λαού αυτού αγνοήθηκαν. Έχω μια ερώτηση για μας, για σας και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε πολίτες. Είμαστε 4,5 εκατομμύρια. And thank you for... Σας ευχαριστούμε πολύ που ταξιδέψατε τόσο μακριά έτσι ώστε ε, να υποβάλλετε το ερώτημα αυτό, αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς αυτό το ερώτημα. Ε, η ίδια η παρουσία σας εδώ είναι η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε εμείς. Την ε, ερώτηση όμως πρέπει να την υποβάλλετε τουλάχιστον στην Βρετανική κυβέρνηση, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά σας. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναφέρει ότι η κατάσταση της ηθαγένειας των, της Ευρωπαϊκής είναι επιπρόσθετη ε, της ε, ε, που έχουν από το κράτος μέλος το οποίο, ε, από το οποίο προέρχονται. Και βάσει του άρθρου 21 της Συνθήκης Λειτουργίας τους επιτρέπεται η ε, ελεύθερη κυκλοφορία, όπως επίσης και δυνάμει το άρθρο 45 της, ε, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, ε, τους δίνεται το δικαίωμα να ψηφίζουν σε ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές στην ευρωπαϊκή χώρα στην οποία διαμένουν με ίδιες συνθήκες με τους πολίτες της χώρας αυτής. Ωστόσο, ε, τα δικαιώματα αυτά δεν επεκτείνονται έτσι ώστε να συμπεριλάβουν και τις εθνικές εκλογές. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν και είναι δικιά τους αποκλειστική αρμοδιότητα ε, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές. Ορισμένες χώρες-μέλη έχουν ήδη θεσπίσει νόμους ε, που εξισούν τα περισσότερα ε, δικαιώματα ψήφου και στις εθνικές εκλογές που ε, ζουν ε, ε, είτε για πολίτες της δικής τους χώρας που ζουν αλλού, είτε για πολίτες άλλων χωρών που ζουν στις δικές τους χώρες. Πάντως, δεν υπάρχει γενική πολιτική όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή δικαιώματα ψήφου στι εθνικέ εκλογέ ε, για τους πολίτε που ζουν αλλού. Και επομένω, υπάρχουν ε, κάποιοι πολίτε ε, οι οποίοι βρίσκονται εν τέλει χωρίς δικαίωμα ψήφου στην νέα χώρα μέλο στην οποία ζουν. Η Κομισιόν ήδη το 2010 ε, στην έκθεση για την ε, ηθαγένεια ε, θεώρησε ότι αυτό το θέμα της απώλειας του δικαιώματος ψήφου είναι ένα πρόβλημα. Εξού και ξεκίνησε με έναν προβληματισμό και μια συζήτηση έτσι ώστε να βρεθούν οι πολιτικές εναλλακτικέ οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Κάλεσε επίσης η Κομισιόν τα μέλη, τα κράτη-μέλη να βρουν μια λογική λύση όσον αφορά το πρόβλημα αυτό. Σε βάση αυτού του πολιτικού διαλόγου, η Κομισιόν τρία χρόνια μετά, το 2013, στη νέα έκθεση για την ε, ε, ηθαγένεια, έδωσε κάποιες ε, εναλλακτικές για την δυνατότητα πλήρους δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών που ζουν σε άλλη χώρα από την χώρα της γέννησής τους. Γενικώ από τον Ιανουάριο του 2014 υπάρχει και μια γενική πρόταση έτσι ώστε ε, σύσταση, συγγνώμη, έτσι ώστε ε, να κληθούν τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένου και του, Συμπεριλαμβανομένου και της Μεγάλης Βρετανίας ε, να διευκολύνουν βάσει της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας το δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική στις εθνικές εκλογές εάν και εφόσον εξακολουθούν να δείχνουν ε, ενδιαφέρον για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας ε, συμπεριλαμβανομένου ε, και του εργαλείου της ηλεκτρονικής ψήφου. Θεωρεί η Κομισιόν ότι αυτή η προσέγγιση ήταν μάλλον ισορροπημένη. Παρ' όλα αυτά εξακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί το θέμα. Ωστόσο, όπως και αναφέρθηκε προηγουμένως, αλλά ε, και όπως συζητήθηκε και τον Ιούνιο του 2016 σε αντίστοιχη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών, η Κομισιόν επανέλαβε ότι ε, η σύσταση του εκλογικού σώματος ε, για τις εθνικές εκλογές αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έκτοτε δεν έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στοιχεία σε γνώση της που να την οδηγήσουν σε τροποποίηση των ε, θέσεών της. Πρόεδρος, ε, ξεκινά τώρα η συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων. Κύριε πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και την Επιτροπή. Αλλά ιδιαίτερε ευχαριστίε μου ε, πηγαίνουν στι αναφέρουσε που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα, τις οποίες υποστήριζα από τότε που εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω πραγματικά ότι αν είναι κανεί δημοκράτη θεωρεί τα δικαιώματα ψήφου και τα πολιτικά δικαιώματα ως θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και οποιαδήποτε ιδέα ότι οποιοδήποτε πολίτης υπάρχει περίπτωση να στερηθεί τέτοιων δικαιωμάτων, κάτι που βλέπουμε εδώ να συμβαίνει στην πραγματικότητα με τους Βρετανούς πολίτες οι οποίοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό για πάνω από 15 χρόνια, ε, θεωρώ αποτελεί προσβολή της δημοκρατίας και κατά οποιασδήποτε έννοια θεμελιωδών πολιτικών δικαιωμάτων. Το λέω αυτό ξεκινώντας διότι το έχω συζητήσει με το δικό μου κόμμα, το εργατικό κόμμα, το οποίο έφερε τον κανόνα των 15 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με το σκεπτικό ότι αν ζούσε κάποιο στο εξωτερικό για πάνω από 15 χρόνια, τότε έχει απολέσει τους δεσμούς του με το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει μάλλον χαλαρότερου δεσμούς από τη... με τη χώρα όπου κατοικεί. Αυτό μπορεί να ισχύσει για τι περισσότερε ε, πολιτικέ αποφάσεις, αλλά όταν παρατηρεί κάποιο ότι κάποιο έχει μετακινηθεί εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας το δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τη χώρα μα ω μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξαφνικά βλέπει να υπονομεύονται τα πολιτικά του δικαιώματα εξαιτία του γεγονότο ότι στο άλλο κράτο μέλο δεν του δέχτηκαν ω ανθρώπου που έχουν δικαίωμα ψήφου σε εθνικέ εκλογέ, τότε εκεί έχουμε μια γενιά ανθρώπων ουσιαστικά οι οποίοι έχουν χάσει το δικαίωμα ψήφου του. Ε, τη θεμελιώδη ε, δύναμή τους να εκφράσουν την άποψή τους. Ε, αυτός λοιπόν ο οίκος της δημοκρατίας πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανησυχίες. Όταν εγώ και οι συναδέλφοι μου αναχωρήσουμε από εδώ, από αυτόν τον οίκο, ελπίζω να αντικατασταθούμε από άλλους Βρετανούς βουλευτές. Αυτή είναι η ελπίδα μου, αλλά το πρόβλημα αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Όποιο και αν είναι εδώ, δεν μιλάμε μόνο για τη Βρετανία, μιλάμε για πέντε κράτη-μέλη που έχουν στερήσει τέτοια δικαιώματα από του πολίτε του. Και έχουμε δει διάφορες αναφορές ε, που υπερασπίζονται τα δημοκρατικά δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Το ζήτημα λοιπόν τη ελεύθερη κυκλοφορία και των πολιτικών δικαιωμάτων δεν αφορά μόνο το Brexit και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η όλη υπεράσπιση του κανόνα των 15 ετών ουσιαστικά είναι ε, αυτή η πολιτική η οποία ε, δείχνει τι συνέπειε έχει λόγω του Brexit. Τελικά αυτοί οι άνθρωποι που έφτιαξαν τι ζωέ του σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και οι Ευρωπαίοι πολίτε που αποφάσισαν να φτιάξουν τι ζωέ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και οι δύο αυτέ ομάδε πολιτών παραμελήθηκαν πλήρω. Δεν μπόρεσαν να εκφέρουν άποψη στο δημοψήφισμα. Και οι ζωέ του αναποδογυρίστηκαν. Πολλοί είναι ε, εξαιρετικά ε, προβληματισμένοι, αγχωμένοι για το τι θα συμβεί δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα κοινωνικά τους δικαιώματα, τα οικονομικά τους δικαιώματα, την κατάσταση που θα τους πλήττει στην, ε, την κατάστασή τους στη χώρα που ζουν και εμείς στο Κοινοβούλιο λέμε ότι οι πολίτες είναι η προτεραιότητά μας. Σε οποιαδήποτε θέση υιοθετούμε στην Ολομελία αυτού του οίκου λέμε ότι τα δικαιώματα των πολιτών είναι η κόκκινη μας γραμμή για μια μελλοντική συμφωνία για τον Brexit η συμφωνία που γίνεται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταβατική περίοδο δεν κάνει καμία αναφορά στα πολιτικά δικαιώματα, παρότι το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κάνει αναφορά στα πολιτικά δικαιώματα. Έχουμε το δικαίωμα ω Ευρωπαίοι πολίτε να ψηφίζουμε σε ευρωεκλογέ και σε τοπικέ εκλογέ. Είτε ζούμε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είτε ζούμε ε, είτε είστε Ευρωπαίος πολίτης και ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξαφνικά τεινάσσονται στον αέρα όλα αυτά τα δικαιώματα λόγω της ε, κοινή συμφωνίας και διότι ε, κάποιος υποβάθμισε αυτή την ιδέα και είπε ότι απλά είναι εθνική αρμοδιότητα. ενώ ε, επανειλημμένω έχει υποθεί ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά του Ευρωπαίου πολίτε και του Βρετανού πολίτε και πρέπει να επιληθεί και σα παρακαλώ, σα εκλυπαρώ να το πάρετε σοβαρά. Περνάει ο χρόνο, οι διαπραγματεύσει για το Brexit έχουν στόχο να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο φέτο. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Σα εκλυπαρώ λοιπόν, α απευθύνουμε μια προφορική ερώτηση εκ μέρου τη Επιτροπή μα στην Ολομέλεια για να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του Brexit. Λαμβάνοντας, εκλαμβάνοντας όλες αυτές τις αναφορές ως ένα κομμάτι. Παρότι είχαμε και αναφορές από Ευρωπαίους πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που μας επιτρέπει να συντάξουμε μια προφορική ερώτηση που θα καλύπτει και τις δύο ομάδες πολιτών. Κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι για αυτές τις ανησυχίες. Εξετάζεται νομοθεσία στο Westminster για τον κανόνα των 15 ετών. Έχει την υποστήριξη της κυβέρνηση. Ελπίζω έτσι να καταργηθεί αυτός ο κανόνας των 15 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά όπως είπε και Τζάκη, δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτή την νομοθεσία για οποιοδήποτε δημοψήφισμα. Και δεν υπάρχει... Πιστεύω εγώ ότι όλο ένα και περισσότεροι Βρετανοί αντιλαμβάνονται πώς ε, θα εξελιχθούν οι ζωές τους μετά από το Brexit. Όπως αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τις ζωές των υπέρμαχων του Brexit, όλο και περισσότερο το κοινό θεωρεί ότι πρέπει να εκφέρει μια άποψη για την τελική συμφωνία, να υπάρξει μια ψήφος του λαού για την τελική συμφωνία και η ιδέα ότι οι άνθρωποι θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτή τη... Συγγνώμη, έχω συγκινηθεί διότι μιλάμε για φίλους μου, για συγγενείς μου. Η ιδέα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι για άλλη μια φορά δεν θα μπορέσουν να εκφέρουν άποψη σε κάτι που θα επηρεάσει τις ζωές τους τόσο πολύ είναι προσβολή για οποιονδήποτε ονομάζεται πολίτης δημοκρατικός. Σισίλια πρέπει να δράσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη. Δεν μπορούμε να το παραμερίσουμε. Δεν μπορούμε να το αναθέσουμε σε κάποιον άλλον. Ούτε θα το αφήσουμε στα χέρια Εμείς Επιτροπή υπερασπίζουμε τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη και εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση και εγώ μιλώ εκπροσωπώντας τους γιατί έχουμε κάποια εξουσία, έχουμε φωνή και πιστεύω ότι πρέπει να γράψουμε να απευθύνουμε επιστολή στην Βρετανική κυβέρνηση και να ζητήσουμε να συμπεριληφθεί αυτό στη Συμφωνία Αποχώρησης. Να ε, υπάρχει μια εγγύηση για του Ευρωπαίου πολίτε στο Ηνωμένο Βασίλειο και για του Βρετανού πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να του εγγυηθούν αυτά τα δικαιώματα. Είμαστε ένα χρόνο πριν από τι ευρωεκλογέ και έχει έρθει η ώρα επιτέλου. Είναι κατάλληλη στιγμή για να πούμε κάτι. Ευχαριστώ. Thank you, Jude. And I cannot think... Ευχαριστώ πολύ, Τζουντ. Δεν έχω ακούσει κανένα να είναι τόσο συναισθηματικός αλλά και συγκεκριμένος. Ίσως τη γιαγιά σας, η οποία έκανε μια καταπληκτική δήλωση αμέσως μετά το Brexit δεν θα την ξεχάσω. Ε, δείτε ακριβώς το τι είχε πει. Έχει μεγάλη σημασία. Περνάω στους υπόλοιπους ομιλητές, η Άγγελα. Μετά από αυτά τα οποία είπε η Τζουντ δεν νομίζω ότι μένουν πολλά να υποθούν. Νομίζω ότι έχουμε ουσιαστικά μια μελέτη των επιπτώσεων για το Brexit και εκεί λέγεται ότι πρέπει να υπάρξουν ακριβώς τα σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών και υπάρχει και μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με το Brexit. Νομίζω ότι έχουμε σαν στόχο μέσω και αυτών των αναφορών να στηρίξουμε τα δικαιώματα των προσώπων και των οικογενειών τους και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και την προστασία των πολιτών των υπολείπων πολιτών. Θυμίζω ότι ε, θα μπορούσαν ε, δύο εκατομμύρια άνθρωποι να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές στην Ισπανία, επειδή ζουν εκεί. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι <clears throat> εμείς πρέπει να δώσουμε εγγυήσει για την ελεύθερη διακίνηση, για τη δημοκρατία, για το άνοιγμα του ενός τον και δεν θα πρέπει να υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήταν αντιφατικό με αυτά τα οποία εμείς κάνουμε. <clears throat> θα συμφωνήσω λοιπόν με τις προτάσεις οι οποίες έκανε, τις οποίες έκανε η Τζούντ και θα στηρίξω την αναφορά να μείνει ανοιχτή. Ο κύριος Τέρι Κάμπρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που ζητά ε, που ζητούν οι αναφέροντες. Είπατε εξ ονόματός μας ότι καλό θα ήταν να είχαμε, ότι μάλλον εκτιμούμε για τρίτη, παρουσία για τρίτη φορά ε, της ε, πρώτης ε, αναφερόμενας. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι πρέπει να έρθει και τρίτη φορά, ε, δεν είναι και πολύ ωραίο και δεν ε, μας ενθουσιάζει με την έννοια ότι πρέπει διαρκώς να επιμένει και να ξαναεπιμένει για κάτι που αποτελεί απλώς το δικαίωμά της και είναι πολύ το σωστό. Η δημοκρατία όπως γνωρίζουμε όλοι δεν αφορά μονάχα την ψηφοφορία ή τις εκλογές. Αν και μερικές φορές σε μερικές χώρες και αυτό είναι το αρνητικό, ε, η δημοκρατία εξαντλείται στο δικαίωμα ψήφου και όχι στο διάλογο κτλ. Ωστόσο, Ωστόσο και η στιγμή των εκλογών είναι μια σημαντική στιγμή ε, της δημοκρατικής διαδικασίας και επομένως ε, είναι σοκαριστικό να βλέπει κανείς τέτοιες καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να έχει μία παρουσία λίγο πιο ε, δραστήρια, proactive. Να ζητήσουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο να συμπεριλάβει ε, αυτά τα αυτό το δικαίωμα ψήφου στο τελική συμφωνία, στο τελικό deal που θα γίνει και στον κατάλογο με τις επιθυμίες της κάθε πλευράς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν έχει κανείς δύο αξίες ε, ή δύο αρχές, ε, το δικαίωμα ε, ψήφου και το δικαίωμα κυκλοφορίας, δεν είναι δυνατόν το ένα δικαίωμα να υπερισχύει του άλλου ή μάλλον το ένα να έρχεται σε αντιπαράθεση με το άλλο. Πρέπει να έχουμε και το δικαίωμα να μετακινούμαστε και το δικαίωμα να ψηφίζουμε. Και δεν πρέπει κανείς να πέσει στην παγίδα να πιστεύει ότι η προσθήκη δικαιωμάτων θα μειώσει το σεβασμό στα αρχικά δικαιώματα του ναντίωνα. Πολύ σωστά Πολύ καλά τα λέτε, γιατί είτε σέβεται κανείς κάποιο δικαίωμα, είτε δεν το σέβεται. Ε, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ναι, αλλά πρέπει να γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα. Αυτή πρέπει να είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τάνοκ, ορίσατε. Σας δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω τους ε, αναφερόμενους πριν από έξι μήνες ε, είχαμε συζητήσει με τον Σάντρο Φερχόφστατ ε, το θέμα του δικαιώματος που ε, πρέπει να διατηρήσουν οι πολίτες όσον αφορά τα εκλογικά τους δικαιώματα και μάλιστα το συμπεριλάβαμε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου και σε ένα ψήφισμα, αλλά μετά δυστυχώς αφαιρέθηκε. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι απολύτως κατά του Brexit, αλλά ε, από την άλλη πλευρά ε, εάν ε, ε, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από το Brexit θα πρέπει να ξαναδούμε πώς θα είναι τα πράγματα στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων. Είναι γεγονός ότι δεν είχαμε την δυνατότητα σε επίπεδο 27 κρατών να συμφωνήσουμε για αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι έχω και ένα προσωπικό πρόβλημα. Δηλαδή οι δύο αδερφές μου και η μητέρα μου ε, και ο θείος μου ε, έχουν χάσει ε, το δικαίωμα και δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα για το Brexit είχαν, γιατί το κόμμα μου το 2015 άλλαξε, δεν, δεν μπόρεσε να αλλάξει το, τον νόμο και ε, ε είπαν ότι δεν υπήρχε χρόνος ε, για να ε, αλλάξει ο νόμος. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αληθές, γιατί φαίνεται ότι ε, ακόμα και μέλη της Βουλής των Λόρδων δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις ε, γενικές εκλογές και πολίτες ε, του Γιβραλτάρ επίσης δεν ψήφισαν στις γενικές εκλογές. Δηλαδή μπόρεσαν μέσω κάποιων αλλαγών να ψηφίσουν οι κάτοικοι του, οι πολίτες του Γιβραλτάρ αλλά δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν κάποια μέλη της Βουλής των Λόρδων. Επίσης ε, είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι ήταν αντίθετοι με μια πολύ γενική επέκταση του δικαιώματος ε, γιατί φοβήθηκαν ότι θα σήμαιναν και κάποια άλλα προβλήματα. Ας πούμε, εάν ε, στη Νέα Ζηλανδία επίσης αν ε, φύγεις και δεν ζεις πια στην ε, Νέα Ζηλανδία πρέπει κάθε τόσο να ξαναπηγαίνεις να επισκέπτεσαι τη χώρα έτσι ώστε να δείξεις ότι έχεις τους ε, δεσμούς γιατί διαφορετικά εάν θεωρηθεί ότι έχεις χάσει κάθε επαφή με τη χώρα τότε δεν έχεις και δικαίωμα ψήφου. η, νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν κάποιες νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε κάποιο τρόπο έτσι ώστε ε, οι ε, Βρετανοί που ζουν αλλού στην Ευρώπη να μπορούν να ψηφίσουν. Ε, και η και οι Κύπροι όταν φεύγουν να εγκαταλείπουν την Κύπρο χάνουν το δικαίωμα ψήφου. Από την άλλη μεριά μπορούν να ψηφίσουν σε κάποιες Βρετανικές εκλογές από τη στιγμή που είναι μέρος του Commonwealth. Και mm ε, επίσης, άλλες χώρες οι οποίες έχουν ενδεχομένως ε, την Αγγλική ως επίσημη γλώσσα μπορούν να ε, μπόρεσαν να ψηφίσουν μέσω των πολιτών τους στο δημοψήφισμα. Κοιτάξτε, τώρα τα λέμε όλα ξεκάθαρα. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει δικαίωμα ψήφου σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σε δημοψηφίσματα λόγω λόγω του θέματος ε, της Σκοτίας ε, και ε, γι' αυτό είδαμε τι αντίκτυπο είχε η ψήφος τους στο θέμα του δημοψηφίσματος της Σκοτίας και επομένως γι' αυτό ήταν λίγο διστακτική στο να επεκτείνουν τα δικαιώματα. Εν πάση περιπτώσει ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ε, μία γενική ανησυχία και κάποιο άγχος όσον αφορά αυτές τις ε, ψήφους και την παροχή δικαιώματος γιατί θεωρούν ότι ενδεχομένως δυναμητίζεται κάπως η κατάσταση και όσον αφορά το Brexit. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει της συνθήκης λειτουργίας και καταπατώνται τα δικαιώματα αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκα. Ο κύριος Μασελέζη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους αναφερομένους, τις αναφερόμενες μάλλον, συζητάμε θέματα όπως το δικαίωμα ψήφου, τα πολιτικά δικαιώματα, όλα αυτά τα πολιτικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα, είναι θέμα λοιπόν αρχής, είναι ένα θέμα δημοκρατίας και ποιότητας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Για μένα σήμερα είναι εντελώς ακατανόητο κάποιοι πολίτες που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζουν σε μια άλλη χώρα να μην έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ή περιφερειακές εκλογές. κάποιος να μου εξηγήσει πώς ο Τζάκι Κοτερίλ ας πούμε μπορεί να είναι σύμβουλος δημοτικής στην Ισπανία αλλά δεν μπορεί να είναι βουλευτής ή μπορεί να είναι ευρωβουλευτής της Ισπανίας αλλά να μην είναι βουλευτής. Τώρα δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εμείς ότι υπάρχει το δικαίωμα ψήφου για όλους τους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στην Ευρώπη ανεξαρτήτως χώρας. Το δικαίωμα αυτό είναι θεμελιώδες και πρέπει να το διεκδικήσουμε. Και υπάρχουν και χειρότερα, διότι υπάρχουν ε, πολίτες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στη Μάλτα κτλ που έχουν απολέσει το δικαίωμα να ψηφίζουν σε οποιαδήποτε χώρα. Δεν μπορούν να ψηφίσουν δηλαδή στη χώρα προέλευσής τους, δεν μπορούν να ψηφίσουν και στην χώρα παραμονής τους και υποδοχής. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτε μας σήμερα. Ε, αν θέλουμε να έχουμε μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρούμε λύσεις. Και τι να πούμε για το Ηνωμένο Βασούλιο λοιπόν. Για το Ηνωμένο Βασίλειο ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν το δικαίωμα ψήφου σε μια την πιο σημαντική αν θέλετε εκλογική διαδικασία, δημοψηφισματική διαδικασία της ζωής τους εξαιρέθησαν από την <clears throat> ψηφοφορία για το δημοψήφισμα. Ελπίζω λοιπόν στο επόμενο να μπορέσουν να ψηφίσουν. Και θα ήθελα να θέσω τις εξής ερωτήσεις. Μιλάμε για το δικαίωμα ψήφου και στις ευρωεκλογέ και στις εθνικές εκλογές. Πρέπει να στείλουμε λοιπόν μια επιστολή ζητώντας κοινά κριτήρια για τους κατοίκους μιας χώρας και προς την Προεδρία, τη Βουλγαρική Προεδρία και προς τις μόνιμες αντιπροσωπείες έχει πάρα πολύ σημασία να γνωρίζουν ποιο είναι το πρόβλημα και να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις και σε σχέση με την πεφορική ερώτηση η οποία έχει ήδη προταθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος να στείλουμε μία επιστολή στη Βρετανική κυβέρνηση αμφισβητώντας τις αποφάσεις αυτές και επίσης μία επιστολή στο Μισελ για να είναι ξεκάθαρη η πολιτική θέση μας στις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστώ. Το θέμα είναι ξεκάθαρα δημοκρατικό. Τώρα έχουμε αρχίσει να καθυστερούμε και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Στέιλα. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί έρχονται ήδη αναφερόμενοι και δεν είναι σωστό να μην τους δώσουμε το λόγο. Σύμφωνο απόλυτα μαζί σα ε, και συμφωνώ. Θέλω να υποστηρίξω τα όσα είπαν οι αναφερομένε ε, και οι συναδελφοί μου. Ο Τσάρλ ανέφερε αυτό που θέλω να πω ότι στο σκοτσέζικο δημοψήφισμα θα δώσουμε το δικαίωμα ψήφου σε Ευρωπαίου πολίτε, Οπότε μπορούν να υπάρχουν διαφορετικά δικαιώματα σε διάφορε χώρε, Γιατί δεν το είχαμε ρυθμίσει αυτό πριν από το δημοψήφισμα για την ιδιότητα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Δεν το πιστεύω. Θέλω να το αναφέρουμε στην Ολομέλεια Εκεί θα γίνει ευρύτερη συζήτηση και εκεί θα ακουστούν οι φωνές μας σε τόσο σημαντικές στιγμές. Είναι, εγώ ξέρετε, σε λίγο θα χάσω την ευρωπαϊκή μου Γεννήθηκα το 1973 και θα χάσω την ευρωπαϊκή μου ταυτότητα λόγω μιας ψηφοφορίας που πολύ ειλικρινά έγινε υπό συνθήκε ποιος ξέρει με ποιες επιρροές, από ποιες επιχειρήσεις. Ε, ε, είναι πολύ σημαντικό και η, στιγμή, η κύρια στιγμή είναι τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τζακλίν, να ξαναέρθω σε εσά και στην Κριστίν. Έχετε χρόνο και μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Να προσθέσετε κάτι που δεν υπόθηκε, γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα, σχεδόν τα πάντα, έχουν υποθεί. Ναι, ευχαριστώ. Άκουσα πολλέ φορέ αυτή την επίσκεψη στο Κοινοβούλιο ότι υπάρχει κάποια κόποση σχετική με το Brexit, ότι είναι πολύ αργά να υπερασπιστούμε του Βρετανού πολίτε Γι' αυτό ή για άλλα ζητήματα. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα συνεχίσουν να αναγνωρίζουν ότι η ηθαγένειά μα εξακολουθεί να είναι ευρωπαϊκή και ότι θα διατηρήσουμε τα δικαιώματά μα μέχρι το τέλο. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτε. Ακόμη σήμερα εξακολουθούμε να έχουμε όλα μα τα δικαιώματα. Και ελπίζω να μην τα χάσουμε με ενθαρρύνουν οι απαντήσει σα σήμερα αγαπητοί βουλευτέ. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σα, ειδικώ εσεί, κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ για την πολύ συναισθηματική σα παρέμβαση. Δείχνει πόσο συναισθηματικά φορτισμένο είναι το ζήτημα του Brexit ε, μαζί με τι πρακτικέ του πτυχέ. Ελπίζω το Κοινοβουλίο να κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το ζήτημα που δεν επηρεάζει μόνο εμά ε, το Brexit αγγίζει την καρδιά των δημοκρατικών διαδικασιών της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Σα ευχαριστώ όλους. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι πέραν του ότι νιώθω καταπληκτικά που επιτέλους κάποιος άκουσε αυτό που είχα να πω. Διότι στο δημοψήφισμα δεν μπόρεσα να πω αυτό που ήθελα. Ξέρετε, κάποιες στιγμές αισθάνομαι περήφανη που είμαι πρόεδρος αυτής της ε, Επιτροπής. Μερικές φορές είναι δύσκολο, αλλά πάντα είναι σημαντικός πιστεύω ο ρόλος μου και αυτή είναι τέτοια στιγμή, στιγμή όπου είμαι περήφανη που βλέπω ότι αυτή η Επιτροπή μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει η Επιτροπή αυτή ως γέφυρα μεταξύ πολιτών κυβερνήσεων και ούτω καθεξής. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι είναι δυνατόν για να γεφυρώσουμε το χάσμα το οποίο βλέπουμε εδώ. Ας ε, εξάγουμε ένα συμπέρασμα από όλα αυτά για το τι θα κάνουμε. Να επιστήσω την προσοχή σας στην επικαιροποιημένη μελέτη. Πάρτε μαζί σας ένα αντίτυπο, μην το ξεχάσετε πριν φύγετε από την αίθουσα. Και φυσικά θα διατηρήσουμε ανοιχτέ τι αναφορέ και προτείνω να τις στείλουμε στην ε, διοικητική ομάδα για τον Brexit ώστε να τις λάβουν υπόψη στις τρέψεις διαπραγματεύσεις αλλά και όταν θα εκπονηθεί το επόμενο ψήφισμα και εκεί πιστεύω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης πρέπει να σταλεί μια επιστολή στην Βρετανική κυβέρνηση στο Μισελ Μπαρνιέ και ενδεχομένω και στην Προεδρία, όπω όπως κάποιο κάποιος πολύ σωστά, υπάρχουν πέντε κράτη-μέλη που κάνουν την ίδια, ε, ακολουθούν την ίδια τακτική. Πρέπει να το δούμε λοιπόν. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα δικαιώματα ψήφου θα συμπεριληφθούν στην τελική συμφωνία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβεί αυτό. Όπω γνωρίζετε, ο Μισελ Μπαρνιέ δεν επιτρέπεται ή μάλλον έχει συμφωνηθεί να μην έρχεται σε επιτροπές Τίποτα όμως δεν με εμποδίζει να του μιλήσω εγώ. Ούτως ή άλλως συνομιλώ μαζί του και συχνά μάλιστα. Και αν μου δώσει ε, κάποια άποψη ότι καλό θα ήταν να το συζητήσουμε και την επόμενη, στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων, ευχαρίστω. Ναι. Όσον αφορά την προφορική ερώτηση όμως, δεν μπορούμε να λάβουμε σχετική απόφαση αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ καλή ως ιδέα, αλλά όπως γνωρίζετε οι συντονιστές πρέπει να λάβουν τέτοια απόφαση. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε όλοι σας, πηγαίνετε στον δικό σας συντονισμό, στη δική σας πολιτική ομάδα και φροντίστε να τους πείστε να το θέσουν ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση συντονιστών. Και ευχαριστώ να το ξανασυζητήσουμε, εφόσον το επιθυμεί η Επιτροπή. Με αυτό ε, θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου εκ μέρους της Επιτροπής προς όλους εσάς που ταξιδέψατε μέχρι εδώ για να μα πείτε ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα και από παλιότερα. Μερικέ φορέ πρέπει να επαναλάβει κανεί τα ίδια και τα ίδια. Αλλά ξέρετε τελικά ο σκοπό που επιδιώκεται είναι θεμητό. Και ελπίζω να νικήσετε. Η νίκη είναι στα χέρια σας, ελπίζω. Ευχαριστώ λοιπόν που βρεθήκατε εδώ. Καλή επιστροφή. Και θα συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο σημείο. Το Εργαστήριο Μελέτης για τα Πολιτικά και τα Εκλογικά Δικαιώματα των Λαδαπών Κατοίκων στη Λετωνία και την Εστονία. Το εργαστήριο αυτό οργανώθηκε από το Θεματικό Τμήμα Πολιτικής ΓΑΜΑ για την Επιτροπή μας. Και ας ξεκινήσουμε αμέσως γιατί έχουμε χάσει λίγο χρόνο. So, dear colleagues, uh, speakers... Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ομιλητές συμμετέχοντες με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω εδώ σε αυτό το εργαστήριο που οργάνωσε το θεματικό τμήμα ΓΑΜΑ για την Επιτροπορών μετά από έτοιμά μας. Κάποιες τεχνικές πληροφορίες. Η διερμηνία υπάρχει σήμερα σε, και στις 24 επίσημες γλώσσες με κάποιες εξαιρέσεις. Τα τσεχικά, κροατικά, φιλανδικά, πορτογαλικά, σλοβακικά και σλοβένικα δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή. Να γνωρίζετε ότι το εργαστήριο αυτό μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο και θα εγγραφούν, θα ε, μαγνητοσκοπηθούν οι παρεμβάσεις των ομιλητών. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και εμπειρογνώμονες ε, να μας πούν τις απόψεις τους ε, για το θέμα των πολιτών αυτών της Λετωνίας και της Εστονίας ή των μη πολιτών. Δεν θα συζητήσουμε επιμέρους αναφορές στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ούτε θα λάβουμε αποφάσεις. Η απόφαση για την αναφορά 747 του 2016 για τα πολιτικά δικαιώματα Λετωνών και Εστονών ε, μόνιμων κατοίκων που δεν είναι ε, υπήκοοι θα λάβει χώρα ε, μετά από το εργαστήριο και όχι κατά τη διάρκειά του. Σήμερα έχουμε εμπειρογνώμονες ακαδημαϊκούς που θα μας προσφέρουν τρία ενημερωτικά έγγραφα για τα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματα των επωνομαζόμενων μόνιμων κατοίκων μη πολιτών, μη υπηκών στη Λετωνία και στην Εστονία. Χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει κάποια νομικά καθεστώτα του μη ε, πολίτη στη Λετωνία και του ε, ακαθόριστης ταγένειας στην Εστονία. Κάτι μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πολύ συναισθηματικό και επίμαχο ζήτημα αυτό το ζήτημα της ηθαγένειας στις χώρες αυτές. Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να περιγράψουμε τις συνθήκες, το πλαίσιο και τις εξελίξεις ε, για αυτό το θέμα της υπηκότητας ε, στη, Λιθουαν... Λετωνία και στην Εστονία. Εστιαζόμενοι ειδικότερα στην κατάσταση των εκλογικών και πολιτικών δικαιωμάτων των μη υπηκών μόνιμων κατοίκων στη Λετωνία και στην Εστονία με μια ιστορική, κοινωνιολογική και νομική ε, οπτική γωνία. Το εργαστήριο θα μας βοηθήσει, ελπίζουμε, να καταλάβουμε και το πλαίσιο 0707 ε, του 2007 της ε, αναφοράς 0707 που ανέφερα ε, και η συζήτηση όπως είπα θα ξεκινήσει αμέσως μετά από την ακρόαση αυτή η αναφορά αριθμός 747 του 2016 δίνω το λόγο στον πρώτο ομιλητή από το Πανεπιστήμιο της Ζηρίχης ε, στην κυρία Τόμσμαν συγγνώμη η οποία θα μας παρουσιάσει την κατάσταση της απόψη ηθαγένεια, τη πολιτογράφηση και τη υπηκότητα στη Λετωνία και στην Εσθονία. Και με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω εδώ στην Επιτροπή. Σας δίνω το λόγο για 20 λεπτά. Okay. Okay. Great. Thank you very much. Um, thank you very much for the uh, for the kind introduction uh, and. Ευχαριστώ πολύ για την uh, πρόσκληση την οποία μου απευθύνετε την εκτιμώ ιδιαίτερο. Ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει για να οργανωθεί αυτή ε, η ε, συζήτηση. Είμαι Γερμανίδα, ζω τώρα στην Ελβετία ε, και είμαι υπέρμαχος θερμότατη της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Σήμερα θέλω να σας κάνω μια παρουσίαση η οποία θα βασίζεται σε κάποια, θα περιστρέφεται μάλλον γύρω από κάποια στοιχεία. Γιατί είναι σημαντική ε, η ε, ηθαγένεια, ε, επίσης κάποια ιστορία όσον αφορά την Εστονία γιατί είναι ε, τόσο αργή η διαδικασία της ε, πολιτογράφησης ε, και επίσης γιατί θέλει κάποιος να αποκτήσει την την πόλη, την, την ηθαγένεια. Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, και επομένως πρέπει να συζητηθούν. Ε, υπάρχει ε, μια ιδέα ότι έχει κανείς το δικαίωμα να έχει δικαιώματα και άλλα βέβαια πριν από οποιοδήποτε δικαίωμα πρέπει κανείς να έχει ακριβώς την ηθαγένεια. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη αρχή. Εγώ προτείνω ε, την ανάγνωση που έχουν κάνει και άλλοι πριν από μένα, δηλαδή ότι η ηθαγένεια είναι ένα, ε, ε, ένα σύνολο που αφορά τα δικαιώματα, την, την συμμετοχή, πρακτικές αλλά και υποχρεώσεις. Και σε πολλές περιπτώσεις τα κοινωνικά δικαιώματα ας πούμε είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά μπορούν να διευκολυνθούν από την ηθαγένεια. Ένα άλλο θέμα ε, είναι ότι ε, το να έχεις την ηθαγένεια σημαίνει ότι συμμετέχεις κάπου, σε μια ομάδα, σε μια διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες ε, είναι συνδεδεμένοι με τους δε, έχουν ε, κάποιες, κάποιους ε, δεσμούς και ενδεχομένως έχουν την ίδια ας πούμε την, την ίδια αίσθηση ότι ανήκουν σε κάποιες φανταστικές εντός εισαγωγικών κοινότητες. Ε, αυτά είναι στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά τα οποία αποτελούν ε, την ιστορία ή την ε, καταβολή των ανθρώπων. Επίσης, κάποια από τα δικαιώματα που έχουμε έχουν προκύψει από τις πρακτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί. Οι υποχρεώσεις τώρα που είναι το τελευταίο που αναφέρω εδώ σε στοιχείο της ηθαγένειας είναι ας πούμε ε, η στρατιωτική θητεία έστω και αναφορά μονάχα τους άντρες ε, είναι το, η καταβολή των φόρων ε, είναι επίσης η ε, σωστή αντιμετώπιση του κράτους ε, με την έννοια ε, του κράτους το οποίο ανήκει κάποιος. Ε, δηλαδή αυτό το είδος της πίστης που πρέπει να δείχνει κανείς προς την χώρα στην οποία ανήκει. Επίσης, ε, σημαίνει ότι ε, δεχόμαστε και κάποια στοιχεία τα οποία απορρέουν από το κράτος χωρίς να τα αμφισβητούμε συστηματικά όπως δεχόμαστε ας πούμε ότι τα παιδιά δεν έχουν όλων των ειδών ε, τα δικαιώματα. Και φυσικά αυτές οι αρχές αλλάζουν. Αυτές οι τέσσερις ε, αρχές ε, των ε, δικαιωμάτων, των πρακτικών, των υποχρεώσεων και της, του ανήκειν είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία αφορούν την ηθαγένεια και που εάν δεν υπάρχουν μπορούν να αποκλείσουν κάποιους πολίτες, κάποια άτομα. και είπα βεβαίως και προηγουμένως ότι η ηθαγένεια είναι ε, αραγώς συνδεδεμένη με την δημοκρατία. Ένας άλλος τρόπος ε, ε, αντιμετώπισης της ε, ηθαγένειας είναι να το δει κανείς, να την δει την ηθαγένεια κανείς σαν μία σχέση ανάμεσα, μία σχέση σαν μία σύμβαση ας πούμε, συμβατική σχέση με δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ανάμεσα στο άτομο και το κράτος. Θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτήν την έννοια αργότερα για να δούμε ακριβώς το, τη, συγκεκριμένη περίπτωση της Λετωνίας και της Εστονίας γιατί νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις σημερινές ε, πολιτικές. Γιατί είναι σημαντική η ηθαγένεια σε αυτή την ερώτηση μπορώ να πω ότι σημαίνει ότι τα άτομα μετρούν, είναι υπολογίσιμα, ε, συμπεριλαμβάνονται ε, και είναι σημαντικό όμως θέμα η ηθαγένεια και για τα κράτη, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμπεριλάβουν ή να αποκλείσουν άτομα. Από τη στιγμή που ε, έχουμε πει ε, λοιπόν ότι και έχουμε καθορίσει ότι η ηθαγένεια είναι κάτι σημαντικό, θα πρέπει να δούμε και τα πρακτικά στοιχεία. Αν δει κανεί πώς έχουν τα πράγματα στην Λετωνία και την ε, Εστονία, είναι ε, καλό να τα ε, θυμίσουμε. Ε, ήταν μέλη η Εστονία, μέρη Εστονία και η ε, Λετονία ε, της ε, Ένωσης των Σοβιετικών Δημοκρατιών αλλά είχαν ανεξάρτητο καθεστώς από το 1918 μέχρι το 1940 και όσοι ήταν πολίτες το 1940 έγιναν πολίτες αυτής της νέας χώρας με την αποκατεστημένη ας πούμε ε, δημοκρατία. Ο... Όμως η σύσταση, η σύνθεση του πληθυσμού άλλαξε στη διάρκεια της σοβιετικής επιρροής. Είχα εδώ κάτι γραφήματα. Α, να, είναι κάποια στοιχεία όσον αφορά τη δημογραφική ε, σύνθεση αναεθνότητα της Εστονίας. Βλέπετε ότι από το 35 μέχρι το 1989 υπήρξε μια ε, σημαντική ε, τροποποίηση της σύνθεσης. Βλέπετε ότι ο λετονικός ε, πληθυσμός έπεσε στο 52% το 1989 και αν δούμε και την Εστονία δεν είναι τόσο μεγάλη η μείωση αλλά πάντως ε, έχει αλλάξει η σύνθεση του πληθυσμού. Εδώ βλέπουμε επίσης ότι οι χώρες αυτές ε, δεν είχαν ομοιογένεια. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Το 1991 τα πράγματα άλλαξαν ε, και επομένως τι πρέπει να κάνει το κράτος. Ε, συνήθως ξέρουν ποιοι είναι οι πολίτες τους αλλά από τη στιγμή που υπήρξε αυτή ε, η μεγάλη διαφοροποίηση, αυτή η καμπή, ε, ε, σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Και τότε αποφασίστηκε ότι όποιος είχε το δικαίωμα παραμονής μπορούσε να γίνει πολίτης. Και επομένως οι άνθρωποι οι οποίοι στη δεκαετία του 50, του 60, του 70 είχαν μετακινηθεί και είχαν εγκατασταθεί στις χώρες της ε, Βαλτικής δεν μπορούσαν να έχουν δικαίωμα ε, στην ηθαγένεια και αυτό ε, και ούτε και τα παιδιά τους βέβαια και αυτό ήταν κάτι περίεργο, ιδιαίτερο μάλλον. Το 1995 ε, αποφάσισαν οι χώρες αυτές να δημιουργήσουν ε, μία διασύνδεση ε, με μία άλλη δομή, την οποία διασύνδεση συνήθως καλύπτει η ηθαγένεια. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η ηθαγένεια μπορεί να σημάνει συμπερίληψη ή αποκλεισμό και ακριβώς η ιστορία χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να συμπεριληφθούν κάποια άτομα και ώστε να αποκλειστούν κάποια άλλα. Επίσης σήμαινε ότι στην αρχή του 90 όπου υπήρχαν πολλές ασάφειες ε, Βέβαια το 2004, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Μιλήτρια, έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον ε, η Εστονία και η Λετωνία, αλλά τότε ε, ακόμα ήταν πολύ μακρινά, το 90-92 ήταν ακόμα πάρα πολύ μακρινά ε, όλα αυτά. Βλέπετε εδώ ότι στην αρχή στη Λετωνία περίπου 30% δεν ήταν πολίτες, λίγο λιγότερο από 30% στην ε, Λετωνία και λίγο παραπάνω από 30% στην ε, ε, Εστονία. Έχουμε λοιπόν μια ιδιάζουσα κατάσταση και φαντάζομαι ότι ο επόμενος ομιλητής θα μιλήσει και για τα εθνοτικά ζητήματα. Αλλά θα ήθελα ε, τι σημαίνει ε, non-citizenship status, ε, τι σημαίνει καθεστώς μη ηθαγένειας. Υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με αυτήν την έννοια του απάτριδος. Ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν δικαιώματα, ε, μπορεί σε περίπτωση προβλήματος πραγματικά ε, οι καταστάσεις να γίνουν εφιαλτικές. Ε, αργότερα ε, προσπάθησαν οι χώρες να βρουν κάποια λύση ε, δίνοντας τους απάτριδες το καθεστώς της μη ηθαγένειας με βάση τις οποίες είχαν το δικαίωμα να ταξιδέψουν, να φύγουν από τη χώρα, να επιστρέψουν και να ζήσουν εκεί. Βέβαια είχε, έχει υπάρξει και μια ολόκληρη διοικητική ή ε, συνταγματική διαδικασία, αλλά όλες αυτές είναι πολιτικές ε, διεργασίες οι οποίες ήταν αρκετά αντιφατικές και οι οποίες δεν προχώρησαν εύκολα. Και όπως είπα και προηγουμένως, η κατάσταση ε, στις αρχές της δεκαετίας του 90 ε, ήταν ε, ασαφής, υπήρχαν ακόμα στρατιωτικές μονάδες στο έδαφος των χωρών της Βαλτικής και δεν υπήρχε καθό καμία σταθερότητα και καμία βεβαιότητα. Και ξεκίνησε λοιπόν η, μια διαδικασία πολιτογράφησης. Ε, η πολιτογράφηση είναι μια διαδικασία πολύ κοινή σε πολλές χώρες, ε, είναι, ε, ε εντάσσεται στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η Εστονία λοιπόν και η Λετωνία ξεκίνησαν, θέσπισαν αυτές τις διαδικασίες πολιτογράφησης που συμπεριέλαβαν πολλά στοιχεία. Ε, βασιζόμενες σε, διάφορες, διάφορα κριτήρια όπως ε, είναι ας πούμε ε, το νόμιμο εισόδημα, η γνώση της γλώσσας της χώρας κλπ. Η διαδικασία ήταν αρκετά γρήγορη και προσιτή όσον αφορά το οικονομικό βάρος. βλέπουμε εδώ ότι ο αριθμός των πολιτών ε, σιγά σιγά αυξάνεται και ο αριθμός των μη πολιτών, ε, μη εχόντων δηλαδή την ηθαγένεια, ε, μειώνεται. Βέβαια, θα περίμενε κανείς όλοι οι πολίτες να θέλουν να γίνουν, να αποκτήσουν την ε, ηθαγένεια, θεωρώντας και όλος ότι αυτή η ενδιάμεση λύση της ε, μη ηθαγένειας ήταν ακριβώς μία απολύτως ενδιάμεση ε, λύση. Αλλά το καθεστώς δεν ήταν καθόλου πρόσκαιρο. Και έχουμε ακόμα ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών που βρίσκονται σε αυτό το ενδιάμεσο καθεστώς των μη πολιτών. Γιατί τώρα η διαδικασία πολιτογράφησης είναι αργή ε, οφείλεται σε μια σειρά στοιχείων. Βλέποντας έρευνες και ε, στοιχεία, το θέμα της ε, γνώσης της γλώσσας ε, ήταν ε, πολύ σημαντικό γιατί ας πούμε ε, πιο γυρεοί πολίτες ε, δεν ήταν εύκολο να περάσουν αυτές τις γλωσσικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η γνώση. Το ιστορι... τεστ ιστορίας επίσης και αυτό αναφέρθηκε ως λόγος για τον οποίο κάποιοι απέφευγαν να ξεκινήσουν τη διαδικασία πολιτογράφησης και το θέμα της ε, υποχρέωσης ε, της πίστης προς το κράτος και αυτό ήταν ε, ένα σημαντικό στοιχείο. Υπάρχουν βέβαια και ψυχολογικοί παράγοντες που είναι πολύ σημαντικοί. Ας πούμε το θέμα της ιστορίας. Στην, στις χώρες της Βαλτικής ε, ο τρόπος με τον οποίο ναι, η αντιμετώπιση της ιστορικής πραγματικότητας ε, μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ ε, από πολίτη σε πολίτη. Η αντιμετώπιση της ιστορίας, κυρίως όσον αφορά την διαδικασία ανεξαρτητοποίησης, δεν είναι τόσο σαφής. Επίσης υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μετανάστευσαν εντό εισαγωγικών, μετακινήθηκαν στις χώρες αυτές όταν δεν υπήρχε ακόμα η έννοια της μετανάστευσης και από την μία πλευρά ε, ε θεωρήθησαν και ως ε, κατακτητές. Και επομένως κάποιοι μπορούσαν να σκεφτούν ότι μέσω της πολιτογράφησης, ναι, γίνεσαι μέλος της κοινωνίας στην οποία ζεις, αλλά ε, οι απέξω ε, ε, είχαν την τάση επίσης να πιστεύουν ότι μέσω της πολιτογράφησης θα αρνιόντουσαν τη δικιά τους κατάσταση. Απ' την άλλη πλευρά ε, είναι γεγονός ότι είναι χρήσιμο να έχει κανείς την ηθαγένεια. Μπορεί να ψηφίσει, μπορεί να έχει ε, ε χέρι όλων των δικαιωμάτων. Άρα ήταν χρήσιμο πράγμα και η πολιτογράφηση. Υπήρχε πάντως η αίσθηση ότι αν ας πούμε πολιτογραφούν το, ε, οι πολίτες αυτοί που δεν είχαν την υπηκότητα, την ηθαγένεια μάλλον ε, ε, και γίνονταν πολίτες της Εστονίας ή της Λετωνίας θα έπρεπε μετά ε, να ζητούν βίζα για να πάνε να επισκεφθούν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η, το αρχικό κείμενο υπήρξαν πολλές τροποποιήσεις συμβολές από κάθε πλευρά έτσι ώστε ε, να δημιουργηθεί ένα κανονικό καθεστώς ηθαγένεια. Σε κάποιες πρόσφατες ε, έρευνες ε, κάποιοι δήλωσαν ότι το καθεστώς του non-citizen, ε, του μη ε, πολίτη, ήταν ένα καθεστώς που δεν τους δημιουργούσε ιδιαίτερο πρόβλημα και ότι θεωρούσαν ότι με τον τρόπο αυτό μπορούσαν να ενταχθούν καλύτερα στην κοινωνία. Θα τα πω γρήγορα τώρα, λέει η ομιλήτρια, δεν μου έχουν μείνει πολλά. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα όσον αφορά ε, κάποιες, ε, κάποια προγνωστικά που έχουν γίνει, κάποιες ε, μελέτες προοπτικής. Βλέπουμε ότι ο βαθμός πολιτογράφησης είναι βραδύτερος από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Πάντως, το νόμιμο καθεστώς οπωσδήποτε θα υπερισχύσει Αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό σε τούτη τη συζήτηση είναι ότι το θέμα της ηθαγένειας μπορεί να συζητηθεί σαν νομικό ζήτημα από νομική σκοπιά, ωστόσο αφορά την ίδια, τον ίδιο τον πυρήνα της κοινωνίας. Ε, δηλαδή αφορά, απαντά μάλλον στο ερώτημα τι σημαίνει το ανήκειν σε αυτές τις χώρες τι ε, αίσθηση προκαλεί ε, αυτή η αίσθηση του είναι στους ε, ε, πολίτες που ανήκουν σε αυτήν την ειδική κατηγορία. Είχα κι άλλα να σας πω, αλλά δεν προλαβαίνω. Thank you, Dr. Thank you. Ευχαριστούμε, Dr. Τονσμάν. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Φωτίσατε κάποιες πτυχές αρκετά περίπλοκες για μας. Θα στραφώ τώρα στον Δ. Μάρτιν Παπαρίνσκι από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Θα μας δώσετε μια γενική εικόνα της σημερινής κατάστασης και των προοπτικών για τα εκλογικά και πολιτικά δικαιώματα των Εστονών και Λετωνών μόνιμων κατοίκων που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ για τα ευγενικά σας λόγια κυρία Πρόεδρα. Όπως είπε πολύ σωστά η προηγούμενη ομιλήτρια, μπορεί να δει κανείς το ζήτημα των μη πολιτών με, από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η δική μου οπτική γωνία είναι νομική. Αντικείμενο της παρουσίασής μου λοιπόν, που βλέπετε και στις διαφάνειες ε, συνειδητά περιορίζεται σε στενό πεδίο. Το ζήτημα του εργαστηρίου αυτού και της αναφοράς αφορά το δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογέ για τους πληθυσμούς αυτούς. Εδώ θα εστιαστώ. Και καλό θα είναι να σημειωθεί και αυτό που δεν θα συζητήσω θα συζητήσω, όπως θα έχετε σημειώσει, την ε, παρουσία αυτών των μη πολιτών ε, στη Λετωνία και στην Εστονία. Αυτούς που ονομάζει η Επιτροπή Αντίστοιχους ε, Μη Ιθαγενείς Πληθυσμούς. Δεν θα μιλήσω για τους άλλους μη πολίτες της Εστονίας και της Λετωνίας, ούτε για άλλα παρόμοια πολιτικά και εκλογικά δικαιώματα, ούτε για δικαιώματα κοινοβουλευτικών εκλογών, δημοκρατικών εκλογών, ούτε για άλλα δικαιώματα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι θέμα της συζήτησής μου. Σας προτείνω να ακολουθήσουμε τέσσερα βήματα στην παρουσίαση της έκθεσής μου. Πρώτα θα σας παρουσιάσω τις ε, εστονικές και λετονικές οπτικές γωνίες όσον αφορά τα καθεστώτα αυτά. Βάσει των όσων είπε και η προηγούμενη μιλήτρια, παρατηρείται κάποια ένταση μεταξύ ατόμων που δεν είναι υπήκοοι της Εστονίας και της Λετωνίας και που παρόλα αυτά διαθέτουν ένα εύρος δικαιωμάτων που συνήθως δεν χορηγούνται σε απάτριδες, σε ανηθαγενείς. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τη θέση της Εστονίας και της Λετωνίας επί του θέματος. Μετά θα εξετάσουμε την οπτική γωνία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου. Εδώ θα τονίσω ότι το βασικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι η θέση του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου ότι ο έλεγχος υπό το Διεθνές Δίκαιο ακόμη και αν φέρει αποτέλεσμα, δεν δημιουργεί αναγνωρισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτή η θέση θα πρέπει να σας είναι γνωστή ε, από άλλα πλαίσια ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε την Δημοκρατία της Βορειάς Κύπρου, την Κρυμαία, τι περιπτώσεις της Δυτικής Σαχάρας, ε, για την υπόθεση Πολυσάριο και εδώ αναφερόμαστε στα δικαιώματα ε, Ρώσων ε, ε, απίκων και των απογόνων τους. Το τρίτο σημείο που θα αναφέρω σχετίζεται με την οπτική γωνία της, νομοθεσίας περί της Διεθνούς Νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποιο είναι ο χαρακτήρας αυτής της μη... του μη σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών των ε, πληθυσμών. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο πιθανοί και δύο ε, λογική τρόπο να διαβάσει κανείς, ε, να καταλάβει κανείς αυτό το καθεστώς. Το πρώτο ε, είναι το να δούμε το καθεστώς ως κάτι γενικό, ως προτείνει το συνταγματικό δικαστήριο της Λετωνίας είναι θεωρηθούν απάτριδες όπως προτείνουν κάποια ανθρωπιστικοί οργανισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο για τους σκοπούς της συζήτησής μας νομίζω ότι όποιο εδώ και να ακολουθήσουμε καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή ότι είτε το αντιληφθούμε και το καθαρίσουμε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο ή μάλλον με κανέναν από τους δύο τρόπους δεν αφαιρεί τα δικαιώματα επικότητας από τα άτομα αυτό ε, ούτε από το δικαίωμα του να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ. Τέλος, θα δούμε την οπτική γωνία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και εγώ κάπως βαρετά θα κλείσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο. Δίθεται το νομικό θέμα, μεν, ε, παραβίαση του τρέχοντος καθεστώτος. Ταυτόχρονα, όπως βλέπουμε και από την ομολογία του Ηνωμένου Βασιλείου, τα κράτη-μέλη μπορούν να λαβούν την απόφαση να επεκτείνουν το δικαίωμα ψήφου στους ε, ε, μη Αυτό είναι επιλογή πολιτικής αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως είναι αυτονόητο. Είχε υποθεί κάποτε ότι τα άρθρα 9 και 10 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προβλέπουν ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πήκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της των κρατών μελών, συγγνώμη, είναι υπήκοοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, συνεπώ έχουν δικαίωμα ψήφου στι ευρωεκλογέ. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί στην Εστονία και τη Λατωνία μας οδηγούν σε άλλο συμπέρασμα. Ποιο είναι το παρελθόν ε, στην Εστονία και στη Λετωνία. Δεν θα σας μιλήσω ως εκπρόσωπος κράτους, αλλά τι τελευταίε δεκαετίες αυτές οι θέσει έχουν παγιωθεί που θα σα αναφέρω τώρα. Εγώ έχω δεχθεί στι εκθέσει μου προ τα Ηνωμένα Έθνη ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, βάσει αυτών των θέσεων. Υπάρχουν κάποιε ομοιότητε και κάποιες διαφορές. Η σχετική έκθεση εξετάζει περαιτέρω λεπτομέρειες των θεμάτων αυτών. Όπως είπα, οι ομοιότητες, όπως εγώ ε, λέω στις προκατακτικές μου παρατηρήσεις, ε, οι ομοιότητες είναι λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν αναγνωρισμένους νομικούς δεσμούς με συγκεκριμένα κράτη, αλλά δεν είναι υπήκοοι. Στα πλαίσια του εγχώριου του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η θέση των κρατών. Το εύρος των δικαιωμάτων τους Μερικές φορές μοιάζει, μερικές φορές διαφέρει. Όσον αφορά το ίδιο το καθεστώς τους, η λεπτονική θέση είναι ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ρητό καθεστώς, ρητά αναγνωρισμένο καθεστώς. Είναι λίγο περίεργη η φράση αυτή. Πρόκειται για άτομα που είναι πρώην υπήκοοι της Σοβιετικής Ένωσης και δεν είναι υπήκοοι καμιάς άλλης χώρας. Για την Εστονία είναι απλά άνθρωποι που δεν έχουν λάβει την υπηκότητα. Υπάρχει λοιπόν κάποια διαφορά όσον αφορά το καθεστώς, έτσι όπως περιγράφεται. Επίσης έχουμε τα δικαιώματα ψήφου στις δημοτικές εκλογές για τους αλλά όχι μη πολίτες, αλλά όχι για τους Λετωνούς μη πολίτες. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, ως μικρή διαφορά, συζητείται στη Λετωνία τα τελευταία χρόνια, ότι η πολιτονικό δίκαιο υπάρχει ένας κανόνας προαιρετικής επιλογής πολιτογράφησης των νεογέννητων. Με άλλα λόγια τα παιδιά μη πολιτών ε, μπορούν να πολιτογραφηθούν εφόσον οι γονείς το αποφασίσουν. Και υπάρχει και ένας κανόνας opt-out. Υπάρχουν λοιπόν ε, στην Εστονία, υπάρχουν λοιπόν κάποιες ομοιότητες και κάποιες διαφορές. Πώς φτάσαμε εδώ. Έχουμε το υποβαθρό του διεθνούς ε, δικαίου, του δημόσιου διεθνούς δικαίου. Έχουμε τη θέση από το δεκαετία του 30 και μετά ότι ο παράνομος έλεγχος επικράτειας δεν δημιουργεί δικαιώματα ε, που να προστατεύονται υπό το διεθνές δίκαιο. Ορισμένα από αυτά είναι σημαντικά, ορισμένα λιγότερο. Αλλά δικαιώματα υπέρπτυσης, αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων, χορήγησης ε, αδειών ε, ε, για διάφορα θέματα. Όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζουμε, ε, που αναγνωρίζουμε στα παραδείγματα που ανέφερα στη Βόρεια Κύπρο, στην Κρυμαία, στη Δυτική Σαχάρα. Εκεί παντού λοιπόν το ερώτημα κλειδί είναι θα είμαστε της άποψης ότι οι χώρες της Βαλτικής βρίσκονταν υπό νόμιμο έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης και συνεπώς οι νέες χώρες που δημιουργήθηκαν το 1991 ήταν τελείως νέες και συνεπώς είχαν την υποχρέωση να χορηγήσουν πολυ... Ε, ηθαγένεια σε όσους βρίσκονταν στην επικράτεια ή μήπως ε, ο έλεγχος αυτός της Σοβιετικής Ένωσης ήταν παράνομος οπότε εκεί βρισκόμαστε στο παράνομη κατάληψη μιας χώρας οπότε τέτοια υποχρέωση δεν υπάρχει. Για να το πω δηλαδή πιο συνοπτικά η mainstream άποψη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται ότι ο έλεγχος της Σοβιετικής Ένωσης δεν ήταν νόμιμος. Οπότε βρισκόμαστε στη δεύτερη περίπτωση, όπου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, παρότι μπορεί να υπάρχει ένα δικαίωμα, όπως βλέπουμε στο λιθανικό παράδειγμα, να χορηγηθεί τέτοιου είδους ε, ηθαγένεια. Ποιο είναι η κατάσταση λοιπόν που έχουμε στα κράτη της Βαλτικής ε, πώς ε, κάλυψαν το χάσμα οι χώρες όπως η Εσθονία και η Λετωνία και όπως είπα υπάρχουν τρεις πιθανές ερμηνείες και δύο λογικές. Οι τρεις πιθανές ε, ερμηνείες, ειδικότερα να δούμε τη λετωνική προοπτική, είναι ότι πρόκειται για, μια ειδική, για ένα ειδικό καθεστώς. Για τους νομικούς αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα ειδικό καθεστώς, ε, ιδιαίτερο καθεστώς, ε, που ισχύει για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση όπου το παρανόμος έλεγχων ε, κράτος δεν χορήγησε υπηκότητα στο επικράτεια που ελέγχε στους απίκους, μετά αποσύρθηκε από εκεί και το νέο κράτος συμπληρώνει το κενό. Ο άλλος τρόπος που θα μπορούσαμε να το δούμε είναι λίγο πιο τυπικό. Θα λέγαμε ότι μπορεί κανείς να έχει μετρημένους αριθμούς, ε, μετρημένα καθεστώτα, κάποια συγκεκριμένα καθεστώτα υπό το διεθνές ε, δημοσιοδίκαιο. οπότε κατ' εξαίρεση, ε, από απαγωγή καταλήγουμε στο ότι πρόκειται για απάτριδες και η τρίτη ερμηνεία είναι ότι είναι υπήκοοι με περιορισμένα πολιτικά δικαιώματα. Ποιο είναι το πιο λογικό. Νομίζω ότι η τρίτη εκδοχή Ο φίλοι μου Αλεξέ Δημητρόφ και Δημήτρη Κότσενοφ θεωρούν ότι η τρίτη λύση είναι η λιγότερο πιστική ως ακαδημαϊκοί ε, το θεωρούν αυτό διότι αντίκειται στις περισσότερες θεσμικές και κρατικές πρακτικές. Κανένα κρατός μόλις δεν αναγνωρίζει κάποιο τέτοιο καθεστώς και όσοι επικρίνουν τα κράτη της Βαλτικής θα επικρίνουν από την άποψη ότι εκεί υπάρχουν απάκριβες. Οπότε το ερώτημα είναι κατά πόσο πρόκειται για ένα ειδικό καθεστώς ευρέως αποδεκτό, κάτι το οποίο το διεθνές δίκαιο μπορεί να αναγνωρίσει, δεν υπάρχει ένα παγιωμένο σύστημα, αν τα πράγματα αλλάξουν μπορεί να γίνει δεκτό. Και εδώ μιλάμε για απάτριδες ουσιαστικά. Και έχω παραδείγματα στον εγγραφό μου που κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Έχουμε ε, τις του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την πλευρά σου Generis ε, στη Λετωνία. Νομίζω ότι στις υποθέσεις Λεβέκο και Ανδρέα έγινε δεκτή αυτή η θέση ως αυτονόητη και οι πρακτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης συνάδουν με αυτό, οπότε αν ενδιαφέρεται κανείς σε διεθνή οικονομικά θέματα θα παρατηρήσει ότι στην πρόσφατη συμφωνία επενδύσεων μεταξύ Σιγκαπούρης και Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επενδυτές αναγνωρίζονται ως ε, υπήκοοι συγκεκριμένων κρατών μελών ε, και όχι ως οι ε, πολιτές της Λετωνίας. Οπότε υπάρχει κάποια αναγνώριση. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνάδει απόλυτα με αυτό. Είπατε εκπρόσωπος για τους πρόσφυγες. Είπατε αρμοστία για τους πρόσφυγες. Συγγνώμη, στα Ηνωμένα Έθνη έχει συμπεριλάβει τους πρόσφυγες στην κατηγορία των απάτριδων. Αλλά δούμε τι γίνεται πρακτικά στι διάφορε επιτροπέ. Διάφορε απόψει έχουν επικρατήσει στα Ηνωμένα Έθνη. Κατά την άποψή μου, τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των απάτριδων, αλλά όχι με απόλυτη συνοχή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παγιώσουμε άποψη για το κατά πόσο η θέση αυτή έχει γίνει αποδεκτή ή όχι, διότι όπως και να το διαβάσουμε, Εάν δεχθούμε ότι ήταν παράνομη η κατοχή της Λετωνίας, σημαίνει ότι δεν ήταν το κράτη της Βαλτικής αυτά που αρνήθηκαν το δικαίωμα υπηκότητας και ψήφου. Όπως και αν το δούμε λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθουμε στο συμπέρασμα ότι δεν τίθεται τεχνικό ζήτημα στέρησης εκλογικών δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο και στις ευρωεκλογέ. Τι μας λέει αυτό ως συμπέρασμα για την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για τη δική σας ε, ε οπτική γωνία όσον αφορά το δικό σας δίκαιο. Και όπως είπα, οι ακαδημικοί συχνά ενθουσιάζονται να κατηγορούν τα θεσμικά όργανα για το ότι κάνουν λάθος. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο. Δεν μιλάμε για καμία παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης. Έχουμε απλή εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η νομολογία του μας οδηγεί προς άλλη κατεύθυνση. Η υπόθεση Αντρέιεβα εναντί Λετωνίας αφορούσε δικαιώματα ιδιοκτησίας όπου στο συμπέρασμα αναφέρεται ρητά ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με διεθνή χαρακτήρα, δεν έχει να κάνει καθόλου με διεθνή χαρακτήρα. Ωστόσο, και εδώ έρχομαι στην περίπτωση της ψηφοφορίας στο Γιβραλτάρ ε, μεταξύ Ισπανίας και Ενωμένου Βασιλείου. Ε, η Επιτροπή δεν έχει αποκλείσει ούτε εκεί, οτιδήποτε. Θα θυμάστε, η Ισπανία ισχυριστήκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίασε την ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας ε, δικαιώματα ψήφου στους κατοίκους του Γιβραλτάρ και το δικαστήριο το απέρριψε. ήταν κάτι που μπορούσε να επιχειρηθεί από πολιτική άποψη. Μερικέ φορέ οι νομικοί λένε ότι αυτό είναι θέμα πολιτική και όχι νομικό. Τι εννοούν, ότι είναι πιο εύκολο, και, αλλά δεν προσπαθώ εγώ να πω αυτό. Η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο μα δίνουν ένα εξαιρετικό παράδειγμα τη πολυπλοκότητα και, και των πολιτικών ευαισθησιών που παρουσιάζονται σε τέτοιε περιπτώσει. Να υπενθυμίσω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έδρασε ω απάντηση σε μια πολύ ε, σημαντική απόφαση του δικαστηρίου στο Great Matthews και United Kingdom σε αυτή την υπόθεση. Ήταν ε, κάποιες επιλογές που ελήφθησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο πολιτικής ευαισθησίας. Σήμερα η νομική τάξη στην Ευρώπη θεωρεί ότι αυτές οι επιλογές πολιτικής ε, ανήκουν στο επίπεδο των κρατών μελών. Εγώ και το έχω συμπεριλάβει σε υποσημείωση στην εκθεσή μου. Θεωρώ ότι εκεί ανήκει η πολιτική συζήτηση, εκεί λαμβάνει χώρα. Στη Λετωνία είδαμε πέρυσι ότι ξεκίνησε ο πρόεδρος μας μια αλλαγή στην πολιτογράφηση των παιδιών. Από τον κανόνα opt-in περάσαμε στον κανόνα opt-out. Ο Παργά και εγώ μια γνωμοδότηση για το θέμα των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έγινε απολύτως δεκτό, αλλά αποτελεί κομμάτι της πολιτικής συζήτησης. Θεσμικά εκεί ανήκει, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Είναι διαθέσιμο το έγγραφό σας, αν κάποιος θέλει να το μελετήσει. Καλό θα είναι να ακούσουμε προσεκτικά αυτά τα οποία μας είπε ο κ. Παπαρίνσκης. Θα ήθελα τώρα να σταθώ στην κυρία Ντεγκρεγόριο. Η κυρία Ντεγκρεγόριο είναι καθηγήτρια συγκριτικού διεθνού δικαίου και ιστορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Θα ακούσουμε με ενδιαφέρον την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ. Με χαρά παίρνω το λόγο ανάμεσά σας και θα ομιλήσω την Ιταλική. Στην τελική αυτή παρουσίαση θα ήθελα να παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία, θα έλεγα, πλαισίωσης ε, του θέματος, για να το καταλάβουμε καλύτερα. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ε, πολλά στοιχεία τα οποία έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Από τη μία υπάρχουν κάποιες ιστορικές και ιστορικογεωγραφικές εικόνες. Υπάρχουν επίσης κάποιες πλευρές διεθνούς δικαίου που έχουν σχέση με την έννοια της διαδοχής των κρατών, όπως επίσης και της δημοκρατικής αιρεσιμότητας και του ανήκειν σε διεθνείς οργανισμούς. Υπάρχουν επίσης και συνταγματικά θέματα η ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ τους αντιφατικών αξιών, αλλά πρέπει να γίνουν όλες σεβαστές προστασία των δικαιωμάτων από τη μία προστασία της κυριαρχίας και της εθνικής ταυτότητας από την άλλη. Υπάρχουν επίσης πολιτικά και γεωπολιτικά θέματα και υπάρχουν επίσης και θέματα ευρωπαϊκού δικαίου όπως και της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Για όλους αυτούς τους ιστορικούς και γεωπολιτικούς λόγους λοιπόν η προστασία των εθνοτικογλωσσικών μειονοτήτων ξεκινά από την εποχή της αποχώρησης της Σοβιετικής Ένωσης και εντάσσεται στις συνταγματικές ρυθμίσεις που συνέβησαν σε όλες αυτές τις βαλτικές δημοκρατίες υπήρξε μια καθυστέρηση στην κεντροανατολική Ευρώπη στην δημιουργία του κρατική της κρατικής δομής. Οι διαδικασίες ξεκινάνε πιο αργά από τη Δυτική Ευρώπη μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκινούν να δημιουργούνται κράτη ε, τα οποία δεν συμπίπτουν με τα έθνη που τα κατοικούν λόγω ακριβώς της αφαίρετης χάραξης των σύνορων μετά από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν δεν γνωρίζουμε το πλαίσιο αυτό δεν κατανοούμε και το τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως υπενθύμησαν οι συνάδελφοι, μιλάμε για χώρες οι οποίες αντίθετα με τις άλλες δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης είχαν μια τυπική ε, είχαν κρατική οντότητα το 1918 και επίσης ε, στις αρχές του 1940. Και γι' αυτό λοιπόν κατά την κομμουνιστική περίοδο η προβληματική της ε, δημιουργίας και της γένεσης του έθνους και του κράτους είναι κάτι το οποίο κατεστάλλει βιαίως και ήρθε στην επιφάνεια πάλι βιαίως μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Πρόκειται για τις μοναδικές δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης που εκτός από την προηγούμενη ιδιότητα κράτους την οποία είχαν το 20 και το 40 είχαν κάποιες παραδόσεις κοινοβουλευτικού τύπου και δημοκρατικού τύπου. Ιδιαίτερα στη δεκαετία του 20 οι χώρες αυτές ήσαν δημοκρατικά στο ίδιο επίπεδο αν όχι ανώτερα από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η περίοδοι αυτοί, οι παραδόσεις αυτές στην ουσία ήταν ε, βασικό χαρακτηριστικό του αγώνα τους για την απελευθέρωσή τους από την Σοβιετική Ένωση και ήταν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της πολιτικής προστασίας του έθνους και της γλώσσας τους. Και οι τρεις βαλτικές χώρες υπάρχουν ρουσόφωνες μειονότητες και όχι απλά ρωσικές, υπήρχαν και πριν από το 1918, ιδιαίτερα στη Λετωνία, υπήρχαν ρωσόφωνες ε, ε, με ρίζες παλαιές κοινότητες. Και από το 1990 και 1991 και μετά, στην ουσία έπρεπε να τους επιστραφεί η ιδιότητα από πολίτη την οποία είχαν, ήταν στην ουσία αυτόχθονες οι ρωσόφωνες αυτοί. Κατά τη διάρκεια όμως της ε, παρουσίας της Σοβιετικής Ένωσης όπως γνωρίζουμε, ε, η ηγεσία στη Σοβιετική Ένωση ε, εφάρμοζε μέτρα μετακίνησης πληθυσμών και μετεγκαταστάσεων σε όλες τις ρωσικές δημοκρατίες και αναμείγνυε συνεχώς τον πληθυσμό. Είχε δηλαδή μια πολύ συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική και οι Ρούσοι και οι Ρουσόφωνοι αποτελούσαν την ελίτ και των τριών ε, δημοκρατιών. Μετά την πτώση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης, αυτή η πολιτική των εθνοτήτων μας δείχνει 25 εκατομμύρια Ρώσων να βρίσκονται στις ε, τέως Σοβιετικές Δημοκρατίες. Σε ορισμένες από αυτές όπως τη Λετωνία, δημογραφικά τη στιγμή της απομάρσαφρωσης της ε, της Σοβιετικής Ένωσης ε, τα ποσοστά έφταναν το 50% του πληθυσμού. Το 52% του πληθυσμού της Εσθονίας ήταν Εσθονή το 1991. Τώρα πώς συμπεριφέρθησαν οι διάφορες δημοκρατίες απέναντι στους Ρωσόφινους, τους 25 εκατομμύρια αυτούς Ρώσους. Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν ήταν διαφορετικός. Στις περισσότερες περιπτώσεις τους δόθηκε η δυνατότητα μηδενικής εκκίνησης, δηλαδή δόθηκε η ιδιότητα του πολίτη στους μόνιμους κατοίκους της χώρας τη στιγμή που απέκτησε την ανεξαρτησία της. Αυτό έκανε η Λιθουανία, διαφορετικό από την Λετωνία. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι η σχέση ανάμεσα στους ρωσόφωνους και στους τοπικούς πληθυσμούς στις υπόλοιπες δημοκρατίες δεν ήταν τόσο ε, σε τέτοια δύσκολη κατάσταση και έτσι ε, τα ποσοστά τους ήταν χαμηλότερα. Στη Λιθουανία η Ρώσοι είναι 10% ας πούμε. Όπως υπενθύμησαν οι συνάδελφοι, οι τρεις βαλτικές χώρες ήταν οι πρώτες οι οποίες πήραν μέτρα αποστασιοποίησης από την Σοβιετική Ένωση και θεώρησαν ότι η ένταξή τους στη Σοβιετική Ένωση του 1940 ήταν υποχρεωτική και βίαιη. Και έτσι λοιπόν το 1991 δεν μίλησαν για αναξαρτησία, αλλά για επαναφορά στην κρατική του οντότητα του 1940. Στην ουσία δηλαδή ε, σβήσαν την ε, σοβιετική κατοχή. Αυτό εν πολλής τεκμηριώνει την λογική της συνέχειας του κράτους και της συνέχειας του κράτους δικαίου και της εφαρμογής ορισμένων μέτρων υπέρ των πολιτών που είχαν χρησιμοποιηθεί στις δεκαετίες του 20 και του 40. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε λοιπόν την ομοθεσία για την πολιτογράφηση των δυτικών χωρών με την Εσθονία και τη Λετωνία γιατί ενώ σε άλλες χώρες η νομοθεσία για την πολιτογράφηση αναφέρεται στην μελλοντική κατά κάποιο τρόπο μετανάστευση, προβλεπτικά δηλαδή, στην Εστονία και τη Λιθουανία μιλάμε για νομοθετικές ρυθμίσεις αναδρομικού αυστηρά χαρακτήρα. Δηλαδή μιλάμε για το στάσος των ανθρώπων οι οποίοι μόλις απέκτησαν την ιδιότητά τους ήταν ήδη τη στιγμή που επέξαν την ιδιότητα του πολίτη ήταν ήδη μόνιμη κάτοικοι. Εδώ τίθεται και το θέμα του σεβασμού των διεθνών υποχρεώσεων των χωρών. Από τη μία έχουμε την έξοδο από την Σοβιετική κατοχή και έχουμε και 50 χρόνια στα οποία ο πληθυσμός αυτός με την εγκατάστασή του απέκτησε δεσμούς με το έδαφος και την συγκεκριμένη περιοχή και δημοκρατία. Τα μέτρα λοιπόν αποκλεισμού, τα μέτρα διακρίσεων που ακολούθησαν την γέννηση εκ νέου των κρατών αυτών δεν είχε σαν στόχο μόνο τις κυρώσεις και τα μέτρα εις βάρος των ρωσόφωνων αλλά είχε σαν στόχο την διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας. Πρόκειται για μία θα έλεγα προσπάθεια οικοδόμησης εκ νέου του κράτους τους. Σαν άμεσο αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών δημιουργήθηκε στις δύο αυτές δημοκρατίες ένα υψηλό ποσοστό τέως Σοβιετικών πολιτών που παρέμειναν απλά μόνιμοι κάτοικοι. Με την πίεση των διεθνών οργανισμών ελήφθησαν ορισμένα μέτρα υπέρ του πλαθισμού αυτού, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει θα έλεγα ένα πυρήνας ανθρώπων που δεν έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στις διαδικασίες πολιτογράφησης ή δεν θέλουν να το κάνουν. Επαναλαμβάνοντας κάτι εδώ θα πω ότι στην περίπτωση της Λετωνίας χρησιμοποιείται ο όρος μη πολίτης ενώ στην Εσθονία ε, αναφέρεται ο όρος πολίτης ακαθόριστης ηθαγένειας. Μιλάμε για δύο διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού και για δύο διαφορετικούς τρόπους πολιτογράφησης. Στη Λετωνία υπάρχει ένας νόμος το 1995 με τροπολογήσεις εκ των υστέρων. Ενώ στην Εσθονία για να υπάρξει ε, καθορισμός του νομικού καθεστώτος των ανθρώπων αυτών ε, πρέπει να προσφύγουμε στον νόμο για τους αλλοδαπούς του 1993. Τώρα η κατάσταση στις δύο αυτές χώρες πως έχει σήμερα. Αν δούμε τους συνταγματικού χάρτες των χωρών αυτών και την προστασία των μειονοτήτων, βλέπουμε ότι οι δύο χώρες αυτές είναι συμβατές με τις γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως επίσης και με τα διεθνή πρότυπα γενικά. Και τα δύο συντάγματα και το λεκτονικό του 22 στο οποίο υπήρξε μια προσθήκη δικαιωμάτων το 98 και το εσθονικό δίδουν δικαιώματα στις ε, μειονότητες χωρίς να τους αποδίδουν την ε, ιδιότητα του πολίτη. Στην Εσθονία δίδονται όχι μόνο με μονομένα ατομικά δικαιώματα αλλά και συλλογικά δικαιώματα που σε επίπεδο συγκριτικού δικαίου διεθνούς είναι θα έλεγα κάτι το ιδιαίτερα ευνοϊκό απέναντι στις μειονότητες. Πέραν όμως αυτού του συνταγματικού απλά πλαισίου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και κάποιες αρνητικές πλευρές. Σχετικά με την Εστονία βλέπουμε ότι το δικαίωμα της χρήσης της ρωσικής γλώσσας στις τοπικές περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι ε, μειονότητες τους δίδονται μόνο όταν ξεπεράσουν το 50%. Στην ανάλυση την οποία έχει κάνει το ειδικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρείται το 50% υπερβολικά απαιτητικό και υψηλό. Σχετικά με τη Λετωνία θυμίζω ότι τον Ιούνιο του 2014 η υιοθέτηση του νέου προημίου του συντάγματος υπογραμμίζει ε, την ε, έννοια του λετονικού έθνους και της λετονικής γλώσσας. Τώρα, εμείς σήμερα μιλάμε κυρίως για την πολιτογράφηση αυτών των μειονοτήτων, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και γενικότερα την νόμοι ισχύουν σχετικά με την εκπαίδευση, τη διδασκαλία της γλώσσας και εκεί υπάρχουν κάποιες απαιτήσει ιδιαίτερα υψηλέ από τους ρωσόφωνους πολίτες και έχουν δημιουργήσει επίσης, οδηγήσει και σε υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό το οποίο παρατηρώ εγώ συγκρίνοντας τις χώρες αυτές και εξετάζοντας τις νομοθετικές σχετικές ρυθμίσεις, αυτό το οποίο έρχεται στην επικαιρότητα είναι η ύπαρξη κάποιων διαφορετικών καθεστώτων ιδιότητας πολίτη και ηθαγένειας που περιπλέκουν τις διαφορές ανάμεσα στους πολίτες και αποδίδουν στους πολίτες εντελώς διαφορετικά καθεστώτα. Υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 τέτοια καθεστώτα. Στις χώρες αυτές έχουμε από τη μία τους πολίτες της χώρας αυτούς, τους αλλοδαπούς, τους ε, κοινοτικούς αλλοδαπούς ή μη κοινοτικούς, τους μη πολίτες και τους μόνιμους πολίτες, ε, μόνιμους κατοίκους μη πολίτες. Χάρη ακριβώς και στον λετονικό νόμο του 95 και η διεθνής κοινότητα σταδιακά αναγνώρισε αυτό το ενδιάμεσο καθεστώς ανάμεσα στους πολλατογραφημένους και τους μη πολίτες, τους απάτηρες ουσιαστικά. Και εκεί βέβαια υπάρχει στέρηση ορισμένων δικαιωμάτων, κυρίως των πολιτικών. Νομίζω ότι η φάση αυτή είναι μεταβατική, αλλά με τα χρόνια να περνούν φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο μεταβατική. Δεν θα επανέλθω τώρα στα θέματα των διαφορών της νομοθεσίας ανάμεσα στις χώρες. Να πω ότι με την πίεση των διεθνών οργανώσεων, του Συμβουλίου της Ευρώπης κυρίως, η νομοθεσία για την ιδιότητα του πολίτη και οι απαιτήσει για την πολιτογράφηση σταδιακά έχουν καταστεί ευκολότερες. Αν και υπογραμμίζω ότι η τελευταία τροποποίηση του λετονικού νόμου του 2013 από τη μία ευνοεί την πολιτογράφηση των ανηλίκων, από την άλλη την περιπλέκει κιολα λόγω ακριβώς των διαδικασιών κυδαιμονίας από τους ενηλίκους και από την άλλη δημιουργεί την δυνατότητα μιας διπλής ηθαγένειας και για τους λετονούς της ιστορικής διασποράς αλλά και για τους λετονούς πρόσφατης μετανάστευσης σε άλλες κοινοτικές χώρες ανάμεσα στις άλλες χώρες όπου έχουν μεταναστεύσει και των οποίων γίνεται δεκτή η διπλή υπηκότητα δεν υπάρχουν σοβιετές σοβιετικές δημοκρατίες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση οι πολλοί από τους μη πολίτες έχουν μεταναστεύσει. Το αίτημα του είπα του εκπροσώπου της ΟΑΣΕ είναι να δώσουμε με αυτόματο τρόπο στους ανήλικους την πολιτογράφηση. Και αυτό έγινε στην Εστονία με την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου που από το 2016, την 1η Ιανουαρίου, αποδίδει αυτόματα στους ανηλίκους ανάμεσα στα 15 με 18 την ιδιότητα του αισθανού πολίτη χωρίς να υπάρξει αίτημα από πλευράς των γονέων τους. Οι βασικές διαφορές λοιπόν ανάμεσα στην Εστονία και τη Λετωνία να δούμε τελικά ποιες είναι. Από τη μία έχουμε την αυτόματη απόδοση της ηθαγένειας στους ανηλίκους και από την άλλη και έχει ενδιαφέρον αυτό από το, από το 1992 και μετά η Εσθονία δίδει δικαίωμα ψήφου ενεργό και στους μη πολίτες δηλαδή τους επιτρέπει να ασκήσουν πλήρως τα πολιτικά τους δικαιώματα αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές και σε σχέση με την συμβατότητα αλλά και τις ρίζες αυτών των μειονοτήτων στην Εστονία και τη Λετωνία. Έχουν <clears throat> τα δικαιώματά τους στην Εστονία περισσότερα από ό,τι στη Λετωνία αλλά υπάρχουν όμως και ομάδες ε, οργανωμένες πολιτών ρωσόφωνων που ισχύουν από την πρώτη στιγμή δημιουργίας του νέου κράτους ερεσιμότητα και συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς. Το ανέφερα ήδη, είναι σαφές ότι το θέμα έχει τεθεί στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο ε, δήλωσε αναρμόδιο γιατί το θέμα της ιδιότητας του πολίτη παραμένει πάντα ένα εσωτερικό θέμα σε αυτές τις χώρες. Αν και το δικαστήριο ασχολήθηκε με διάφορα περιφοριακά θέματα όπως ε, το θέμα της προστασίας της ε, οικογενειακής ε, γαλήνης και ελευθερίας. Το ίδιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη φορά στην απόφαση Μικελέτη και σε διάφορες άλλες διαδοχικές αποφάσεις αναγνωρίζει μεν ότι το θέμα της ιδιότητας του πολίτη είναι ένα θέμα το οποίο χαίνει στις χώρες αυτές σε σχέση με την απόδοσή της, αλλά ζητεί από τις χώρες να σεβαστούν πλήρως τις αξίες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, τα θέματα τα οποία τίθενται είναι περίπλοκα και δύσκολες θα είναι οι λύσεις και εμπλέκουν πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Όπως είπα εγώ σε επίπεδο συνταγματικό, διότι με αυτά ασχολούμαι, πρέπει να εξισορροπηθεί. Από τη μία το συμφέρον προστασίας και κυδαιμονίας και από την άλλη οι προτεραιότητες τις οποίες έχουν οι χώρες αυτές σχετικά με την προστασία της κυριαρχίας τους αλλά και τη συμμετοχή τους και σεβασμό τον οποίο πρέπει να επιδεικνύουν στις διεθνείς συμφωνίες ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς λοιπόν ε, είπαμε ότι τα μέτρα αυτά διακρίσεων σε εισαγωγικά, αποκλεισμού σε εισαγωγικά των μειονοτήτων είχαν ε, λυθεί για να βοηθηθεί η ανοικοδόμηση του κράτους. Αλλά τώρα πια έχουν αρχίσει και αλλάζουν σιγά σιγά. Διευρύνεται η συζήτηση στα ειδική βιβλιογραφία σε επίπεδο διεθνού συνταγματικού και ευρωπαϊκού διεθνούς. Πολύ συχνά ε, λέγεται ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, αγκυρώνοντας την ιδιότητα αυτή με ε, την ε, αντίστοιχη ιδιότητα του κράτους. Μπορούμε να μην μιλάμε δηλαδή μόνο για, να μιλάμε μάλλον μόνο, όχι μόνο για μη Εστονούς και μη Λετονούς πολίτες αλλά και μη Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την ολοκλήρωση της Ευρώπης η οποία δείχνει να αγνοεί μια σημαντική ομάδα πολιτών. Οι πολιτικές λύσεις οι οποίες προτείνονται και οι οποίες είναι αρκετά πρωτότυπες, κυρίως δύο από αυτές, η μία προέρχεται από τους Δημητρόφ και Κοτσενόφ, και αναφέρονται ε, στην ιδιότητα των πολιτών ε, με αναφορά τον κοινοτικό νόμο. Στην ουσία δηλαδή αναφέρονται στο βρετανικό προηγούμενο των overseas citizens. Συνεπώς λοιπόν η πρόταση αυτή από τη μία δημιουργεί κάποια θέματα γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς γιατί κάτι τέτοιο να ισχύσει μόνο για τη Λετωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση και όχι για την Εστονία. Και πώς τα δικαιώματα αυτά θα μπορούσαν να δοθούν στους πολίτες αυτούς γιατί τα δικαιώματα τα οποία έχουν και των οποίων χαίρουν οι πολίτες αυτοί Υπάρχουν και άλλα δικαιώματα όπως η ελεύθερη διακίνηση, το δικαίωμα εγκατάστασης και λοιπά Τους αποδίδονται ήδη εφόσον θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι σε τρίτες χώρες. Υπάρχει και μία άλλη πρόταση ενός Ιταλού όπως του Φόρνη, το οποίο αναφέρονται σε μία ενδιάμεση πρόταση ευρωπαϊκής ιδιότητας πολίτη. Στην κατηγορία αυτή θα δοθούν ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα όπως το δικαίωμα της παθητικής συμμετοχής στις ευρωεκλογές όπως ακούσαμε από κάποιες αναφορές σήμερα, είναι σαφές ότι η ιδιότητα του μη πολίτη ε, δίδει ορισμένα δικαιώματα, αλλά τα πολιτικά δικαιώματα παραδοσιακά είναι τα πιο σημαντικά και η ιδιότητα του πολίτη συνδέεται με την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη. Πάντως, δεν μπορεί κανείς να μην κάνει την αναλογία ανάμεσα στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την ιδιότητα του πολίτη και τα μέτρα εκαθάρισης τα οποία ελήφθησαν στην αρχή της νέας περίοδου ιστορίας των κρατών αυτών απέναντι στους πολίτες του τέος κατακτητή. Πάνω σε αυτά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων εννοώ, έχει εκφραστεί επανειλημμένα και έχουν σχολιαστεί τα μέτρα αυτά. Και είπαμε ότι στην αρχή της ε, οικοδόμησης της κρατικής ήταν ε, νομιμοποιημένα τα κράτη αυτά για να πάρουν κάποια τέτοια μέτρα. Αλλά τώρα πια με τον χρόνο είναι σαφές ότι θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ντιγκρεγόριου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ε, μέρος ε, οι συνάδελφοι σε αυτήν την συζήτηση μετά από τις τρεις εξαιρετικές ε, παρουσιάσεις. Προσπαθήστε αν κάνετε ερωτήσεις να τις απευθύνετε στον συγκεκριμένο άτομο θα δώσω το λόγο πρώτα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να πάρετε το λόγο εάν το επιθυμείτε φυσικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ίσως πιο σκόπιμο θα ήταν να μιλήσω για το επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως, όχι για τους εδώ. Πολύ ωραία. Ε, κυρία Γιάννα τον πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Δεν ήθελα να είμαι πρώτη ε, έτσι ώστε να μπορώ να κριτικάρω άνετα οποιονδήποτε ότι είπε κάτι που ήταν ανόητο. Αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω, δεν πειράζει. Ε, είχα πολλές παρατηρήσεις ακούγοντας ε, και μια και έχουμε μονάχα έξι ε, βουλευτές θα έχω ίσως και αργότερα τη δυνατότητα να ξαναπάρω το λόγο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κανένας δεν αναφέρθηκε σε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ε, πολλούς, ε, για τον μεγάλο αριθμό των Ρώσων πολιτών ε, στην Εστονία και μιλάμε για τον αριθμό των μη πολιτών που διαρκώς μειώνεται, αλλά δεν αναφέρατε γιατί. Πρώτον είναι ο θάνατος, δεύτερον είναι τα ρωσικά διαβατήρια και το τρίτο είναι η πολιτογράφηση αν μιλάμε για όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερο σόφρον να έχουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό Ρώσων πολιτών που ζουν εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Επικρατείας. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως είναι βέβαιο ότι ε, πολύ εύκολα μπορούν ε, οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν ε, ε, να πάρουν την ε, υπηκότητα τη ρωσική αν δεν θέλουν να έχουν αυτά τα λεγόμενα γκρίζα διαβατήρια. Επίσης, πριν γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η Εστονία, είχαμε πολλές συστάσεις από πολλούς διεθνούς οργανισμούς ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Και τώρα έχουμε μία σύσταση κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον. Τι γίνεται με αυτό, γιατί δεν έχουν ε, καλυφθεί τα όσα αναφέρονται στις συστάσεις. Επίσης, κανείς από τους τρεις σας ε, δεν αναφέρθηκε ε, σε μια ομάδα ανθρώπων στην Εστονία, τουλάχιστον δεν ξέρω πώς είναι στη Λετωνία, γιατί η Εστονία έδωσε ηθαγένεια όχι μονάχα σε αυτούς που ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο, αλλά και σε εθνοτικά στο νους, ε, χωρίς, καμία, χωρίς καθόλου εξετάσεις. Δεν μιλούσε στονικά γεννήθηκε η μάνα μου, γεννήθηκε στην ε, Ρωσία. Κανένας ε, δεν της ζήτησε να, να πει που ήταν στη διάρκεια της κατοχής. Και επίσης για την τελευταία ομιλήτρια, δεν είναι αλήθεια ότι οι μη πολίτες μπορούν να ασκήσουν την ελεύθερη, το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας ούτε ως εργαζόμενοι ε, ούτε όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες. Εάν έχω μια μικρή επιχείρηση στην Εστονία, ναι, εγώ μπορώ να την μετακινήσω σε μια άλλη χώρα, αλλά εγώ ως εστονός δεν μπορώ να πάω ε, κάπου αλλού παρά μόνο για 90 μέρες. Δεν έχω ελευθερία κίνησης και μετακίνησης. Ίσως δεν ήταν ακριβώς ερώτηση, έκανα σχόλια τα οποία ίσως μπορείτε να σχολιάσετε. Ναι, και όταν θα ε, μαζευτούν όλες οι ερωτήσεις θα απαντήσετε ε, μία προς μία. Μήτρος Άνιψ, ζητώ συγγνώμη για την προφορά, λέει η προεδρο Μια... Μητροφάνοφ λέγομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Βεβαίως για μας που ερχόμαστε από τις βαλτικές ε, χώρες που εκπροσωπούμε εθνοτικές ε, ε, μειονότητες και ρωσόφωνους όλα αυτά δεν είναι καινούρια. Τα γνωρίζουμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Ελπίζω πάντως ότι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα βρήκαν χρήσιμες αυτές τις νέες για αυτούς ίσως πληροφορίες. Άκουσα μία λέξη στην τελευταία παρουσίαση της κυρίας Δεγκριγόριο. Αν κατάλαβα καλά, είπε ότι πρέπει να δούμε ότι η στάση προς τους non-citizens μάλλον η στάση το, όσον αφορά την πολιτογράφηση είναι λίγο η αίσθηση ότι αποτελεί τιμωρία ε, για ε, τους ρωσόφωνους. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μην κάνουμε τόσο απλουστευτική προσέγγιση. Εδώ δεν μιλάμε μονάχα ε, για την ιδιότητα του πολίτη. Περιπλέκεται το θέμα και με άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τις χώρες της Βαλτικής. Αναφέρομαι ας πούμε στις τελευταίες πρόσφατες εξελίξεις της κρατικής πολιτικής όσον αφορά τα μειονοτικά σχολεία τι, αυτά που συνέβησαν τα τελευταία 27 χρόνια επίσης, γιατί βλέπουμε ότι ναι, αυτά αποτελούσαν κατά κάποιο τρόπο ε, ε, ε, τιμωρία ε, για το, τα όσα συνέβησαν στη διάρκεια του σταλινικού ε, καθεστώτος το, οι διαδικασίες που ξεκίνησαν το 1991, ε, ναι, ε, είναι μια τιμωρητική διαδικασία, καθώς επίσης και μια προσπάθεια εξέβρεσης ε, πόρων. Υπήρξαν δημεύσεις περιουσιών έτσι ώστε να αποκλειστούν οι άνθρωποι αυτοί από τις περιουσίες τους και από, τις, από τη δυνατότητα να ασκήσουν κάποια επαγγέλματα. Ε, και επίσης ε, ε, να μην έχουν δικαιώματα να λάβουν καλή εκπαίδευση στην δική τους γλώσσα έτσι ώστε να μπορέσουν μετά να ακολουθήσουν μια καλή καριέρα στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο. Επίσης δεν άκουσα Ίσως δεν το κατάλαβα, το είπατε, αλλά δεν το κατάλαβα. Ποια μπορεί να είναι ε, τα πολιτικά, ε, ε, ποιες μπορεί να είναι οι πολιτικές ε, και εθνικές αποφάσεις. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να πιέσουν κατά κάποιο τρόπο τις χώρες της Βαλτικής να λύσουν το πρόβλημα αυτό. Γιατί εμείς είμαστε εδώ τρεις εκπρόσωποι μειονοτήτων από τις ε, χώρες της Βαλτικής. Είμαστε εδώ, σας μιλούμε, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν συνάδελφοι. Α, θα έρθουν να ψηφίσουν λέτε. Ναι, αλλά πάντως φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει ε, το, η επίλυση των ζητημάτων αυτών. Ερώτηση παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος. Όχι, ήθελα να κάνω σχόλιο. Το κύριο ερώτημα είναι το εξής. Ποια θα μπορούσε να είναι η λύση αυτού του προβλήματος ε, ε, με νομικούς και πρακτικούς όρους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάνικινς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Τρεις ερωτήσεις, ε, μία για τον καθένα. Πρώτα για την κυρία Τόνισπαν. Ε, υπάρχουν πολίτες που βρίσκονται στην ε, Λετωνία τέσσερα, εδώ και τέσσερις ε, γένες και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές. Το, οι άνθρωποι αυτοί ήταν ε, μερικές χιλιάδες άνθρωποι αλλά οι πολιτογραφήσεις ε, είναι περίπου χίλιες ε, το χρόνο. Ε, βέβαια όταν η Λετωνία ήταν υποψήφια χώρα είχε υποσχεθεί ότι θα λύσει αυτό το θέμα των μη των μη πολιτών. Αλλά 14 χρόνια μετά νομίζω ότι οι αυταπάτες έχουν λήψει. Ερώτηση με ποιο τρόπο βλέπετε ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα ε, των Λετωνών και Εστονών που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Δεύτερη ερώτηση στον κύριο Μάρτης Παπαρίνσκης. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι το 1995 ε, στην ε, Λετωνία θεσπίστηκε ο νόμος για τους πρώην Ρώσους υπηκόους. Η Σοβιετική Ένωση ε, ε, ε, κατέρευσε περίπου 25 χρόνια πριν αλλά υπάρχουν στις χώρες μας παιδιά τα οποία είναι παιδιά πρώην πολιτών της Σοβιετικής Ένωσης και εν τέλει συνεχίζουμε στις χώρες αυτές να παράγουμε κατά κάποιο τρόπο σοβιετικούς πολίτες το 2016 ε, ε, ε, και παραθέτω σε μία έκθεση αναφέρθηκε και παραθέτω ότι είναι πολλά τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί στην Λετωνία από ανθρώπους που έχουν αυτό το καθεστώς μη πολίτη και είναι παιδιά με ρωσική υπηκότητα. Τι μπορεί να γίνει από άποψη νομική αλλά και άποψη πρακτική έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα των νεογέννητων, των νέων ε, Ρώσων πολιτών. Και στην κυρία Άντζελα Δεγκριγκόριο, ε, Εσείς συγκρίνατε λίγο τις ε, καταστάσεις στις τρεις χώρες της Βαλτικής. Ήταν καλή η εικόνα που δώσατε. Ωστόσο, ξέρετε ότι η Λιθουανία είχε επιλέξει το δικό της τρόπο και έδωσε αυτόματα ε, την ιδιότητα του πολίτη σε όλους τους ε, πολίτες της πρώην Λιθουανικής ε, Δημοκρατίας, Σοβιετικής Δημοκρατίας της Λιθουανίας. In And in March of 1990... Όταν τον Μάρτιο του το 1990 ένας φίλος μου, ο οποίος είχε έρθει μόλις μερικούς μήνες πριν στη Λιθουανία, έγινε ε, Λιθουανός υπήκος. Γιατί αυτή η κατάσταση ήταν δυνατή στην Λιθουανία και όχι στη Λετωνία και την Εστονία. Ε, αυτά ήθελα να σας ρωτήσω και σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Δεν βλέπω να ζητά κάποιο το λόγο, αλλά η συνάδελφο θέλει μία επιπλέον ερώτηση. Ναι, μια ερώτηση εξ ονόματο τη αδερφή μου, η οποία δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει γιατί επισήμω είναι μη ε, ε η υπήκο και τώρα ζει ευτυχώς στην Ολλανδία και είναι Ολλανδή Υπήκο. Για τον κύριο Παπαδίνσκη, λέτε στο έγγραφό σα ότι δεν συμφωνείτε ότι οι πολίτες αυτοί ε, ή πρέπει να θεωρούνται ε, ε, ενωσιακοί πολίτες γιατί αυτό δεν είναι δεν συνάδει με τις αρχές του ενωσιακού νόμου. Αυτό όμως τι σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ζητήματα ηθαγένειας θα πρέπει να αγγίζουν τις ενωσιακές αρμοδιότητες. Παρακαλώ κύριε Πάμπριξ. Thank Άκουσα προσεκτικά ε, από την οθόνη ε, τη συζήτηση και τις παρουσιάσεις των τριών εμπειρογνωμών και πρέπει να πω ότι ε, ο επαγγελματισμό τους είναι ύψιστο του επίπεδου. Από αυτή την άποψη λοιπόν να σα κάνω και εγώ κάποια σχόλια Ε, τότε που σπούδαζα και δίδασκα για τις εθνικότητες και για την εθνική πολιτική. Ξέρετε, μπορούμε να συζητήσουμε εκτενώς πολλά ζητήματα για μειωνοτικά δικαιώματα, δικαιώματα πολιτών, διότι καμία χώρα δεν είναι απολύτως τέλεια. Προκλήσεις υπάρχουν πάντοτε. Ειδικότερα τώρα για το ζήτημα των χωρών της Βαλτικής και αυτό το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε σήμερα, ε, θα ήθελα να πω ότι από πολλές απόψεις, κατά την προσωπική μου γνώμη και οι δύο χώρες και οι τρεις χώρες της Βαλτικής έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των μειονοτήτων γενικότερα αν το δούμε από άψη ευρωπαϊκών προτύπων. Οπότε εδώ θα μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται με την παιδεία στις μετρικές τους γλώσσες μέχρι ένα επίπεδο στο σχολείο, τη δυνατότητα να έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στις δικές τους γλώσσες και πολλά άλλα. Ε, έχουν τέτοια δικαιώματα λοιπόν σε αυτέ τι χώρε, κάτι που δεν υπάρχει σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά πάντα τίθεται ένα ζήτημα μειονοτήτων, ε, ε, κατά πόσο αρκούν όλα αυτά που του προσφέρονται ή όχι και να υπενθυμίσω εδώ γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα γενικότερα. Γιατί τέθηκε αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα ότι γενικά η συζήτηση δεν αφορά το πόσα θα είναι τα δικαιώματα που δίνουμε στις μειονότητες και ποιος τα έχει διότι εδώ οι χώρες της Βαλτικής δεν μπορούν να ανταγωνιστούν Γαλλία, Γερμανία και άλλες, άλλες, χώρες, πολλές χώρες. Το ερώτημα εδώ είναι πιο σημαντικό για αυτές τις χώρες της Βαλτικής. Είναι ερώτημα ε, ύπαρξης ουσιαστικά, είναι θέμα ύπαρξης. Και για πολλούς από τους συναδέλφους μου υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ του να θέτουμε το ζήτημα των μη πολιτών, μειονοτήτων, που είναι δύο διαφορετικά θέματα, διότι αυτοί οι εθνοτικοί Ρώσοι, για παράδειγμα, που υπήρξαν πολίτες ε, ε, στη Λετωνία και στην Εστονία και πριν τον πόλεμο, πριν από την κατοχή της Σοβιετικής Ένωσης, αυτοί έλαβαν ε, πολιτογράφηση αυτόματα, χωρίς καμία ερώτηση. Χωρίς να μιλούν λετωνικά, ούτε τίποτα άλλο. Τους δόθηκε απλά η θαγένεια όπως και στους άλλους. Η διαδικασία πολιτογράφησης αφορά μόνο εκείνους που απήκησαν την περιοχή κατά το χρόνο κατοχής ε, όταν δεν υπήρχαν αυτές οι χώρες οπότε ήταν κυρίαρχο δικαίωμα και το ανέφερε και ο κύριος Παπαρίνσκι οπότε μπορούμε να συζητάμε ό,τι θέλουμε για τα εθνικά δικαιώματα είτε τους αρέσει είτε όχι είναι κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών αυτό αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά αν συμφωνήσουμε με εκείνους που στηρίζουν αυτή την αναφορά για να το πω έτσι. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπους, όχι μόνο που ανησυχούν για αυτές τις χώρες. Μιλάμε, να παρέμβουν λίγο. Κάνουμε ερωτήσεις σε σχέση με τις παρουσιάσεις αυτή τη στιγμή. Σε λίγα λεπτά θα έρθουμε στην αναφορά 747. Ε, Οπότε παρακαλώ μην θέσετε το ζήτημα τώρα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πολύ σύντομη. Μπορείτε να μας ξαναπείτε και να μας πείτε ότι συμφωνείτε με το ότι αν συμφωνήσει κανείς με αυτούς τους αναφερόμενους ουσιαστικά συμφωνεί και με το ότι οι χώρες της Βαλτικής δεν είναι κατεχόμενα δάφη τη Σοβιετικής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, πολύ ισχυρή αυτή η δήλωση. Παρακαλώ κύριε ε, Πέιτ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είναι ώρα για ερωτήσεις, θα τις θέσω ως εξής. Μήπως θα μας βοηθούσε να βρούμε μια λύση το να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το παράδειγμα αυτών των 161.000 ανθρώπων στην Εστονία η οποία ε, τα τελευταία 27 χρόνια ε, ε, ακολούθησαν, ε, πέρασαν εξετάσεις, ε, διαγωνίσματα και στα, στην εστονική γλώσσα. 161.000 άνθρωποι οι οποίοι έγιναν ε, στον ή, πολίτε χωρίς κανένα πρόβλημα. Φανταζούμε ότι κάθε ανθρώπινο όν θα πρέπει να έχει την, ε, την ικανότητα να μάθει μία γλώσσα, όποια γλώσσα έκανε αυτή σε περίοδο 27 ετών. Όταν λοιπόν συζητάμε αυτό το ζήτημα σήμερα, θεωρώ ότι το βασικό ερώτημα τελικά είναι ποιο είναι το κίνητρο. Έτσι λοιπόν και ο τίτλος ε, της σημερινής εκδήλωσης, της σημερινής ε, παρουσίασης, ε, το μη ε, πολίτες δεν στέκει, διότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πολίτες εφόσον πληρώνουν τα κριτήρια. Γι' αυτό τον λόγο πιστεύω καλύτερα θα ήταν να πούμε άνθρωποι με ακαθόριστη ηθαγένεια. Οπότε υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πού υπάρχει δυνατότητα να πάρει κανεί την υπηκότητα χωρί να γνωρίζει την εθνική γλώσσα ή την επίσημη γλώσσα. Πόσε περιπτώσει τέτοιε έχουμε. Και ποια είναι η ιδιαίτερη ιστορία τέτοιων χωρών όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μετά, όταν έχουμε μια πλήρη κρατική υποστήριξη σε ένα δίκτυο σχολείων που διδάσκουν σε ανθρώπους την γλώσσα που δεν είναι η επίσημη γλώσσα, έχετε τέτοιο πράγμα στην Γερμανία δημόσια σχολεία που να τα πληρώνει η κυβέρνηση και να διδάσκουν στην τουρκική γλώσσα. Στο Βέλγιο έχετε εδώ ε, σχολεία πολλά αραβικά που να χρηματοδοτούνται από το κράτος. Πώς σχολιάζετε δηλαδή αν κάνουμε τη σύγκριση της σημερινής κατάστασης με αυτή άλλων χωρών στην Ευρώπη. Οπότε ε, θα ήθελα ταπεινά να ζητήσω το εξής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, παρακαλώ, να μην υποβαθμίζουν τα κίνητρα αυτών των ανθρώπων, να τους ενθαρρύνουν αντιθέτως, να λάβουν την ηθαγένεια, να μάθουν την εστονική γλώσσα, τη λετωνική γλώσσα και το πρόβλημα θα έχει τελειώσει. Θα γίνουν πολίτες με όλα τα δικαιώματα, Εστονοί ή Λετωνοί, και θα πάψει να υπάρχει αυτό το ζήτημα και να το αποτελείται αντικείμενο εκμετάλλευση στην καθημερινή πολιτική. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννα. Και εσεί θέλετε να κάνετε μια επιπλέον ερώτηση. Συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν ήταν ερώτηση. Απλά ήθελα να αναφερθώ στο αυτό που είπε ο κύριο Πάπρεξ, που ήρθε να κάτσει εδώ δίπλα μου. Εγώ όταν γεννήθηκα το 1966 στο Ταλίνι, η μητέρα μου ήταν στον ο πατέρα μου ήταν Ρώσος. Και εγώ δεν πήρα τόσο εύκολα υπηκότητα. Χρειάστηκε να περάσω το διαγώνισμα. Ε, ε, και η πολιτική, η, η συγγνώμη, ε, δεν, πρόεδρος, δεν έχουμε άλλο χρόνο για προσωπικές μαρτυρίες. Να δώσω ξανά τον λόγο στους συμπρογνώμονες για να μας σχολιάσουν και να απαντήσουν τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Θα πάμε αντίστροφα. Πάμε σε εσά πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι ε, ειδικό σε νομικά θέματα. Δεν θέλω να εμπλακώ σε πολιτικά θέματα, αν είναι δυνατόν, γιατί δεν έχω προετοιμαστεί για να απαντήσω πολιτικά ερωτήματα. Ήθελα να υπογραμμίσω λοιπόν ένα πράγμα. Οι περισσότερε ε, πρώην δημοκρατίε της Σοβιετική Ένωση υιοθέτησαν την απόφαση να δώσουν υπηκότητα στους ε, πολίτες, στους μόνιμους κατοίκους που είναι μόνιμοι κάτοικοι για κάποια χρόνια, κάποιο συγκεκριμένο αριθμό χρόνων. Γιατί, διότι με εξαίρεση την Εστονία και τη Λετωνία, το ποσοστό ρωσόφωνων, επιμένω, τους ονομάζω ρωσόφωνους, είναι άνθρωποι που έχουν τα ρωσικά ως γλώσσα, δεν ήταν τόσο υψηλό ώστε να αποτελέσει αιτία δημογραφικού προβλήματος. Ε, εδώ στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι πρωταρχικά δημογραφικό πρόβλημα. Όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ξέρω, θυμάμαι ότι για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Ευρώπη επιμελείται το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οπότε ίσως να είναι καλύτερο να γίνει αυτή η συζήτηση σε έναν άλλο χώρο. να στραφούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να βρεθεί μια λύση τουλάχιστον για τα γλωσσικά προβλήματα, τα προβλήματα παιδείας. Τι άλλο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αλληλογία των κρατών στο διεθνές δίκαιο. Είναι παραδεκτό ότι οι επόμενες χώρες δίνουν, δίνουν ε, σε μια τέτοια περίπτωση ε, την υπηκότητα τα διάδοχα κράτη, αλλά σε αυτή τη στιγμή μιλάμε για συνέξι κρατών που γεννήθηκαν ήδη από το 1980. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν απάντησα σε ερωτήσεις. Thank Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις νομίζω απευθυνθήκαν σε μένα, οπότε θα τις απαντήσω. Η πρώτη ήταν κάπως ευρύτερη, οι άλλες δύο πιο εστιασμένες. Η πρώτη από τον κύριο Μητροφάνοφ ε, ρώτησε κάπως έτσι γενικόλογα τι μπορεί να γίνει για αυτόν τον πληθυσμό των μη υπηκόων. Κατά την προετοιμασία αυτής της έκθεσης ε, αντιληφθήκα ότι η διεθνής κοινότητα γενικά στρέφει την προσοχή της μακριά από το καθεστώς και προς συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αν δούμε λοιπόν πώς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΠΑ ασχολήθηκε με το ζήτημα, πώς το σχολίασαν τα κράτη, όσοι επέκριναν το καθεστώς και όσοι δεν το επέκριναν, αν δούμε λοιπόν, πιστεύω, ότι την οριζόντια συνένεση περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σε εντυπωσιακό βαθμό υπάρχει συμφωνία. Και αυτό μου φαίνεται ότι είναι ο πιο παραγωγικός τρόπος ε, ε, εξέταση του ζητήματο. Ο κ. Μαμικίνης ανέφερε το δικαίωμα για τα παιδιά, αλλά πιστεύω ότι σε όλα τα επίπεδα αυτό είναι το καλύτερο που μαθαίνουμε από την περίπτωση Ανδρέα ότι έχουμε πολλά ανθρώπινα δικαιώματα που ίσως ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα από τη θέση που λαμβάνει κανείς για το καθεστώς. Ε, για τις εθνικές μειονότητες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το δικό μας συνταγματικό δικαστήριο έχει λάβει διάφορες αποφάσεις που έχουν αποτελέσει νομολογία τα τελευταία χρόνια. Έτσι ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε περίπλοκα συνταγματικά ερωτήματα. Είμαστε κράτος δικαίου και αυτό θεωρώ ότι και εγώ είναι σωστό, να εξετάσουμε τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει και όχι το καθεστώ. Ο κ. Μαμίγκη με έκανε μια ερώτηση για την κατάσταση των παιδιών που γεννιούνται ως μη πολίτες. Και πολύ σωστά ανέφερε δύο συστάσει τη επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού. Ναι, αυτό συζητείται αυτή τη στιγμή πολιτικά, το γνωρίζετε. Ο πρόεδρος μας έκανε μια παρόμοια δήλωση το Σεπτέμβριο. Δεν εστέφθη με επιτυχία μέχρι στιγμής. Ίσως εγώ επειδή είμαι ακαδημαϊκός στον Ρωμανό Βασίλειο το βλέπω έτσι ε, με την αντιμετώπιση ρεαλιστικά ενός ζητήματος ε, μετά το άλλο σταδιακά έτσι θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση. Μετά η κυρία μου έκανε μια ερώτηση ε, Η απάντηση βρίσκεται, κάποια έδειξη βρίσκεται στην υποσημείωση 17. Ρώτησε αν η κατάσταση έχει αλλάξει μετά το 2015. Δεν νομίζω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εγώ πιστεύω ότι η αφετηρία εξακολουθούν να είναι τα άρθρα 9 και 10 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βαθμό που δεν έχουν αλλάξει κιόλας. Οπότε όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Η, η ευρωπαϊκή υπηκότητα, η υπηκότητα ενός κράτους μέλους και τα ευρωπαϊκά εκλογικά δικαιώματα είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν νομίζω ότι η κατάσταση μετά το 2015 άλλαξε. Ε, αλλά και πάλι να συγχαρώ τη βοηθό σα. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία ακούστηκαν. Είπατε ότι δεν ε, αναφέρθηκαν, δεν αναφέρθηκα σε κάποια θέματα, μα είναι πολλά αυτά τα οποία δεν είχα χρόνο να αναφέρω. Θα δω κάτι που μου φαίνεται πιο σοβαρό και κάτι πιο μικρή σημασία ο λόγος για, τον, ε, για την εξέλιξη <clears throat> της διαδικασίας ε, πολιτογράφησης. Ναι, έχετε δίκιο ότι αφενός υπάρχουν οι θάνατοι και φετέρου υπάρχει και η αποδοχή άλλων, ε, άλλων ηθαγενειών. και σιγά σιγά είναι όλο και περισσότεροι ε, οι πολίτες που έχουν την ιδιότητα του πολίτη. Στην συνολική συζήτηση θεωρώ πολύ ενδιαφέρον που συζητιέται το ζήτημα αυτό ως καθαρά νομικό ζήτημα και στο με τη συνάδελφο που ασχολείται, βλέπει το θέμα από αυτή την πλευρά το ζήτημα είναι όμως πώς μπορεί να προκύψει η κοινωνική αλλαγή, πώς είναι δυνατόν τα κοινωνικά ζητήματα, η καρδιά των ανθρώπων αν θέλετε ε, να αλλάξει. πώς μπορεί κανείς ε, να συμμετάσχει σε αυτήν την ε, ε, εμπειρία της κοινωνίας. Ε, και νομίζω ότι ε, μερικές φορές συνήθω έχουμε την κοινωνική αλλαγή η οποία φέρνει μαζί της την νομική αλλαγή. Άλλες φορές όμως ε, η κοινωνική αλλαγή προκύπτει μετά από την νομική αλλαγή. Να μην ξεχνάμε ότι η εστίαση είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια κοινωνική συζήτηση εντός των κοινωνιών. Δηλαδή πού βρισκόμαστε ω κοινωνίε, πώ αποδεχόμαστε, πώ βλέπουμε την ιστορία μας πώς ε, ζούμε και πώς ε, αντιδρούμε απέναντι στην πραγματική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και στην οποία ζούμε. Ποια θα μπορούσε να είναι ε, η λύση για την κοινωνία. Τα προβλήματά μας θα λυθούν εάν όλοι γίνουμε πολίτες. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Κάποια ζητήματα ναι. Ίσως θα υπήρχαν λιγότερα προβλήματα αλλά δεν μπορεί να ε, ξεφορτωθούμε τα προβλήματά μας μόνο μέσω ε, της, ε, της ιδιότητας του πολίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Σας ευχαριστούμε που παρουσιάσατε τα θέματά σας και βεβαίως εάν θέλετε σας παρακαλώ να παραμείνετε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επόμενης αναφοράς. Εάν θέλετε να φύγετε πάλι παρακαλώ ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως όπως και να έχει το θέμα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, συμβολή σας, ε, την πολύτιμη σε αυτό το πολύ δύσκολο ζήτημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω ότι ξαφνικά έρχονται και περισσότεροι συνάδελφοι και πρέπει οπωσδήποτε τώρα να ξεκινήσουμε τη μελέτη του θέματος 23 αναφορά υπαριθμών 747 του 2016 του Στεργέη Στεπανόφ, κατοίκου Εστονίας, που συνοδεύεται από 19.552 υπογραφές σχετικά με τα εκλογικά και πολιτικά δικαιώματα των κατοίκων Εστονίας και Λετωνίας που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, είναι παρόν ο ίδιος ο αναφέρον, αλλά ο κύριος Χάουρ Κέντερ τον εκπροσωπεί. Και χαίρομαι που μπορώ να σας δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αισθάνομαι λίγο απελπισμένος εδώ. Είμαι βέβαια ευγνώμων που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, αλλά το πρόβλημα των απάτριδων βλέπω ότι δυσκολεύει όλο και περισσότερο Ε, βρίσκεσαι έτσι, δεν, ε, δεν έχεις δικαιώματα ε, και αν δείτε ας πούμε στις εστονικές φυλακές βρίθουν κρατουμένων ρωσικής ρωσοφόνων γιατί πραγματικά γίνεσαι βόρα εγκληματικών οργανώσεων. Επίσης βλέπουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή η οποία ένα δράμα το οποίο συνεχίζεται. για αυτούς που πιστεύουν ότι οι ε, ε, η εθνοτική καθαρότητα ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ έχουν πεδίο δόξης λαμπρών, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και αυτά που ακούσαμε εδώ, ναι, ίσως είναι ενδιαφέροντα αλλά πραγματικά με απελπίζουν γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση γιατί δεν αγγίζουμε την καρδιά τον πυρήνα του προβλήματος. Οι εθνικιστές ε, θέλουν ε, να συγκρίνουν ε, τους εαυτούς τους με άλλες χώρες αλλά δεν την συγκρίνουν την Εστονία με τη Φιλανδία ας πούμε που είναι μια μικρή χώρα αλλά που Ε, και ε, που ε, λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και που κανείς δεν αισθάνεται να απειλείται, που έχει ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα, που οι φυλακές και το, το, το, το σύστημα το δικαστικό αντιμετωπίζει όλους με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε, εδώ δεν έχουμε τον πολιτικό χώρο για να κάνουμε τέτοια συζήτηση στην χώρα μου. Και σιγά σιγά πέφτουν στην λησμονιά ορισμένα ζητήματα, ξεχνιούνται. Ethnical Russians, but ethnical Estonians are disappearing, and everyone because because the I think this is the most. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το θέμα αυτό, το ζήτημα είναι εξαιρετικά τοξικό στην ε, Εστονία. Οι Εστονοί, αυτοί που είναι πολίτες της Εστονίας, είναι καλοί άνθρωποι. Ε, και θυμάμαι πάντως ότι ε, πραγματικά και αυτοί ε, έχουν δίκιο όταν λένε ότι πέρασαν μια περίοδο όπου υπέστησαν πιέσεις έτσι ώστε η πρώτη γλώσσα που διδάσκονταν στα σχολεία να είναι η ρωσική. Ε, το ίδιο πράγμα είναι. Και έχω την αίσθηση ότι τώρα πια ε, ε, λειτουργούν σαν να έχουν όλα τα δικαιώματα. Λίγο σκεπτόμενοι, εμείς είμαστε οι πολίτες ε, της Εστονίας, εμείς έχουμε την εστονική υπηκότητα, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμως και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα πρέπει πια να αφήσουμε πίσω μας όλες αυτές τις πολυεθνικιστικές και ιδιαίτερως τοξικές συζητήσεις. Δεν το βλέπω όμως να γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να περάσω όλη μου τη ζωή συζητώντας για αυτά τα θέματα και μυρικάζοντας το θέμα του Στάλιν και αν οι Ρώσοι ήταν κατακτητές ή ξέρω εγώ τι. Όταν το θέμα θα έλεγα τίθεται σε επίπεδο ασφάλειας, της ύπαρξης δηλαδή των Εσθονών και των Λετωνών, μου θυμίζει ένα άλλο κράτος όπου είχε υποστεί ο λαός του κράτους αυτού, οι Ισραηλίνοι σαν παράδειγμα, μια υπαρξιακού τύπου απειλή θα έλεγα και την είχαν αισθανθεί. Συνεπώς λοιπόν αυτή η υπαρξιακή αίσθηση απειλής είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερα στην καρδιά της Ευρώπης. Αλλά το άκουσα σήμερα αυτό. Ελπίζω κάτι να γίνει τελικά. Όταν δημιουργήθηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν σαν βασική αρχή το όχι φορολογία αν δεν υπάρχει το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε ενώ εμείς πληρώνουμε φόρους χωρίς να έχουμε το δικαίωμα αυτό εδώ και 27 χρόνια. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εκπροσωπηθούμε πλέον σε όλα τα επίπεδα. Η κατάσταση έχει γίνει δηλητηριώδης πλέον για τους ε, πολίτες αυτούς της Εστονίας, γιατί για αυτήν μιλάω. Δεν μας είπατε πολλά για την αναφορά, αλλά όλοι οι συνάδελφοι έχουν πλήρη πρόσβαση στην αναφορά στο ίντρανετ του Κοινοβουλίου και πρέπει να τους έχει δοθεί και περίληψη στα αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο αναφερόμενος έχει α, ε, καταγγείλει την έλλειψη εκλογικών δικαιωμάτων των μη πολιτών, των λεγόμενων μη αναγνωριζόμενων πολιτών στην Εσθονία και τη Λετωνία. Τα εκλογικά θέματα είναι αυστηρά αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά σε σεβασμό βέβαια με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το ευρωπαϊκό δίκαιο δίδει κάποια εκλογικά δικαιώματα στους πολίτες, ιδιαίτερα όμως για τις ευρωεκλογές. Η συνθήκη της Ευρω... Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγει ότι οι βουλευτές εκλέγονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά πενταετία με μυστική ψηφοφορία. Και με την απόφαση του 86 το άρθρο 8 προβλέπει ότι η εκλογική διαδικασία ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος μέσω των εθνικών ρυθμίσεων. Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι εκπροσωπούνται άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 22 τμήμα 2, επίσης προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα και για τους εν κινήσει ε, πολίτες ότι ένας πολίτης ο οποίος ε, δεν είναι πολίτης της χώρας στην οποία έχει επίσημα εγκατασταθεί έχει το δικαίωμα όμως να συμμετέχει στις ευρωπαϊκές εκλογές κατά από προϋποθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επίσης έχει διευκρινίσει τα θέματα αυτά σε σχέση με την υπόθεση ε, Ισπανία εναντίον Ηνωμένου Βασιλείου. Προβλέπονται λοιπόν τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών, αλλά αυτό δεν αποκλείει τα κράτη-μέλη να διευρύνουν τα εκλογικά δικαιώματα αυτά και για άλλους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την σύσταση του εκλογικού σώματος. Στην υπόθεση Ντελβίνια επίσης το δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι το κάθε κράτος μέλος ορίζει το ποιος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις ευρωπαϊκές εκλογές σύμφωνα κιόλας με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απόφαση των λετονικών και εσθονικών αρχών να μην δώσουν το δικαίωμα στους, στην κατηγορία αυτών των πληθυσμών δεν θέτει θέμα διακρίσεων σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο για τους λόγους που προανέφερα. Συνειδητοποιούμε ότι η κατάσταση ε, των απροσδιορίστου ε, ηθαγένειας πολιτών στην Εσθονία και την ε, Λετονία είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πάρουν μέτρα και να μειώσουν τον αριθμό των πολιτών αυτών και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να αναφερθώ στην επιστολή που έστειλε ο Φραντ Τίμερμαν, ο πρώτο αντιπρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον προηγούμενο Νοέμβριο. Στην επιστολή αυτή επιβεβαιώνει Συγγνώμη, για μια στιγμή λέει η πρόεδρος, έχω την αίσθηση ότι οι συνάδελφοι έχουν διμερείς συζητήσεις μεταξύ τους και αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Αν θέλετε να κάνετε συζητήσεις παρακαλώ να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Λοιπόν, επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το θέμα της μείωσης του αριθμού των προσώπων χωρίς υπηκότητα, χωρίς ηθαγένεια συγγνώμη, είναι κάτι το σημαντικό Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να μειώσουν τον αριθμό των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Υπό το φως αυτών των σκέψεων θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση όταν ο κόσμος μπαίνω βγαίνει προφανώς αυτό δημιουργεί συχνά προβλήματα στους ομιλητές. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους για να πάρουν τον λόγο για την συγκεκριμένη αναφορά. Παρακαλώ πείτε μου ποιοι θέλετε να πάρετε το λόγο. Τώρα. Ο κύριος Μητροφάνοφ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα χρειαζόμαστε την υποστήριξη των Ευρωβουλευτών και την υποστήριξη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υποστήριξη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό όχι μόνο αναφερόμενος και όχι μόνο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν τις μειονότητες των κρατών μελών αλλά και 20.000 ε, κάτοικοι των χωρών της Βαλτικής έχουν υπογράψει αυτή την αναφορά. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μείνει απαθείς, παθητικοί καθόλου. Οι ΜΚΟ, οι ακτιβιστές, οι πολιτικοί που εκπροσωπούν τις εθνικές, εθνοτικές μειονότητες οργανώνουν δεκάδες συναντήσεις ε, Διαδηλώσει ε, διαμαρτυρίες. Είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στα δικά μα κοινοβούλια. Προτείνουμε δεκάδες ε, τροπολογίες και σχέδια τροπολογιών για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα των ανιθαγενών. Στη Λετωνία το 2012 προσπαθήσαμε να οργανώσουμε ένα δημοψήφισμα ώστε να χορηγηθεί η ηθαγένεια σε όλους, σε όλους τους μη πολίτες. Αλλά το κράτος μας απαγόρεψε να οργανώσουμε τέτοιο δημοψήφισμα. Απαγόρευσε δηλαδή σε πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στου πολίτε τη Λετωνία να ψηφίσουν υπέρ ε, του να γίνουν πολίτε ή μη πολίτε. Το έτος 2013 εμείς οργανώσαμε έναν ε, μη κυβερνητικό οργανισμό με το όνομα Κογκρέσο των Μη Πολιτών και σήμερα ήρθα εδώ φορώντας ε, το μπλουζάκι το οποίο τυπώσαμε πριν από δύο χρόνια με αυτό το σλόγγαν «Αφήστε το λαό μου να ψηφίσει». Αυτό ήταν το σλόγγαν μας ε, κατά τις δραστηριότητες αυτού του μη κυβέρνητου οργανισμού. Είναι πολύ σημαντικό, διότι πριν από τη σημερινή συνεδρίαση η κυβέρνηση της Λετωνίας έστειλε σε αυτή την Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα έναν τέτοιο χαιρετισμό. Μια πρόκληση συλλαμβάνοντας ε, τον αρχηγό του Κογκρέσου των Μη Πολιτών, τον ε, ο οποίος φυλακίστηκε. Άνθρωπος ο οποίος είχε εκλεγεί από μη πολίτες για να συμμετέχει στις συζητήσεις σε ειρηνικό διάλογο με την κυβέρνηση και τώρα τον έβαλαν στη φυλακή. Γιατί μόνο και μόνο διότι πρότεινε κάτι ε, στο διαδίκτυο. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας, χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Επιτροπής ε, και των άλλων ε, θεσμικών οργάνων, ώστε να διερευνήσουμε αυτή την υπόθεση των μη πολιτών και να βρούμε έναν τρόπο επίλυσης του προβλήματος αυτού. Παρακαλώ παραμένετε στο θέμα. Το θέμα είναι η συγκεκριμένη αναφορά. Το θέμα είναι τα δικαιώματα των μη πολιτών. Το θέμα είναι η αναφορά κύριε. Και ο αναφερόμενος που βρίσκεται εδώ εκπροσωπώντας τους υπογράφοντες δεν είναι εκδήλωση εδώ που μπορεί να πει κανείς ότι θέλει και να εκθέσει ό,τι θέλει η Επιτροπή αυτή. Παραμείνετε πιστή στο σημερινό θέμα. Κύριε Μάμικινς, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Για ένα τέταρτο του αιώνα οι μη πολίτε στη Λετωνία δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στις τοπικές, κοινοβουλευτικέ και σε ευρωεκλογέ. Είναι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Λετωνίας σας. Φανταστούμε αυτό το 12% σε ένα άλλο κρατος μέλος να είχε αποκλειστεί θα υπήρχαν ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιδράσει από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, την Κομισιόν, ανακοινώσει, αιτήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αν κανεί δεν βλέπει κάτι περίεργο σε αυτή την υπόθεση, αυτό είναι αυταρχικό. Πηγαίνετε να διαβάσετε ιστορία. Ε, φανταστείτε, ε, θυμηθείτε στην ιστορία όπου έχει χωριστεί ο λαός ενός κράτους σε δύο κατηγορίες, πολίτες και μη πολίτες. Έχω μια ερώτηση λοιπόν προς ε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωπο όλων σας πριν ψηφίσετε αγαπητοί συνάδελφοι. Φανταστείτε μια κατάσταση όπου, το, 12% του πληθυσμού δεν μπορεί να ψηφίσει σε καμία εκλογή σε ένα κράτος μέλος. Αλλά φανταστείτε αυτό να πάει στο 80%. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ρητορική ερώτηση. Mr. Κύριε Τσάκη. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ παλιά η ιστορία αυτή. Πολύ περίπλοκη, πολύ ευαίσθητη, ε, πολιτικά φορτισμένη ιστορία. Ουσιαστικά μία ερώτηση τίθεται εδώ. τίθεται ερώτημα ζήτημα αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ προσωπικά θα μπορέσω να υποστηρίξω αυτό το θέμα της ηθαγένειας για αυτούς τους ανηθαγενείς τους ρωσόφωνους και στις δύο χώρες εγώ να υποστηρίξω και το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές αλλά είμαστε εμεί αρμόδιοι γι' αυτό όπως είπε η Κομισιόν, αυτό είναι αρμοδιότητα του κρατου μέλους, της δικής του χώρας. Κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, θα συνιστούσα να ψηφίσουμε επί του θέματος αυτού. Και όποιος ψηφίσει υπέρ, θα ψηφίσει να κλείσουμε αυτή την αναφορά, αλλά μαζί με μια απόφαση να στείλουμε κάποιον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, μια επιστολή στην Κομισιόν και στη Λετωνική και στην κυβέρνηση ώστε να ξεκινήσει ένας νέος γύρος συζηνομιλιών και να τους απαιτήσουμε να βρουν μια λύση. Και όποιος ψηφίσει κατά ψηφίζει στο να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά αλλά με τον ίδιο τρόπο να στείλουμε μια επιστολή στην Κομισιόν και στα ε, δύο κράτη-μέλη και να τα ρωτήσουμε αν μπορεί να γίνει ένας νέος γύρος εξέφραση λύσεων. Χρειαζόμαστε μια λύση, αλλά η λύση δεν είναι δική μα αρμοδιότητα. Μπορούμε να καθόμαστε να το συζητάμε, να το συζητήσουμε και, το πρωί, και αύριο το πρωί, αν θέλετε, αλλά δεν νομίζω να βρούμε λύση. Θα χρειαστεί να αποφασίσουμε με ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Για πρώτη φορά ακούω κάποιον που μου κάνει μία πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο να προχωρήσουμε. Γι' αυτό είπαμε να έρθει εδώ ο αναφερόμενος έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη. Ευχαριστώ κύριο Μάντα. Ευχαριστώ ε, πολύ. Σύμφωνο απολύτως με τον συνάδελφο Τσάκη που μίλησε προλίγο. Όταν προτείνει να κλείσουμε αυτήν ε, την αναφορά. Όμως θα ήθελα να κάνω και κάποια επιπλέον σχόλια. Πρώτα απ' όλα, έχω την αίσθηση ότι η συζήτηση αυτή έγινε πολύ σε συγκινησιακό επίπεδο και λιγότερο ε, σε όρους ε, ε, δημοκρατίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι η δημοκρατία είναι μια τεράστια εφεύρεση ε, της ε, ε, κοινωνίας και βεβαίως η κοινοβουλευτική δημοκρατία, η δυνατότητα εκπροσώπησης, η δυνατότητα του εκλέγη, του εκλέγεστε φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Όμως είναι γεγονός ότι τα κράτη-μέλη και οι ε, πώς να σας το πω, οι εκλογικές περιφέρειες ας πούμε να, που πρέπει να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εκλογική διαδικασία είναι ένα θέμα που άπτεται της επικουρικότητας και ένα θέμα που άπτεται και της ε, εθνικής ανεξαρτησίας, κυριαρχίας συγγνώμη. Ε, δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν κεντρικά οι Βρυξέλλες για τέτοια πράγματα, για το πώς οι περιφέρειες της Ευρώπης, οι ε, χώρες της Ευρώπης θα λύσουν τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τούμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να πω διάφορα πράγματα. Ακούσαμε σήμερα από κάποιους συναδέλφους ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι υπεύθυνοι, δεν είναι η Εστονία υπεύθυνη για αυτούς. Όχι. Εκεί ζουν, δεν πάνε πουθενά άλλου. Ακούσαμε επίσης ότι η ε, διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορούν να δεχτούν ε, τους απάτριδες. Όχι. Ο, οπουδήποτε της γης καταπολεμάται το φαινόμενο αυτό των απάτριδων Τρίτον, υπόθηκε ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν ε, εστονική υπηκότητα. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι δυνατόν να τα... Ε, ε, είναι λίγο ο φαύλος κύκλος. Εάν δεν έχεις πρόσβαση σε κάτι, μπορεί να βρεις και χίλιους λόγους για να πεις «Μα δεν με ενδιαφέρει αυτό το κάτι». Είναι, είναι αυτό ότι ε, δεν με νοιάζει κιόλας, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά όσα δεν φτάνει η Αλεπού. Είπε η ομιλήτρια. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχει αποδειχθεί επανειλημμένα και από πάρα πολλές μελέτες ότι 54% των απατρίδων ε, στην χώρα μου λένε ότι δεν είναι σε θέση να περάσουν τις εξετάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη γλώσσα, για την ιστορία κτλ. έτσι ώστε να αποκτήσουν μέσω πολιτογραφήσεως την ιδιότητα του πολίτη. Κοιτάξτε, είναι σαφή τα πράγματα. Δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να περάσουν τις εξετάσεις αυτές, γιατί είναι μεγάλοι άνθρωποι. Και ε, την ίδια ώρα, ακριβώς επειδή είναι μεγάλοι άνθρωποι, δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν άλλες εναλλακτικέ λύσεις. Ε, ε, σύμφωνα με τον αριθμό του, του πληθυσμού έχουν δοθεί ε, οι θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά εδώ υπάρχουν, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τον αριθμό αυτών που έχουν την, το καθεστώς του πολίτη. Ε, ε, υπάρχει και κάτι άλλο που αναφέρθηκε ο συνάδελφος ε, προηγουμένως. Είναι το, το είπε ο εκπρόσωπος του Σεργέη Στεπάνοφ προηγουμένως. Δηλαδή ε, ε, το ζήτημα είναι ότι ε, πληρώνουμε φόρους. Πληρώνουμε φόρους στην Εστονία, πληρώνουμε φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουμε την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η Ρωσία. Και ανοίγουμε, στρώνουμε χαλί για τη Ρωσία και αυτό δεν είναι πάρα πολύ έξυπνο. Επίσης υπόθηκε ότι ε, είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους ε, δεν επιλέγουν την πολιτογράφηση ε, κάποιοι πολίτες. Κοιτάξτε, με κάποιο τρόπο όμως θα πρέπει να γίνουν στον οι πολίτες από τη στιγμή που συμμετέχουν στην κοινωνία και πληρώνουν. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε κυρία Πρόεδρε, να, να μου επιτρέψετε λέω να δείξω ένα βίντεο πολύ μικρό, δύο λεπτών δεν θέλω να πείσω απαραίτητα τους ανθρώπους που δεν ήταν πριν εδώ, που δεν άκουσαν την συζήτηση. Ε, και δεν μπορώ ε, να πείσω και τους ανθρώπους που είναι τόσο σίγουροι για αυτό που σκέφτονται, που είναι απλώς ε, έτοιμοι να πατήσουν το κουμπάκι χωρίς να καθίσουν, να σκεφτούν, να ακούσουν κτλ. Ε, πρόεδρος, δεν είναι δυνατόν να σας, ε, να σας δώσω αυτή την άδεια τη στιγμή που κανένας άλλος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, εγώ μίλησα για το θέμα αυτό στην ομάδα, μίλησα και με την γραμματεία της Επιτροπής. Ναι, κοιτάξτε, εγώ έχω το προνόμιο να είμαι πρόεδρος τούτη τη Επιτροπής. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μα. είναι πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι σε άλλες περιπτώσεις θα ήθελαν να δείξουν επίσης παρόμοια βιντεάκια, φιλμάκια κλπ. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε προσκολλημένοι κατά κάποιο τρόπο ε, και να εστιαστούμε μονάχα στο περιεχόμενο αυτής της αναφοράς. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Πάμπλεξ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, έκλεισε το μικρόφωνο. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο σε τούτη την αναφορά και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το εργαστήριο το οποίο οργανώθηκε. Προηγουμένως ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα σχόλια στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου. Νομίζω ότι τώρα έφτασε η ώρα να εξάγουμε τα τελικά συμπεράσματα και να προχωρήσουμε πια νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε να κλείσει αυτή η αναφορά προς ώρας διότι πολύ πολύτιμος χρόνος δαπανήθηκε για το θέμα αυτό. Νομίζω όλοι όσοι ήθελαν να κατανοήσουν το πρόβλημα των απάτριδων ή των ε, ανθρώπων που δεν έχουν ε, ε, την ιδιότητα του πολίτη, άκουσαν, έμαθαν, κατάλαβαν. Ευχαριστώ. Η κυρία Καπεθών Ρουίς. Πολύ σύντομα. επανειλημμένα έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτών των πολιτών. Είναι βεβαίως ένα περίπλοκο ε, ζήτημα ε, και που ε, διαχωρίζει ακόμα και πολιτικές ομάδες. Αλλά εδώ μιλάμε για πολίτες, άνδρες και γυναίκες και μιλάμε και για θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να έχουμε μία σωστή θέση. Τώρα μία μετακίνητη θέση και ρητή είναι δύσκολο να έχουμε για τέτοια θέματα. Στην ε, τελευταία ε, διεύρυνση είχαμε συζητήσει για, τους, για το θέμα των πολιτών. Εδώ βέβαια γίνεται λόγος ε, για αρμοδιότητες. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι η διπλωματική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν νομίζω ότι, νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτήν την αναφορά. Θα πρέπει να στείλουμε ε, ε, επιστολές ε, στα Υπουργεία Εξωτερικών των χωρών και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε και την ενωσιακή διπλωματία υπέρ του θέματος. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κυρία Κούνεβα. και την πρόταση μου μετά. δεν μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά με τίποτα, γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη γνώση εμείς εδώ. Προτείνω αυτή η αναφορά να συζητεί μαζί με την, με Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έτσι ώστε να έχουμε εξειδικευμένους συνάδελφους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε μόνο ουσία. Εδώ μπορούμε να κάνουμε προπαγάνδα, εδώ μπορούμε να έχουμε προσωπικά μα ενδιαφέροντα, αλλά εδώ θέλει ουσία. Γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να ενταχθεί 12% πληθυσμού μια χώρα. Παλεύουμε για τη Ρωμά, οι οποίοι είναι αγράμματοι, δεν ξέρουν τη γλώσσα και δίνουμε τόσο λεφτά και προσπαθούμε να του εντάξουμε στην κοινωνία. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια μόρφωση και λόγω τη αλλαγή δεν έχουν καταφέρει να μάθουν τη γλώσσα και δεν είναι ενταγμένοι στην κοινωνία είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ ακραίο σαν λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν έχουμε υπόψη 12% πολιτών κάποια χώρα. Ευχαριστώ. No, sorry, sorry, I didn't. I, I, I wasn't talking to, to Mr. Pett. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μιλάμε για τις 161.000 στην Εστονία που έμαθαν την εστονική γλώσσα, πέρασαν τις εξετάσεις, και μπόρεσαν να πάρουν την εστονική υπηκότητα. Τα τελευταία 27 χρόνια από τότε που υπάρχει η ανεξαρτησία της χώρας, αυτοί οι άνθρωποι στα 27 χρόνια θα μπορούσαν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία κατοικούν. Γι' αυτό παρακαλώ πρέπει να καταλάβετε ποια είναι τα κίνητρα όλοι οι άνθρωποι αυτοί είχαν την δυνατότητα να πάρουν την υπηκότητα την εσθονική ή την λετονική αν περνούσαν τις εξετάσεις, αν μάθαιναν τη γλώσσα της χώρας που τους φιλοξενεί. Το ίδιο ισχύει για όλες τις χώρες σας. Αν κάποιος θέλει την υπηκότητα της χώρας σας, ε, θα πρέπει κάτι να ξέρει τώρα για τη γλώσσα της χώρας. Θα πρέπει να γνωρίζει λεπτομέρειες για την συνταγματική τάξη, και η Εστονία και η Λετονία δεν είναι διαφορετικές από τις δικές σας χώρες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 161.000 άνθρωποι έμαθαν τα τελευταία 27 χρόνια την εσθονική γλώσσα και πήραν την επικότητα. Πριν μερικά χρόνια, όταν η Ρωσία αποφάσισε να μην ζητά θεωρήσεις για αυτούς οι οποίοι είχαν διπλή υπηκότητα, ε, μειώθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που ζητούσαν την υπηκότητα την εστονική, γιατί κυκλοφορούν ελεύθερα τώρα με τη Ρωσία είναι κάτι το οποίο τους απαλλάσσει από γραφειοκρατικές ενέργειες και από ιδιαίτερο κόστος. Γι' αυτό λοιπόν όταν παίρνετε κάποιες αποφάσεις παρακαλώ να βλέπετε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι ευθύνη έτσι και αλλιώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δημιουργήσετε ένα προηγούμενο με το θέμα αυτό, τότε θα μπορούν να υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα από πάρα πολλές ε, χώρες μέλη που δεν ε, υποτίθεται σέβονται το δίκαιο το ευρωπαϊκό όπως θα έπρεπε. Και είναι δύσκολη η ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις που έχει κάθε χώρα σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι παραδοσιακοί απάτριδες. Όλοι αυτοί έχουν το δικαίωμα να πάρουν την υπηκότητα αρκεί να μάθουν την γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν και να περάσουν από την εξέταση αυτή. Αλλά θα πρέπει να δούμε γιατί δεν το έκαναν αυτό οι άνθρωποι τα τελευταία 27 χρόνια. Σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλους εδώ ομιλητές όχι, δεν πρέπει να σας ξαναδώσω το λόγο για τρίτη φορά. Θα πρέπει να επανέλθουμε στον αναφερόμενο τώρα. Περιμένει υπομονετικά. Θα μας κάνει ένα τελευταίο σχόλιο. Έχετε την δυνατότητα να αντιδράσετε σε αυτά τα οποία μόλις ακούσατε και μετά θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να σας ζητήσω να στείλετε μία επιστολή στα Εθνικά Κοινοβούλια και στις χώρες τις συγκεκριμένες έτσι ώστε να μας βοηθήσετε και οι άνθρωποι αυτοί να ακουστεί η φωνή τους περισσότερο από ό,τι σήμερα. Είναι δύσκολο να ζει κανείς κατά από τις συνθήκες αυτές. Όταν γνωρίζει ότι δεν έχει κανέναν βουλευτή ο οποίος τους εκπροσωπεί. Συνεπώς λοιπόν είτε ψηφίσετε υπέρ του να μείνει ανοιχτή η αναφορά είτε όχι έχει σημασία να στείλετε τις επιστολές αυτές και να επιστήσετε την προσοχή των ενδιαφερομένων. Είναι ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός. Λοιπόν για μένα ήταν ε, χωρίς προηγούμενο η συζήτηση αυτή. Χαίρομαι που θα πάρω την πρότασή σας σοβαρά να κλείσουμε την ε, συζήτηση αυτή όπως είχε πει και ο κύριος Τσάκη, δεν χρειάζεται να στείλουμε επιστολές στην Επιτροπή, έτσι κι αλλιώς είναι παρόντες, αλλά μπορούμε να στείλουμε επιστολές στην μόνιμη, στους μόνιμους αντιπροσώπους και να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Για ένα διαδικαστικό, η κυρία Τούμα. θέλω να κάνω μια άλλη πρόταση. Αν είναι δυνατόν Όπως είπε πολύ σωστά η εκπρόσωπος της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές έχει στείλει ισχυρά πολιτικά μηνύματα ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να επιληθεί. Οπότε προτείνω να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να διοργανώσουμε μια διερευνητική αποστολή. Δεν σημαίνει ότι θα παρέμβουμε σε εσωτερικά θέματα των κρατών μελών, απλά θα δώσει ένα ισχυρό ένα χειρό πολιτικό μήνυμα. Πρόεδρος και όπως γνωρίζετε δεν λαμβάνουμε αποφάσεις για τέτοιες επισκέψεις εδώ. Πρέπει να συζητηθεί στους συντονιστές ε, οι οποίοι θα το παρουσιάσουν στην ομάδα των συντονιστών. Αλλά το σημειώνουμε αυτό που λέτε. Και τώρα λοιπόν ας κάνουμε τα εξή. Θα στείλουμε τις επιστολές, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πρέπει να κλείσουμε εδώ με τον τρόπο που ανέφεραν ε, και οι συνάδελφοι και ο αναφερόμενος. Θα ήθελα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Οπότε σας παρακαλώ, αν δεν έχετε τις κάρτες σας μαζί σας, σηκώστε το χέρι σας και θα προσπαθήσουμε να καταμετρήσουμε όλους. Όσοι έχετε κάρτα ψηφοφορίας, βάλτε τη στο μηχάνημα τώρα. Και καθώς ε, κάνετε αυτό τώρα εγώ θα ήθελα να ζητήσω την προσοχή των Συμβουλών Πολιτικής. Την προσοχή σας παρακαλώ. Βεβαιωθείτε ότι το ΕΛΚ έχει εννέα που να ψηφίσουν ούτε λιγότερους ούτε παραπάνω. Οι σοσιαλιστές το πολύ οκτώ. Το ECR το πολύ τέσσερις ψήφους το ECR το πολύ τέσσερις ψήφους, Άλτε τρεις ψήφοι, το πολύ, Πράσινη το πολύ τρεις ψήφοι, Γκουε τρεις ψήφοι και η FDT επίσης τρεις ψήφους. Είναι απόλυτα σαφές για όλους. Το γνωρίζετε αν έχετε δικαίωμα ψήφου εδώ ή όχι. Οπότε ας ψηφίσουμε. Ποιος θα ήθελε να κλείσουμε την αναφορά και να στείλουμε τις επιστολές όπως μόλις είπα δύο φορές. Πατήστε το πράσινο κουμπάκι, είναι ψήφος ε, ναι αυτή. Και όσοι θέλετε να μην είναι ανοιχτή, ψηφίστε όχι με το κόκκινο κουμπί. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is now open. And you raise your hand. Και σηκώστε και το χέρι σας για ναι ή όχι. Σοσιαλιστές, ε, έχετε μία ψήφο παραπάνω. Βγάλτε μία ψήφο. Ε, κάποιον από τους πληρωτές βγάλτε. Ο συντονιστής ή ο σύμβολος πολιτικής αποφασίζει. it be fine. Τώρα νομίζω είναι εντάξει. Και επίσης έχουμε ανθρώπους που δεν ψηφίζουν εξακολουθεί να είναι ανοιχτή ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε ακόμη. Τώρα έχουμε ένα ΕΛΚ παραπάνω. Τώρα είναι εντάξει. 31 κάρτες έχω στα μηχανήματα, αλλά μόνο 27 έχουν ψηφίσει. Τελειώσαμε όμως, πέρα της ψηφοφορίας. Κλείνουμε την ψηφοφορία. πρέπει να υπολογίσουμε και μία ψήφο με ανάταση χειρός αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι κατά μία ψήφο, με μία ψήφο διαφορά έχουμε αποφασίσει να, κληθεί, να κλείσει αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, δεν θα είναι όλοι παρόντες όταν ασχοληθούμε με την 6.36 παρακαλώ να φύγετε από την αίθουσα ε, αλλιώς ε, ξεκινάμε αμέσως Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την συγκεκριμένη αναφορά 636 εξ ονόματος της ε, Ένωσης αφαράννα και του Φόρου Ανταλούς ΠΑΘΙΕΝΤΕΣ για το σύστημα προμηθειών φαρμακευτικών ε, παρασκευασμάτων στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας. Είναι η Τερέσα Μαρτίν Χιμένες από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Α, όχι, κάποιο λάθος έχω κάνει εδώ. Εσείς είστε πρόεδρος της Αφαράν. Εγώ είμαι η πρόεδρος της Αφαράν. Έχετε το ίδιο σχεδόν όνομα με τη συνάδελφό μας. Α, τι σύμπτωση ένα γράμμα διαφορά έχετε με την άλλη κυρία Χιμένες, την συνάδελφο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα τα πω σχετικά γρήγορα. Λοιπόν, εγώ είμαι υπεύθυνη σε θέματα φαρμακευτικής Δεν έρχομαι εδώ σαν φαρμακόπιος, ε, εκπροσωπώ την Ένωση Ασθενών της ε, Ανδαλουσίας, 50 επιμέρους ε, οργανισμοί εκπροσώπησης ασθενειών και έρχομαι εδώ να σας ζητήσω. Οι ασθενείς της Ανδαλουσίας να σας πω ότι υφίστανται διακρίσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους Ισπανούς. Κοιτάξτε, η περηφάνεια της Ισπανίας είναι το εθνικό σύστημα υγείας και υπάρχει θεωρητικά ε, δωρεάν φαρμακευτική ε, αρρωγή. Αλλά ε, η Υπάρχει ένας κατάλογος φαρμάκων σε όλη την Ισπανία με πάνω από 2.000 φάρμακα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλά ε, στην Ανδαλουσία είναι πάρα πολύ ε, μικρός ο αριθμός αυτός και στην ουσία ο ε, Ανδαλουσιανός ασθενής υφίσταται διακρίσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους Ισπανούς ασθενείς. Προσφεύγει λοιπόν στην κοινωνική ασφάλιση της περιφέρειας με μια συνταγή η οποία όμως σε επίπεδο επιλογής είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Στην ουσία δηλαδή δημιουργούνται προβλήματα γίνεται ένας διαγωνισμός και στην ουσία κερδίζει κάθε φορά ένα εργαστήριο φαρμακευτικό και χρησιμοποιείται για όλες τις ασθένειες της συγκεκριμένης μορφής μία φαρμακευτική ουσία. Τα εργαστήρια τα οποία συμμετέχουν στους διαγωνισμούς αυτούς και δίνουν πρόσφορες είναι σχετικά εξωτικά θα έλεγα και φοβόμαστε ότι δεν έχουν επαρκείς ικανότητες παρασκευής των κατάλληλων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Υπάρχουν επίσης προβλήματα ποσότητας, υπάρχουν φάρμακο όπως το ομοιοπλασόλ τα οποία είναι διαθέσιμα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό και υπάρχει συγκεκριμένη έλλειψη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ναι, μεν εξοικονομεί χρήματα αλλά στην ουσία πολλές φορές παρεμποδίζει την προσφυγή του ασθενού σε συγκεκριμένη θεραπεία, μειώνει την ποιότητα της θεραπείας την, η οποία παρέχεται. Η περιφερειακή κυβέρνηση δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα Στην a Σε περιπτώσει υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν σχέση και με την ονοματολογία των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται. Είναι ανεπαρκείς οι ουσίες αυτές και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Τώρα λοιπόν όπως είπα η περιφερειακή κυβέρνηση δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αλλά στην παρούσα φάση βλέπουμε ότι ενώ είναι 10.000 τα φάρμακα τα οποία είναι διαθέσιμα στο σύνολο της Ισπανίας, ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μικρός ε, στις, ε, στην περιοχή της Ανδαλουσίας και στην ουσία υφιστάμεθα διακρίσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ισπανία και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρόκειται για μια σοβαρή υποβάθμιση σε επίπεδο διάθεσης φαρμακευτικών ουσιών Στόχος των φαρμακοποιών είναι να εξυπηρετούν σωστά τους ασθενείς μετά από τις κατάλληλες σπουδές και να τους διαθέτουν τις καταλληλότερες και καλύτερες φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες είναι κάθε φορά διαθέσιμες. Και ο γιατρός, ο βασικός λόγος ύπαρξης του ιατρού είναι ακριβώς ο ασθενής με τον γιατρό ο ασθενής καταπολεμά την ασθένεια, θεραπεύεται χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες φαρμακευτικές ουσίες. Συνεπώς, θα ήθελα να σας ζητήσω, κοιτάξτε σας έδωσα το λόγο για πέντε λεπτά, έχετε χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο και γι' αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσετε. Έρχομαι λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταπεινά να ζητήσω να ασκήσετε τις αρμοδιότητες τις οποίες έχετε και να κρατήσετε ανοιχτή τη συγκεκριμένη αναφορά. Μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ασθενείς, πρέπει να την χάνουν τη σωστής θεραπείας και γι' αυτό σας ζητώ παρακαλώ να βοηθήσετε έτσι ώστε η μοναδική περιφέρεια της Ευρώπης στην οποία ισχύει αυτή η κατάσταση ε, να αντιμετωπιστεί. Έχει συζητηθεί το θέμα και πρέπει να συζητηθεί εκ νέου και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή ΙΝΚΟ γιατί είναι και θέμα θα έλεγα εμπορικό ε, δεν πρέπει να δημιουργούνται εκ των υστέρων μονοπόλια Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός και σε σχέση με τα φάρμακα και δεν θα πρέπει να παραμείνει έτσι η κατάσταση. Πρόεδρος, νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ποιες είναι οι παρατηρήσεις της Κομισιόν όσον αφορά αυτήν την αναφορά. Ε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά ε, τις ελλείψεις, ε, τις τρελούμενες ελλείψεις φαρμάκων λόγω των διαδικασιών διαγωνισμού. Πρέπει να, σπο, να σας πω ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της ε, ε, πολιτικής υγείας καθώς επίσης και της ε, καθώς επίσης ε, και όλες τις ε, allocation of και όλες τις φροντίδες ε, υγείας και τις θεραπείες. Η διαδικασία διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων λοιπόν βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα στον τομέα των φροντίδων υγείας, παροχής φροντίδων υγείας ε, και ε, δεν ε, καλύπτονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα φάρμακα από τις διαδικασίες διαγωνισμούς. Όσον αφορά τις ελλείψεις φαρμάκων και σκευασμάτων, κατανοούμε το πρόβλημα και πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη ευαισθησία βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά μονάχα την Ανδαλουσία αλλά και άλλες περιφέρειες της Ευρώπης. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα όσον αφορά την οργάνωση ε, του συστήματος ε, υγείας ε, είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε παράγουν αρκετά προγράμματα, συγγνώμη, φάρμακα, προϊόντα έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία έλλειψη φαρμάκων. Μπορούμε επίσης να ε, στείλουμε και να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με τρόπους ε, ώστε να μην προκύψουν ελλείψεις. Όσον αφορά τα όσα καταγγέλει η αναφέρουσα ε, για προβλήματα και κινδύνους που ενέχει το σύστημα, πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά το θέμα αυτό, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φαρμακευτικά προϊόντα ε, είναι πάρα πολύ ε, αυστηρή. Ε, τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά του κράτους μέλους παρά μόνο εάν έχουν ήδη μία αδειοδότηση ε, εμπορίας ε, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ε, του κράτους μέλους ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα γενώσιμα ισχύει αυτό για οποιαδήποτε φαρμακευτικά προϊόντα τοποθετούνται, εισάγονται στην αγορά θα πρέπει να έχει προηγηθεί αυτή η αδειοδότηση. Είναι σαφές ότι με τα χρόνια υπάρχουν όλο και περισσότερες δραστικές ουσίες ε, αλλά όλα τα προϊόντα αυτά οποτεδήποτε και εφόσον ε, μπαίνουν στην αγορά σημαίνει ότι έχουν λάβει εκ των προτέρων ε, αδειοδότηση. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ελέγχονται ε, τα στοιχεία ποιότητας ε, όλων των προϊόντων και όλων των σκευασμάτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ε, η καλή ποιότητα και η υγεία των ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει, επαναλαμβάνω, αυτή η αδειοδότηση, η πρώτερη της εμπορίας του προϊόντος. Όσον αφορά τις δραστικές ουσίες, καθώς επίσης ε, και της ε, πρακτικής που αναφέρει η αναφέρουσα σύμφωνα με την οποία ε, συνταγογραφούνται οι δραστικές ουσίες ε, πρέπει να σας πω ότι και για το θέμα αυτό αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία επιτρέπουν τη συνταγογράφηση είτε μέσω συγκεκριμένου σκευάσματος είτε μέσω της αναφοράς δραστικών ουσιών. Μπορεί να δώσει δηλαδή είτε το brand product είτε το γενώσιμο. Ωστόσο, ε, οποιαδήποτε και αν είναι η επιλογή, ε, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του προϊόντος ε, το οποίο προωθείται στην αγορά. Να σας πω ότι η νέα νομοθεσία αποδίδει την ευθύνη όλου του συστήματος υγείας αλλά και των διαδικασιών διαγωνισμού για φαρμακευτικά ε, προϊόντα στα χέρια των ε, κρατών μελών. Αυτά μπορώ να απαντήσω στην αναφέρουσα. Πρόεδρος, ε, Πληροφορήθηκα επίσης ότι έχουμε εκπρόσωπο της κοινότητας της Ανδαλουσίας και επομένως ε, θα δώσω στην εκπρόσωπο το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε αυτά τα δύο λεπτά εξ ονόματος της κυβέρνησης της ε, Ανδαλουσίας ε, την οποία εκπροσωπώ εδώ στις Βρυξέλλες και ενώπιον του Κοινοβουλίου πρέπει να σας πω ότι είναι η κυβέρνηση της Ανταλουσίας απολύτως δεσμευμένη να ε, ε, διαβολούνται δεσμευμένοι για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις διαδικασίες διαγωνισμών για φαρμακευτικά προϊόντα που είναι άλλωστε ε, δημόσια στοιχεία. Πιστεύουμε ότι το σύστημα αυτό είναι σωστό και εμείς ακολουθούμε αυτήν την φαρμακευτική πολιτική στην οποία εντάσσονται και οι διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ήδη τρεις φορές το συνταγματικό δικαστήριο της Ισπανίας έχει δώσει πράσινο φως αυτή την διαδικασία και άλλωστε ε, έχει ε, δοθεί και πράσινο φως όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα του προγράμματος προγράμματο αυτού, όπως είπε και η εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να πω στην αναφέρουσα ότι οπωσδήποτε ε, και σας διαβεβαιώ έχουν εξοικονομηθεί και πόροι και χρήματα τα οποία ε, δίνονται στη συνέχεια στο σύνολο του συστήματος υγείας της κοινότητας της Ανταλουσίας. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή η επιβεβαίωση του συνταγματικού δικαστηρίου ε, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και επομένως δεν είναι δυνατόν ε, να πει κανείς ε, ότι δεν υπάρχει ελευθερία πρόσβασης στα ε, φάρμακα. Και πρέπει να σας πω ότι το σύνολο των εκπροσώπων των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ισπανία επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα αυτό είναι σωστό και μάλιστα ζητούν να εφαρμοστεί στο σύνολο της Ισπανικής επικρατείας. Is σας έδωσα δύο λεπτά και τα χρησιμοποίησατε. Είχα την εντύπωση ότι είχατε ολοκληρώσει. Ε, ε, ολοκληρώσατε, τελειώσατε, γιατί σας έδωσα δύο λεπτά και ήδη τα ξεπεράσατε. Τώρα, ε, ε θα δώσω το λόγο στα κράτη, στους βουλευτές, η κυρία Καμπεσόν Ρουής. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και την αναφέρουσα. Να σας πω ότι εκπροσωπεί την ε, οργάνωση, των, ε, ε, την οργάνωση Αφαράν και όχι το σύνολο των φαρμακοποιών. Επανειλημμένα συζητήσαμε τα θέματα αυτά στην Ανδαλουσία. Υπάρχουν οι αποφάσεις του ε, συνταγματικού ε, δικαστηρίου και εδώ τελικά ε, προφανώς πρόκειται για μια συζήτηση πολιτική ή μια συζήτηση που αφορά συγκεκριμένα συμφέροντα. Εγώ έγινε λόγος για την ποιότητα των σκευασμάτων και τα λοιπά. Κοιτάξτε, ε, είχαμε τη συζήτηση αυτή ε, όταν σε επίπεδο Ισπανίας και όχι Ανδαλουσίας ε, συζητήθηκε το θέμα των δραστικών ουσιών και οι γιατροί είπαν ότι μπορούμε να γράψουμε και τις, να συνταγογραφήσουμε και τις δραστικές ουσίες. Τώρα, η, αυτό που αποφάσισε η κοινότητα της Ανταλουσίας είναι ότι δεν διαπραγματεύεται το θέμα της επιλογής ε, ο φαρμακοποιός αλλά συνολικά η Ανδαλουσία ε, και, ε, και ότι το σύστημα αυτό μπορεί να αποβεί σε όφελος όλων των πολιτών και όλων των ασθενών. Τώρα, εάν σε κάποιον δεν αρέσει αυτό είναι δικαίωμά του. Ξέρω ότι εδώ έχουμε και εκπρόσωπο ε, των Ισπανών βουλευτών του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας ε, που μπορεί να μην του αρέσει αυτή η κατάσταση αλλά δεν είναι δικό μας θέμα. Ε, φαντάζομαι ότι θα, θα μου πείτε κι εσείς διάφορα στοιχεία. Κοιτάξτε, εγώ εκπροσωπώ τους, ε, τους ε, ασθενείς της Ανδαλουσίας. Δεν θέλω τίποτα άλλο να εκπροσωπήσω. Κοιτάξτε, λέει η πρόεδρος, εγώ είμαι πρόεδρο. Εάν θέλετε να πάρετε τον λόγο, θα σηκώσετε το χέρι σα, θα σα τον, τον δώσω. Δεν μου αρέσουν αυτού του είδου οι παρεμβάσει δεξια δεξιά-αριστερά. Ζητώ συγγνώμη, λέει η κυρία Καμπεσόν Ρουίς. Εγώ απλώ ε, ήθελα να πω ότι ότι φαίνεται ότι όλα αυτά τα ζητήματα ε, ε, κεντρίζουν την περιέργεια των βουλευτών του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι στην Ισπανία ε, είναι η ισπανική κυβέρνηση αυτή η οποία καθορίζει ε, τα φάρμακα τα οποία ε, πληρώνει, για τα οποία πληρώνει η κοινωνική ασφάλιση. Καθορίζεται στην, σε, επίπεδο Ισπανίας. Ωστόσο, ο, ο νόμος στο σύνολο των περιφερειών και όχι μονάχα στην Ανδαλουσία προβλέπει ότι μπορεί να γίνει συνταγογράφηση βάσει των δραστικών ουσιών ε, στην Ανδαλουσία έγινε η επιλογή για μια δημόσια και διαφανή διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση γιατί οι δραστικέ ουσίε ε, είναι ποιοτικέ, το είπε και η εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να σα πω ότι και η Ισπανική Οργάνωση Φαρμάκου, όχι τη Ανδαλουσία, τη Ισπανία, ε, ε, δεν αμφισβήτησε ότι η συνταγογράφηση τη δραστική ουσία είναι κάτι σύνομο και ε, ε, ε, υπάρχουν σε όλες τις χώρες ένα σωρό φάρμακα τα οποία έχουν γίνει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προέρχονται από την Ασία, προέρχονται από αλλού. Εν πάση περιπτώσει, εδώ το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί εδώ μιλάμε για, μια, για ένα ζήτημα το οποίο είναι δεοντολογικό, το οποίο άπτεται της ηθικής γιατί εδώ υπάρχει η υπόνοια και η καταγγελία ότι στην Ανταλουσία δίνουμε φάρμακα τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία. Έχουμε 200 φάρμακα, ναι, 216 για την ώρα, ε, τα οποία δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου από τη διαδικασία διαγωνισμού ε, της ε, Ανδαλουσίας. και, ε, και ο ίδιος ο διαμεσολαβητής ε, ανέφερε ότι το 90% των φαρμάκων δεν έχουν κανένα ε, πρόβλημα, δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα για την υγεία. Και όταν λείπει ένα φάρμακο, όχι λόγω της διαδικασίας διαγωνισμού, όχι δηλαδή από τα φάρμακα αυτά τα οποία περνούν μέσα από τη διαδικασία των διαγωνισμών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, αυτό οφείλεται σε άλλους λόγους και όχι στη διαδικασία διαγωνισμού για τα φαρμακευτικά Νομίζω λοιπόν ότι ε, το θέμα ε, δεν είναι ε, πόσα φάρμακα φτάνουν στο φαρμακείο ή αν υπάρχει κάποια έλλειψη ή οτιδήποτε. Όταν πάει κάποιος ε, στο φαρμακείο, το φάρμακο το οποίο ζητήσει, έχει ζητήσει να του δώσουν. Το φάρμακο το οποίο έχει συνταγογραφήσει ο, ο γιατρός. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αποτελεσματικότητας, κανένα πρόβλημα υγείας. Είναι καθαρά πρόβλημα πολιτικών σκοπιμοτήτων. 70% των ε, ε, γενοσύμων ε, περνάει μέσα από διαγωνισμούς προβλήμα. Από διαγωνισμού για φαρμακευτικά προϊόντα στη Γερμανία. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πρόβλημα αυτό στην Ανδαλουσία. Τελειώνω λέγοντα το εξή. Από το 2012, 426 φάρμακα έχουν βγει από την δημόσια κρατική ε, ε, παρέμβαση. Ε, αυτό σημαίνει ότι 4 εκατομμύρια από το 12 που πλήρωνε το δημόσιο σύστημα υγείας άρχισαν να το πληρώνουν οι, οι ασθενείς, οι πολίτες εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνταξιούχοι. Μη μου λέτε λοιπόν αυτά για την αποταμίευση ή για τη φαρμακευτική δαπάνη. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση μόνο. Ε, θα έχουμε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον χρόνο τον οποίο είχε η κυρία Καμπεθόν. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε. Ξέρετε, μερικές φορές ε, Έχουμε ελάχιστο στην αρχή, όπω συνέβη όταν ήθελε να πάρει το λόγο η κυρία Καμπεσόν. Οπότε εκεί μπορώ να τη δώσω χρόνο. Προσπάθησα να τη πω πολλέ φορέ ότι δεν υπήρχε αρκετό χρόνο. Έχουμε μέχρι τι 6 και μισή. Και οι συνάδελφοι εδώ δυστυχώ δεν θα μπορέσουν να έχουν τον ίδιο χρόνο, διότι προσθέθηκε κόσμο στον κατάλογο καθώ αυτή μιλούσε. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Τι να κάνω. Η κυρία Τερέσια Χιμένε Μπεσερή, λεχτέ το λόγο παρακαλώ να είστε σύντομοι αφού αποφασίσετε και εσείς να πάρετε τον λόγο χωρίς να σε έχει δοθεί ο λόγος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή λέγει ότι δεν μπορεί να ζητήσει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά Δεν άκουσα όμως ε, να πει οποιοδήποτε επιχείρημα σε σχέση με την συγκεκριμένη αυτή αναφορά. Όσο για την ε, εκπρόσωπο της τοπικής κυβέρνησης είπε ότι το σύστημα των προμηθειών είναι ένα μικρό θαύμα στην Ισπανία. Ε, είναι κάτι το οποίο ισχύει μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν λειτουργεί με τον υπόλοιπο κόσμο με τον ίδιο τρόπο το σύστημα. Εγώ ως Ανδαλουσιανή, ως Ευρωπαία, ως Ισπανίδα, εγώ θα ήθελα να γνωρίζω περισσότερο για ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο η προμήθεια των φαρμάκων που επηρεάζει την υγεία των Ανδαλουσιανών. Θέλω περισσότερη διαφάνεια, θέλω περισσότερες πληροφορίες και απλούστερες απαντήσεις γιατί οι Ανδαλουσιανοί είναι οι μόνοι που δεν έχουν την ίδια ευκαιρία με τους υπόλοιπους Ισπανούς όταν λαμβάνουν φάρμακα τα οποία τους δίδει η, ε, η κοινωνική ασφάλιση. Γιατί έχουν ένα τόσο μικρό ποσοστό, 533, ενώ ε, είναι διαθέσιμα σχεδόν 10.000 σε υπόλοιπες ε, περιοχές της Ισπανίας γιατί συμβαίνει αυτό και με ποιο τρόπο επηρεάζεται η καθημερινότητα και η ζωή των ασθενών ε, και υπάρχει τρομερή ανισότητα με τους υπόλοιπους ασθενείς της Ευρώπης. Ζούνε σε ένα γκέτο φαρμακευτικό, υφίστανται συστηματικά διακρίσεις. Και θα ήθελα λοιπόν να πω ότι οι αναφερομένοι ε, ζήτησε να ακουστεί και έχω την αίσθηση ότι η απάντηση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν σαφής. Επαναλαμβάνω, είναι εκατομμύρια Ανδαλουσιανοί και από αυτούς ένας ήρθε εδώ να μιλήσει. Είναι ευάλωτη η κατάστασή τους, θίγονται τα δικαιώματά τους ιδιαίτερα τη στιγμή που επιλέγονται τα φάρμακα τα οποία θα θεραπεύσουν τους πολίτες αυτούς. Θέλουμε απαντήσεις πιστικές γιατί οι Ανδαλουσιανοί έχουν λιγότερα φάρμακα, γιατί οι Ανδαλουσιανοί έχουν χειρότερα φάρμακα από τις υπόλοιπες περιοχές της Ισπανίας. Πρέπει να δοθεί μια λύση και να εξηγιανθεί επιτέλους η κατάσταση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Βυζίνη. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Δεν τα κατέχομαι από τόσο πάθος, αλλά είναι φυσιολογικό αυτό το πάθος όταν μιλάμε για την δημόσια υγεία. Δεν θα επανελθώ στην ικανότητα των κρατών μελών να οργανώνουν το σύστημα δημόσια υγεία του. Απλά θέλω να ευχαριστήσω το ΕΛΚ. Επέμεινε ώστε να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη αυτή η αναφορά. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να δω τους εκπροσώπους ε, που, του φαρμακευτικού τομέα που ισχυρίζονται ότι μιλούν εξ ονόματος των ασθενών. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κάτω από αυτή την αναφορά είναι να βάλουμε στην άκρη οποιαδήποτε πολιτική δαπανών για τη δημόσια υγεία και τα γενώσιμα και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ΕΛΚ για αυτή την άνευ προηγουμένου στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ και να επιστήσω την προσοχή σας στον κατάλογο, γιατί έχω ακόμα κάποιους, σε 12 λεπτά, σε 18 συγγνώμη, λεπτά, θα χρειαστεί να κλείσουμε τις συνεδρίες, οπότε εσείς είστε όσο πιο, το δυνατόν πιο σύντομοι και κάντε κάποια πρόταση για το τι να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, Φαίνεται ότι μερικοί δεν θέλουν εδώ να εκπροσωπείτε τους ασθενείς. Ε, εσείς εδώ εκπροσωπείτε ε, ε, τους, τους ασθενείς που σας έδωσαν τις υπογραφές τους. 500.000 διαβητικοί, ένα σωρό άλλοι ασθενείς. Αλλά φαίνεται μερικοί δεν θέλουν. Εσείς εκπροσωπείτε 8 εκατομμύρια Ανδαλουσιανών ε, ασθενών και 14 εκατομμύρια ε, φτάνει ο αριθμός αυτός εάν μιλήσουν βάλουμε μέσα και τους τουρίστες. Κοιτάξτε, ε, ε, βλέπετε ότι εδώ φέρατε όλους τους, ε, όλους τους βουλευτές και όλα τα, τους εκπροσώπους των κομμάτων. Εσείς θα κερδίσετε από τις ψήφους και όχι από την ουσία. Το, θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ φτάσαμε να συζητούμε το θέμα αυτό από τη στιγμή και μονάχα επειδή οι σοσιαλιστές έλειπαν, ήταν απόντες από δύο συνεχείς συνεδριάσεις και αυτό αυτό το ΕΛΚ κατάφερε να περάσει αυτήν την ε, αναφορά γιατί όλοι προσπάθησαν να μην είναι εδώ οι αναφέροντες. Οι ε, σοσιαλιστές ε, βουλευτές προσπάθησαν να φημώσουν τους αναφερόμενους. Και τώρα θα μπούμε στην ουσία της συζήτηση. Πρώτα απ' όλα. Toda España uno puede comprar, Cecilia va a venir un día España. Α πούμε ότι η Σεσίλια, η πρόεδρό μα, έρχεται μια μέρα στην Ισπανία και μπαίνει σε ένα φαρμακείο και ζητάει ε, και ε, ένα φάρμακο. Μπορεί να διαλέξει οπουδήποτε στην Ισπανία ανάμεσα από 10.000 φάρμακα, ενώ στην η Ανδαλουσία μπορεί να διαλέξει μεταξύ 533 φαρμάκων. Δεν σταματάω, θα μιλήσω όση ώρα μίλησε η κυρία Καπεθόν Ρούη. λέει ο μιλήτρια. Ε, αυτό, κατά την άποψή μου, έρχεται σε κατάφορη παραβίαση τη αρχή τη ισότητα. 533 φάρμακα, ε, αυτά είναι μόνο στα οποία έχουν πρόσβαση ε, οι πολίτες της ε, Ανδαλουσίας. Όμως υπάρχει μια αρχή ισότητας ανάμεσα στους πολίτες της Ισπανίας και της Ανδαλουσίας και επομένως μια τέτοια πρακτική συστέλει τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορία και των ε, αγαθών και των προϊόντων. Ε, ε, ένας μεγάλος άνθρωπος πηγαίνει στο φαρμακείο δεν μπόρεσε και, πρέπει να αλλάξει φάρμακο γιατί δεν, το χάπι το οποίο παίρνει δεν έχει προμηθευτεί γιατί υπάρχει έλλειψη του φαρμάκου αυτού. Ξέρω ότι είναι ειδικά για τους μεγάλους ανθρώπους πολύ δύσκολο το να αλλάζουν φάρμακα αλλά το, πρόβλημα της προμήθειας είναι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολύ συχνά ε, προβλήματα προμήθειας ε, των φαρμάκων στην Ανδαλουσία. Και αυτό που ζητούν οι αναφερόμενοι είναι πολύ σωστό. Είναι να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και μετά θα δούμε αν έχουν δίκιο ή όχι. Πάντως ε, συζητιέται στην ΕΜΒΗ και στην ΙΝΚΟ και ζητούμε από αυτές τις επιτροπές και από, την, τη διοίκηση της, την κυβέρνηση της Ανδαλουσίας μια σειρά από διευκρινήσεις όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Αλλά εάν κλείσετε την αναφορά αυτή, σημαίνει ότι κλείνετε τα αυτιά σα και στα αιτήματα των πολιτών. Δεν σα ενδιαφέρει τι λένε οι πολίτε. Αυτό που σα ζητούμε είναι να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά, ε, να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίε και μετά αποφασίζουμε αν θα την κλείσουμε. Αν την κλείσουμε σήμερα, σημαίνει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη τα δικαιώματα των πολιτών τη Ισπανία. You Λοιπόν, καταλάβαμε τι θέλετε. Κοιτάξτε συνάδελφοι, προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι. Παρακαλώ πείτε μου τι θέλετε να κάνουμε με τη συγκεκριμένη αναφορά. Άγχελα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Σεσίλια. Εμείς ξεκινάμε λέγοντας ότι είμαστε υπέρ του συστήματος. Αυτού θα θέλαμε να γενικευθεί και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό για να αποκτήσουμε καλύτερες τιμές αγοράς ε, των φαρμάκων και μια καλύτερη βάση διαπραγμάτευσης με τη φαρμακευτική βιομηχανία. Νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει το σύστημα αυτό ε, στο, στις διάφορες χώρες. Έχουν υπάρξει και από από τα ανώτατα συνταγματικά όργανα της Ισπανίας το θέμα είναι νόμιμο, δεν δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Ακούσαμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε η αναφορά θα πρέπει να κλείσει. Τώρα γιατί να χάνουμε το χρόνο μας. Είναι απόλυτα νόμιμη η διαδικασία. Νομίζω ότι η ρόλος ακριβώς των οργάνων των πολιτικών είναι να οδηγούν κατά κάποιο τρόπο τους πολίτες και να τους βοηθούν να κάνουν σωστές επιλογές και σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες, τις συντάξεις που υπάρχουν στην Ισπανία. Εγώ προέρχομαι από τις Αστούριας και βλέπω ε, πολλές φορές τους συνταξιούχους να μην είναι σε θέση να πληρώσουν, να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων. Ακόμα και οι απλές βιταμίνες που κάνουν 2 ευρώ για μια σύνταξη η οποία κοστίζει, ε, η οποία ανέρχεται σε 600 ευρώ συνολικά, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Συνεπώς λοιπόν εμείς εδώ είμαστε για να εκπροσωπήσουμε και για να δουλέψουμε για τους πολίτες και όχι για την φαρμακοβιομηχανία. Καλώς σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες. Η κυρία Χέραντς Γκαρθία. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Λέγει η κυρία Γκαμπεσόν ότι η συζήτηση είναι πολιτική και είναι θέμα συμφερόντων. Πράγματι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα σε σχέση με τη σοσιαλιστική τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ε, αυτοί που μας ενδιαφέρουν όμως είναι ο λαός. Εμείς είμαστε εδώ γιατί ανησυχούμε για το λαό, για τους ασθενείς, είτε είναι Ανδαλουσιανοί είτε όχι. Στην Ανδαλουσία υπάρχει πρόβλημα. Οφείλουμε να το καταγγείλουμε το πρόβλημα αυτό. Α, αν υπάρχουν 10.000 φάρμακα είναι γιατί πουλούνται, είναι απαραίτητα. Γιατί ξαφνικά οι Ανδαλουσιανοί να παίρνουν μόνο το 5% γιατί το αποφασίσει ένα συμβούλιο περιφοριακό ή ένας πρόεδρος δεν θα ήταν λογικό να κάνουμε ό,τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ισπανία, στην Γαλλία κτλ. Συνεπώς λοιπόν μιλάμε για περικοπές στη δημόσια υγεία. Απλά είναι θέμα περικοπών στην δημόσια υγεία. Δεν τους ενδιαφέρουν οι πολίτες, τους ενδιαφέρουν να κυβερνήσουν σύμφωνα με τον τρόπο τους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει από ποια χώρα προέρχονται οι ευρωβουλευτές. Εδώ είμαστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν εκπροσωπούμε στενά τη χώρα μας. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό έχει, ε, ε, έχει μειωθεί τα τελευταία έξι χρόνια ε, η φαρμακευτική και η ιατρική δαπάνη στην Ισπανία και νομίζω ότι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε θα πρέπει να, σε αυτό το στίχημα θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μέσα μας επιτρέπουν και εργαλεία μας επιτρέπουν να μειωθεί η δαπάνη. Αυτό έγινε μέσα από τις διαδικασίες διαγωνισμού του φαρμακευτικού ε, προϊόντος. Ε, στην δική μου, ε, στη δική μου περιφέρεια από το 2015 έχει γίνει μια προσπάθεια μείωσης της δαπάνης. Επανειλημμένα ήρθαμε σε επαφή με τους συνταξιούχους και με τους υπόλοιπους που μας έλεγαν ότι εάν πρέπει να να διαλέξω ή να πληρώσω ένα φάρμακο ή να δώσω φαγητό στα παιδιά μου, προφανώς θα διαλέξω το δεύτερο. Εάν ε, μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα φαρμακευτικά προϊόντα με μικρότερη δαπάνη, ε, Βεβαίω θα το κάνουμε και από τη στιγμή που η Κομισιόν λέει ότι η Ανδαλουσιανή κυβέρνηση είναι υπεύθυνη, ε, μια και οι στόχοι του προγράμματος είναι ε, ακριβώς να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα φαρμακευτικά προϊόντα και η διαδικασία διαγωνισμού απέδειξε την αποτελεσματικότητά της, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον ζήτημα προς συζήτηση και επομένως θα πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αγιούσο. Ναι, Σολευδά, ξέρω ότι ζήτησε και το λόγο, αλλά μίλησε ε, τόση ώρα. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατο το θέμα το οποίο έθιξε. Και εσύ ζητά το λόγο. Ωραία. Ναι, δεν σε είδα μετά την κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί υπόθηκαν όλα αυτά τα οποία έπρεπε ε, να υποθούν έτσι ώστε να κατανοήσουν όλοι το πρόβλημα. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για δραστικές ουσίες, ούτε για φαρμακοποιούς, ούτε για φαρμακεία, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάμε για πρόβλημα ε, καταναλωτών που δεν έχουν πρόσβαση. Ε, είναι γεγονός ότι στην Ισπανία είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή φαρμακευτική υγειονομική πολιτική στην Ευρώπη και είναι γεγονός γεγονός επίσης ότι η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας έχει ε, μεταφέρει αρμοδιότητες στις αυτόνομες ε, περιφέρειες. Εδώ όμως μιλάμε ε, για διαφορετική δυνατότητα πρόσβασης στα φάρμακα η εκπρόσωπος της Ανταλλουσιανής κυβέρνησης ε, ε, είπε ότι ε, συζητήθηκαν τα πάντα και γι' αυτό λοιπόν εγώ ζητώ να είπε ότι είναι διαθέσιμη να δώσει όλες τις πληροφορίες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά έτσι ώστε να δούμε, να μάθουμε αν έχει δίκιο ή αν έχει άδικο. Γιατί αν κλείσουμε τώρα την αναφορά δεν θα μάθουμε τα στοιχεία όλα αυτά, δεν θα ξέρουμε αν έχει δίκιο ή άδικο η εκπρόσωπος όπως τη Ανταλουσία τελευταίος ο ομιλητή ο κ. Ουτεργάης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα όπως σας αρέσει να κάνουμε προτάσεις, θα κάνω μία συγκεκριμένη πρόταση. σέβομαι την εκπρόσωπο της Ανδαλουσιανής κυβέρνησης, σέβομαι και όσους πήραν το λόγο και τους συμβούλους τους και θα ήθελα να κάνω μια πρόταση γιατί εσείς οι ίδια πήρατε μια επιστολή της Συμβούλου για θέματα υγείας της ε, Περιφερειακής Κυβέρνησης με ημερομηνία σημερινή και στο τέλος της επιστολής αυτής το οποίο ε, υπογράφεται από την κυρία Αλβάρο Υπάρχει μια παράγραφος η οποία είναι πολύ σημαντική. Λέγεται και το λέγω στα αγγλικά γιατί απεστάλλει στην αγγλική γλώσσα. Αυτός είναι ο λόγος κυρία Βίξτρομ ο υπεύθυνο για θέματα υγείας υπουργό είναι σε διάθεση να, δια, να διευκρινίσει τις ε, ανησυχίες που μπορεί να δημιουργεί το συγκεκριμένο σύστημα. Κοιτάξτε, εμείς θα επισκεφθούμε στην Ανδαλουσία σε λίγες εβδομάδες, για άλλο θέμα βέβαια. Και νομίζω ότι έχουν υπάρξει ευκαιρίες να πάμε κάπου σε μια χώρα για ένα συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξει μια ρύθμιση έτσι ώστε να προσθεθούν κάποια επιπλέον θέματα. Αν η αρμόδια σύμβουλος είναι σε θέση να έρθει ε, να μας συναντήσει, τόσο το καλύτερο. Θα συναντηθούμε με την Περιφερειακή Κυβέρνηση, θα συναντηθούμε με την Περιφερειακή Υπουργό και θα καταφέρουμε ίσως να διευκρινίσουμε ε, τα θέματα της αμφιβολίας μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε την δυνατότητα να συναντηθούμε με την υπεύθυνη για θέματα υγείας, την Σύμβουλο της Περιφερειακής Κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Χιμένες, την αναφερομένη δύο λεπτά μέγιστος χρόνος. Ήθελα να πω κάτι, εξ και το Αντώνιο Ρωμαίο. Perdón.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 λέω ότι δεν είναι νόμιμη η διαδικασία. Εγώ λέω ότι, η, ε, ε, ότι ε, στο φαρμακείο μου έρχονται ασθενείς οι οποίοι παραπονιούνται. Εγώ δεν είμαι το μακρύ χέρι κανενός. Εγώ λέω απλώς ότι έρχονται και μου παραπονιούνται οι ίδιοι οι ασθενείς. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και θα θέλαμε να εστιάσουμε λίγο τη συζήτηση γιατί ε, κάπως ε, πήγε, ε, ε, ξέφυγε η συζήτηση. Κοιτάξτε, λένε μερικοί ότι δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Υπάρχει όμως, γιατί οποιοδήποτε πολίτης του κόσμου από οπουδήποτε πάει στις στα φαρμακεία της Ανταλουσίας θα έχει πρόσβαση μονάχα στα 533 φάρμακα. Ενώ αν πάνε στη Γαλλική, αν πάνε στη Μαδρίτη θα έχει πρόσβαση σε 10.000 φάρμακα. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι δυνατόν ε, ένας πολίτης, ένας ε, ασθενής να μην έχει πρόσβαση στα φάρμακα τα οποία χρειάζεται και τα οποία επιλέγει. Ε, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερο δικαίωμα ή πιο διευρυμένο δικαίωμα, ναι, αλλά όχι συσταλμένο ε, δικαίωμα ο ασθενής εδώ στην Ανδαλουσία δεν μπορεί να διαλέξει ανάμεσα από τα 10.000 σκευάσματα. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση ήταν πολύμορφη, ε, αλλά πιστεύω ότι πρέπει πλέον να έχετε περισσότερα στοιχεία, να γνωρίσετε τις, ε, τα, τα, συνθήκες ε, συζήτησης, γιατί στην Εστρεμαδούρα, γιατί στην ε, Λαμάντσα, γιατί στην Αστούρια δεν έγινε δεκτό, καταψηφίστηκε το πρόγραμμα αυτό να, να δούμε όλα τα, τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να προσπαθήσω να βρω μια πρόταση που θα βρει όλου σύμφωνου. Κάτι αδύνατο πιστεύω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην Επιτροπή που θα ήθελαν να κλείσει αναφορά και άλλοι που θα ήθελαν να διατηρηθεί ανοιχτή και να αναλυφθεί περαιτέρω δράση. Προτείνω λοιπόν να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε και για την προηγούμενη αναφορά. Βγάλτε τις κάρτες ψηφοφορίας σας, βάλτε τις στα μηχανήματα και θα συζητήσουμε, θα ψηφίσουμε μάλλον για το κατά πώς θα κρατήσουμε ανοιχτή ή θα κλείσουμε την αναφορά. Ούτως και θα πράξουμε. Το άνοιγμα είναι το πράσινο, θα το εξηγήσω σε ένα λεπτό αφού βάλουν όλοι τις κάρτες τους. Everybody have your voting card? Yes. Mr. Marias. Βάλατε όλοι τις κάρτες κύριε Μαριά. Can I have uh, half a minute? Θα μπορούσατε να μου δώσετε μισό λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ως, ως μέλος της Επιτροπής θέλω να επισημάνω ότι μπαίνουμε σε μία πολύ επικίνδυνη ατραπό. Αυτή εδώ η Επιτροπή ως στόχο έχει να εξετάζει τα θέματα. Και στις περισσότερες υποθέσεις που έχουμε εξετάσει, τις έχουμε αφήσει ανοιχτές και προσπαθούμε να δώσουμε λύση υπέρ του πολίτη. Βλέπω και στην προηγούμενη περίπτωση και σε αυτή να ερχόμαστε I'm going to speak because I'm a permanent member of the committee, so I will speak. There is no translation in it. There is no ah, translation. Υπάρχει ένα πρόβλημα μετάφρασης ε, στα ισπανικά ενδεχομένως. Στα ισπανικά υπάρχει ένα πρόβλημα μετάφρασης. Σε μια δύσκολη και άσχημη διαδικασία. Και στην προηγούμενη αναφορά και σε αυτή θα κάνουμε μια ψηφοφορία. Με ψηφοφορία κανείς λύνει πράγματι δημοκρατικά τα ζητήματα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο τρόπος λειτουργίας αυτής της Επιτροπής. Προσπαθούσαμε πάντοτε να βρούμε ένα συμβιβασμό με στόχο να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε τους αναφέροντες. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε στην πράξη είναι το κάθε γκρουπ να φέρνει συναδέλφους που δεν έχουν καν σχέση με την Επιτροπή και να μετράμε το συσχετισμό δύναμης. Βεβαίως θα κάνουμε ψηφοφορία, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που κάνουμε πλέον στην Επιτροπή. Θα το κάνουμε και σήμερα σε αυτή την υπόθεση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό ως διαδικασία. Αυτό θέλω να θίξω και να επισημάνω την επικινδυνότητα της διαδικασίας αυτής, γιατί ο καθένας θα φέρνει ένα συσχετισμό δύναμης ναι. και θα κάνουμε ψηφοφορίες τέτοιου τύπου. Το λέω και ναι. στους συναδέλφους του ΕΛΚ και στους συναδέλφους της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Αυτό να το θυμόσαστε ότι είναι λάθος και θα πρέπει να σταματήσει. Έχεις δίκιο. Ήθελες 30 λεπτά και τώρα δύο παραπάνω. You, actually you asked for half a minute, you two minutes. Ουσιαστικά ζήτησες μισό λεπτό, αλλά μίλησες για δυόμιση. Εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτό που παρατηρούμε εδώ στην Επιτροπή είναι ότι πλησιάζουν οι εκλογές η πόλωση συνεπώς μεταξύ των ομάδων εντείνεται κάθε μέρα. Όχι μόνο σε αυτή την επιτροπή και σε άλλες επιτροπές. Και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι όλοι ε, υπερασπίζονται πολύ στεναρά τη θέση τους. Άλλοι θέλουν να την ανοίξουμε, άλλοι θέλουν να την κλείσουμε. Οπότε εγώ λέω να ψηφίσουμε. Συνήθω δεν πρέπει να κάνουμε έτσι. Σήμερα πρέπει να κάνουμε έτσι. Σας γνωρίζω όμως, ξέρω ότι δεν ε, ε, μπορούμε να αποφύγουμε την ψηφοφορία. Οπότε εγώ προτείνω να την κάνουμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν. Το κλείσιμο της αναφοράς είναι το ναι, το πράσινο κουμπί δηλαδή, για να την κλείσουμε. Για να την κλείσουμε πατάτε το πράσινο, για να την κρατήσουμε ανοιχτή πατάτε το κόκκινο. Σωστά. Άρχεται η ψηφοφορία. S&D have one too. Σοσιαλιστές έχουν μία παραπάνω. we have We have now 25 votes and I think that... Τώρα έχουμε 25 ψήφους, νομίζω ότι είναι σωστός ο αριθμός. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Okay, so we have... Λοιπόν, ψηφίσαμε υπέρ του κλεισίματος αυτής της αναφοράς.